Γεια Liebe Kolleginnen und Kollegen. Αγαπητοί συνάδελφοι, ας ε, ξεκινήσουμε. Ich darf Sie herzlich begrüßen zu unserer heutigen Sitzung. Ας ε, καλωσορίζω στην ε, σημερινή μας συνεδρίαση. Η κυρία Νοαγέ θα έρθει σε λίγο, αλλά έχουμε κάποια διοικητικά θέματα πρώτα απ' όλα που οπωσδήποτε σε ενδιαφέρουν, οπότε ξεκινάω από αυτά. Για τη σημερινή ημερήσια διάταξη υπάρχουν παρατηρήσεις, θέλει κάποιο να αλλάξει κάτι, όχι, οπότε εγκρίνεται. Δεύτερον, ανακοινώσει του Προέδρου, να σας πω τα εξής. Πρώτα απ' όλα, όπως ξέρετε, τα βιογραφικά των συμμετεχόντων είναι διαθέσιμα, οπότε δεν χρειάζεται να τους παρουσιάσω η, τα ταξίδια της αντιπροσωπείας στην Κίνα και της ΕΠΑ έχουν εντωμεταξύ εγκριθεί ημερομηνίε. Σας έχουν ήδη γνωστοποιηθεί, αλλά μπορώ να σας τα ξαναπώ. Στην εβδομάδα 7 Ιουνίου πάμε στις ΕΠΑ και νομίζω πιο πριν το Μάιο μετά την Πεντηκοστή από τις 25 δηλαδή του μηνός, πηγαίνουμε Σανκάι και Πεκίνο και ταυτόχρονα είναι και η αντιπροσωπεία της Κίνας στην Κίνα, μόνο στη Σανγκάη όμως, και ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου, ο κύριος Μπούζεκ. Και ήρθαμε σε επαφή με τον κύριο πρόεδρο και θα είναι ίσως παρόν σε μια εκδήλωσή μας Σανγκάη. Έχουμε σχεδόν ε, καταρτήσει το πάνελ των ειδικών. Έχουν γίνει οι προτάσεις από τις διάφορες ομάδες και θα έχουμε ένα πάνελ έξι ατόμων. Την ε, τελευταία φορά θυμάστε είχαμε συζητήσει δύο έγγραφα. Το ένα ήταν του συναδέλφου του κυρίου Χουντή και είχαμε και αφιερώσει πάρα πολύ χρόνο στο έγγραφο του κυρίου Λαμασούρα αλλά όχι τόσο στο έγγραφο του κυρίου Χουντή και θα μπορούσαμε νομίζω να συνεχίσουμε αυτή τη συζήτηση γιατί πρέπει να γίνει γιατί αφορά τις κοινωνικές ε, πτυχές γιατί δεν πρέπει να δώσουμε την εντύπωση πως αυτή η συζήτηση περικόπηκε. Στον επόμενο κύκλο συζητήσεων, αν μιλάμε για θεμαντικά έγγραφα, θα έχουμε μόνο ένα τη φορά στην ημερήσια διάταξη, αλλά θα έχουμε ένα δύο ώρο, δυόμιση ώρες μάλλον. Και δεν ε, χρειάζεται βεβαίως από τις δυόμιση ώρες ε, Νομίζω, μάλλον στην επόμενη συζήτηση μπορούμε από τι 2,5 ώρε να αφιερώσουμε 45 λεπτά για να ολοκληρώσουμε την ε, συζήτηση για το έγγραφο του κυρίου Χούντι και μετά την υπόλοιπη ώρα για το υπόλοιπο. Όσον αφορά τη σημερινή συζήτηση, για να προετοιμαστείτε υπάρχουν και δύο ενημερωτικά έγγραφα από το Τμήμα πολιτική ε, που αξίζει τον κόπο να τα διαβάσετε. Καταθέσαμε επίσης και αντίγραφα των παρουσιάσεων τις οποίες θα δείτε και υπάρχει και το ενημερωτικό δελτίο παριθμών 2 με μία συνέντευξη με την κυρία Περβάνος Μπερές, την εισηγήτριά μας, που και αυτό είναι στη διάθεσή σας. Περνάμε σημείο 3 της ημερήσιας διάταξης, έγκριση των πρακτικών της 14 Ιανουαρίου. Εγώ και το Προεδρείο εδώ πέρα δεν έχουμε λάβει κάποιο αίτημα για αλλαγή στα πρακτικά, οπότε θεωρούμε ότι εγκρίθηκαν και τα πρακτικά. Περνάμε τώρα στο μοναδικό θέμα της σημερινής συνεδρίασης, χρηματοπιστωτική ρύθμιση και εποπτεία. Ένα θέμα το οποίο νομίζω ταιριάζει πάρα πολύ καλά, είναι πάρα πολύ επίκαιρο αυτή τη στιγμή. Όπως ξέρετε πάρα πολλά από τα δικά μας μέλη είναι και μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και συζητιέται και εκεί πέρα το θέμα αυτό. Υπήρχε η έκθεση Ντελαροζιέρ και, και με βάση αυτή την έκθεση η Κομισιόν έκανε μία δική της πρόταση. Το ΔΕ Συμβούλιο επί Προεδρίας αλλά και τώρα με την Ισπανική Προεδρία ασχολείται αυτό το θέμα και επαφίεται σε εμάς να διαμορφώσουμε τη θέση του Κοινοβουλίου. Στην Επιτροπή Οικονομικών Θεμάτων έχει ήδη γίνει αυτό, οπότε και για την Επιτροπή Κινδύνου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας υπάρχει μια εισηγήτρια, η κυρία Σελβιγκουλά από τους φιλελευθέρους και για τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές υπάρχουν εισηγητέ και η συζήτηση ξεκαθάρισε ένα πράγμα, πως είμαστε ακόμα στην αρχή της συζήτησης, οπωσδήποτε όχι στο τέλος και βεβαίως ε, πρέπει να αλλάξουν κάποια πράγματα στον τεμερή διάλογο. Αλλά ένα πράγμα είναι σαφές. Φαίνεται πως υπάρχει μια διακομματική ε, συμφωνία, άποψη, πως ε, οι αγορές οι οποίες πλέον δρούν σε παγκόσμιο επίπεδο πρέπει να έχουν μια εποπτεία και παρακολούθηση η οποία θα είναι και αυτή υπερεθνική. Οπότε ε, έτσι χαιρετήσαμε όχι μόνο την πρόταση Κομισιόν, αλλά κάναμε και ένα βήμα πάρα πέρα από αυτά τα οποία προτείνει η Κομισιόν και θα δούμε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Αυτό βεβαίως συγκεκριμένα σημαίνει θεμελιώδεις αλλαγές. Εάν οι αρμοδιότητες ε, πάνε από το εθνικό στο ευρωπαϊκό επίπεδο, και οι εξουσίε. Έχει αυτό κάποιε επιπτώσει. Οπότε είναι κατανοητό, χωρί να είναι επιθυμητό, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι κατανοητό ότι τα εθνικά κράτη-μέλη αντιδρούν με διαφορετικού τόνους βεβαίω το καθένα, αλλά θα δούμε τι θα γίνει. Τώρα σε κάποια από τα σημερινά έγγραφα ενημέρωσης αναφέρεται στα συμπεράσματα, θα στο διαβάσω γιατί το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Πράγματι, οι ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές δεν έχουν την εξουσία να κάνουν διαχείριση κρίσεων και να χρησιμοποιήσουν δημόσια κονδύλια για να διορθώσουν συστημικά προβλήματα όπως παραδείγματο χάρη χρεοκοπίες τραπεζών. Οπότε αμφισβητείται η αποτελεσματικότητά τους. Είναι πραγματικά ρεαλιστικό να δημιουργήσουμε ευρωπαϊκούς θεσμούς με Αρμοδιότητε εξάντη για μικρο και μάκρο εποπτεία χωρίς να έχουν την δυνατότητα να διασώσουν, ε, να εθνικοποιήσουν ή με άλλο τρόπο να βοηθήσουν χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Συνεπώ ο σύνδεσμο ανάμεσα στη διαχείριση και την πρόληψη τη κρίση πρέπει να είναι υψηλά στην ατζέντα τη ημερήσια διάταξη, χωρί καλύτερη ισορροπία ανάμεσα σε αυτά τα δύο. Όσο φιλόδοξη και αν είναι οι προτάσει ε, θεσμική μεταρρύθμιση, δεν θα είναι αποτελεσματικέ. Πράγματι, αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό ε, ζήτημα με το οποίο πρέπει να ασχοληθούμε και ελπίζω πως ε, η σημερινή συζήτηση θα μας βοηθήσει σε αυτό. Τώρα, είμαι κάπως ε, αμήχανος βεβαίως γιατί είπα το συμπέρασμα και δεν ε, έχει έρθει ακόμα η ομιλήτρια. Οπότε πρέπει να το σχεδιάσουμε λίγο. Γιατί νομίζω μου είπανε πριν από μισή ώρα όταν στην πόρτα ήδη, αλλά δεν ξέρω ποια πόρτα τελικά ήταν. Γι' αυτό νομίζω θα ξεκινήσουμε με τις αγωγικές ε, παρατηρήσεις ε, του πάνελ 2. Είναι ο επικεφαλής ε, της Εποπτικής Αρχής Μπάφιν στην Γερμανία, ο κ. Γιώχαν Σάνιο, τον οποίον καλώς ορίζω και χαίρομαι για το ότι ανταποκρίθηκε στην πρόσκλησή μας. Πρέπει να πω όμως κάτι. Δεν ξέρω όμως πότε θα έρθει η Κριστιανό Αγέ που ήταν και στην ε, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ο κύριος Κριστιανό Αγέ, με συγχωρείτε, που ήταν βεβαίως και διοικητής της ε, Τράπεζας Γαλλίας. Δεν ξέρω, θα δούμε. Ίσως να μπορέσει και να μιλήσει αν δεν φτάνει ο χρόνο. Θα ήταν λυπηρό βεβαίω. Απλά πρέπει να εκμεταλλευτούμε το χρόνο, μια που ήρθαμε όλοι εδώ πέρα, ξεκινήσουμε. Λοιπόν, κύριε Ζάνιο, έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κλίν. Είμαι ευέλικτο. Μπορείτε να με διακόψετε να πάσα στιγμή, ε, ακόμα και αργότερο. Κυρίες και κύριοι, ο απότομος και βίαιος χαρακτήρας της θηριώδους διέλυση η οποία έπληξε τις χρηματοοικονομικές αγορές και οδήγησε σε όλεθρο του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος, ήταν κάτι το αδιανόητο για αυτούς που χρειάστηκε να το αντιμετωπίσουν. Τέθηκαν σε κίνηση δυνάμεις χωρίς έλεγχο, οι οποίες δημιούργησαν γενικούς κινδύνους και ουσιαστικά διέλυσαν κάθε ψευδέστηση ασφάλειας που οι παράγοντε τη αγοράς και οι ρυθμιστέ είχαν δημιουργήσει τα τελευταία χρόνια. Όσοι είδαν να πέφτει ο ουρανό στο κεφάλι τους και ήμουνα μεταξύ αυτών. Συγγνώμη, μια στιγμή λέει ο πρόεδρο. bonjour. You have to start immediately. Θα ήθελα να χαιρετήσω τον κύριο μιλτή μας, τον κύριο Κριστιανού Αγέ, ο οποίος είναι διοικητής της Τράπεζας της Γαλλίας και με μεγάλο ενδιαφέρον είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε τις εισαγωγικές σας παρατηρήσεις. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, κυρία Εισηγήτρια, κυρίες καθώς και κύριοι, μέλη της ειδικευμένη Επιτροπής για τη Χρηματοοικονομική κρίση. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ καταρχήν που με καλέσατε σήμερα εδώ σε μια πολύ σημαντική στιγμή καθώς ε, προετοιμάζεται την αρχιτεκτονική εποπτεία στην Ευρώπη. Θα ήθελα να προσπαθήσω να απαντήσω σύντομα στα δύο ερωτήματα που θέσατε και που σας απασχολούν και εσάς, δηλαδή σε ποιο βαθμό προσπαθούμε να διορθώσουμε τις ανεπάρκειες της ε, νομοθεσίας και της εποπτείας που φάνηκαν μέσω της κρίσης και έπειτα τη άλλη ερώτηση που ήταν το πιο πρότυπο εποπτείας ε, θα έχουμε για την Ευρώπη. Τώρα φυσικά και υπάρχουν ανεπάρκειες στην νομοθεσία και στην εποπτεία που φάνηκαν από την κρίση, το θέμα είναι να δούμε κατά πόσο όλα τα προγράμματα που ξεκίνησαν από την ομάδα G20 καταρχήν σε διεθνές επίπεδο, επίπεδο όσον αφορά την ε, γενική παγκόσμια μάλλον σταθερότητα αλλά και όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Τραπεζικών Ελεγκτών ε, κατά πόσο αυτά τα προγράμματα θα απαντήσουν στις ανεπάρκειες. Εγώ θα τονίσω τρεις πτυχές των ανεπαρκειών, όπως εγώ τις έχω αντιληφθεί. Αυτό που αφορά τα συμπληρωματικά στοιχεία που είναι πολύ σημαντικά για να μπορέσει να διατηρηθεί η χρηματοπιστωτική σταθερότητα σε περίπτωση κρίσης και κάποιες ε, παρατηρήσεις όσον αφορά το πεδίο της εποπτείας, δηλαδή τους τομείς που θα πρέπει να ρυθμιστούν και να ελέγχονται. Καταρχήν όσον αφορά την πρόνοια. Την προληπτική εποπτεία. Καταρχήν, πρώτος άξονας μεταρρύθμισης που ήταν ο πιο ε, επίγον και ο πιο αναδιαφυσβήτητος, τα μέτρα τα οποία δηλαδή φάνηκε ότι ήταν οπωσδήποτε απαραίτητο να ληφθούν μετά από την κρίση, είναι δύο μορφών. Καταρχήν, οι απαιτήσει όσον αφορά την ε, και τις διάφορε διάφορες συναλλαγές στην αγορά. Είδαμε κατά τη διάρκεια της κρίσης ότι η μεταφορά της κρίσης που επιτρέπει την τιτλοποίηση μεταφράζεται σε μία εξάπλωση των κινδύνων σε όλους τους τομείς της οικονομίας και ε, είναι ένας τομέας όπου οι βασικές απαιτήσει είχαν ε, υποτιμηθεί. Και αυτό σε μεγάλο βαθμό διορθώθηκε με την εφαρμογή του πρώτου σχεδίου ε, σταθερότητας μέσω της οδηγίας ΣΕΡΤΕ 2 και 3 και της οδηγίας για την φερεγγιότητα. Παραμένει ωστόσο ένας τομέας στον οποίο θα εξετάσετε και εσείς εδώ στο Κοινοβούλιο Δηλαδή ότι πρέπει να διαβεβαιώσουμε ότι οι οργανισμοί ε, βαθμολόγησης, αξιολόγησης θα πρέπει ε, και, αυτές να, και αυτοί να επιστοποιηθούν. Ένας άλλος ε, τομέας που μου φαίνεται ότι είναι προτεραιότητας και που πιστεύω ότι θα μελετηθεί μέσα στο πλαίσιο της μελέτης που γίνεται για την μεταρρύθμιση των ισχυών των κανόνων θα πρέπει να διασφαλιστεί καλύτερη κάλυψη των κινδύνων με μια δυναμική πρόβλεψη που θα λαμβάνει υπόψη, θα έλεγα, το σύνολο του οικονομικού κύκλου και του κύκλου πιστώσεων, δηλαδή θα βασίζεται όχι μόνο στην ε, ύπαρξη των επαληθευμένων ε, ζημιών, αλλά και στους κινδύνους που με βάση στατιστικά και μελέτες ε, θα μπορούσαν να παρουσιαστούν. Γενικότερα λοιπόν θα πρέπει να ενισχυθεί ο χειρισμός και η διαχείριση του κινδύνου από όλε τις πλευρές του. Από αυτή την άποψη η Ευρώπη επειδή έχει υιοθετήσει τη Βασιλεία 2 θα βρίσκεται ήδη σε προηγμένη κατάσταση και σε υπόλοιπες περιοχές του κόσμου και κυρίως στις ΗΠΑ θα πρέπει να εφαρμοστεί όσο γίνεται πιο σύντομα το σύστημα Βασιλεία 2, δηλαδή ένα σύστημα που μετρά τους κινδύνους αντιστοιχεί τις ε, απαιτήσεις κεφαλαίων ε, στον βαθμό του κινδύνου και έτσι στηρίζεται στο δεύτερο πυλώνα όπως ε, ονομάζεται, δηλαδή στο είδος κινδύνου που περιέχεται σε κάθε οργανισμό ή φορέα. Δεύτερος άξονας της μεταρρύθμισης είναι τα μέτρα τα οποία δεν χρειαζόταν να υιοθετηθούν τόσο κατεπηγόντως όσο οι απαιτήσει για τις ε, συναλλαγές της αγοράς, για τις, επιχει... για τις ε, συναλλαγές και που θα πρέπει Ωστόσο εδώ να μετρηθεί πολύ συγκεκριμένα ο πιθανός αντίκτυπός του στην πραγματική οικονομία. Είναι δηλαδή δυνητικά μέτρα τα οποία βρίσκονται υπό εξέταση φέτος σε διεθνές επίπεδο και σήμερα και στο πλαίσιο της Επιτροπής της Βασιλείας. Να αναφέρω δύο τομείς που θεωρώ ότι είναι προτεραιότητας. Ο πρώτος αφορά τον ορισμό των ιδίων πόρων και την ποιότητα των ιδίων πόρων. Έχουμε διάφορους ορισμούς, όχι μόνο στο σύνολο του κόσμου, αλλά και ακόμα και εντός Ευρώπης. Θα πρέπει να εναρμονιστεί ο ορισμός για να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη. Και θα πρέπει να εναρμονιστεί ο ορισμός, διότι ο περίπλοκος χαρακτήρας ορισμένων μέσων και ορισμένων μέσων ε, και κινήσεων κεφαλαίων οδήγησαν σε τεράστιες απώλειες και άρα ε, ήταν πολύ πιο δύσκολο να υπολογιστεί η φεργιότητα ορισμένων ιδρυμάτων. Η εγκυρότητα δηλαδή των κεφαλαίων θα πρέπει να καθοριστεί, των ιδίων κεφαλαίων Και αυτό θεωρώ ότι είναι μεγάλη προτεραιότητα. Κάτι ακόμα είναι σημαντικό, είναι η μέτρηση του κινδύνου ρευστότητα. Είναι ένα θέμα επίση περίπλοκο. Μέχρι στιγμή δεν υπήρχαν πρότυπα ρευστότητα σε επίπεδο διεθνέ. Υπήρχαν μάλιστα χώρε ε, συμπεριλαμβανομένων και χωρών εντό τη Ευρώπη που είχαν εγκαταλείψει κάθε ρύθμιση τη τραπεζική ρευστότητα και πιστεύω πως χρειάζεται να παροτρύνουμε τις τράπεζες να μετρήσουν καλύτερα το κίνδυνο της ρευστότητα, η στάθμιση αυτών των μέτρων, δηλαδή συγκεκριμένοι κανόνες, η στάθμιση αυτών είναι πολύ ε, ευαίσθητη υπόθεση και θα πρέπει να προσεχθούν πολλά σημεία. Καταρχήν, να μην κατακαιρματιστεί η ανάλυση γιατί θα ήταν πραγματικά αποφευκταίο το να επανεθνικοποιηθεί η δραστηριότητα η τραπεζική, δηλαδή να περιοριστεί από τα σύνορα όσον αφορά τη ρευστότητα. Θα πρέπει να επιτραπεί η χρήση προηγμένων μεθόδων όταν αυτό είναι δυνατόν, όταν δηλαδή ε, τα ιδρύματα μπορούν να τα εφαρμόσουν, γιατί είναι πιο αποδοτικό κάτι τέτοιο. Και έπειτα γενικότερα δεν θα πρέπει να θάψουμε τις τραπεζικές δραστηριότητες ενώ υποτίθεται ότι προσπαθούμε να τις ε, θεραπεύσουμε. Θα γίνει λοιπόν αυτή η στάθμιση, θα πρέπει να γίνει πολύ προσεκτικά. θα έλεγα λοιπόν ότι υπάρχουν ε, τέλος άλλα μέτρα επί των οποίων εργαζόμαστε σε διεθνές επίπεδο και που μπορεί να είναι ενδιαφέροντα αλλά τα οποία τα βλέπω πιο ε, με μεγαλύτερη προσοχή. Το πρώτο είναι ε, το μέτρο του βαθμού λειτουργίας των τραπεζών ως μοχλού, του βαθμού μόχλευσης των τραπεζών. Να δούμε δηλαδή κατά πόσο ισχύει και ε, να γίνει μια βαθύτερη ανάλυση του φαινομένου της μόχλευσης και αν αυτό ήταν σε αντίθεση με τη μέτρηση των σταθμισμένων κινδύνων όπως αυτός υπάρχει, αυτή υπάρχει στην Βασιλεία 2. Κάτι τέτοιο θα ήταν επικίνδυνο γιατί θα μπορούσε να οθήσει παραδόξως στις τράπεζες να αναλάβουν περισσότερους κινδύνους για να έχουν ενεργητικό πιο κερδοφόρο μέσα στο πλαίσιο ενός συγκεκριμένου χαρτοφυλακίου και έπειτα δεν θα επέτρεπε να μπορούμε να συγκρίνουμε τα ιδρύματα των χωρών μεταξύ τους εάν τα λογιστικά πρότυπα δεν είναι ακριβώς τα ίδια. Θα πρέπει δηλαδή να υπάρχουν μέτρα ανάλυσης και μέσα ανάλυσης ώστε ε, να μπορούν να καταγράφονται και με βάση τον πυλώνα 2. Επίσης θα έπρεπε να έχουμε τα αντικυκλικά Ε, όρια ναι. τα οποία θα, είναι, θα, ε, με βάση τον κύκλο, ένα μέσο το οποίο είναι ωστόσο πολύ δύσκολο να φτιαχτεί και να χρησιμοποιηθεί. Θα πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος ώστε αυτό να προταθεί στον νομοθέτη, αλλά είναι πολύ περίπλοκο ως μέτρο. Να ολοκληρώσω λέγοντας ότι θα πρέπει να μεριμνήσουμε αυτό γίνεται και έχει υποθεί και στην Επιτροπή της Βασιλείας στην μακροοικονομική πλαισίωση των μέτρων που προτείνουμε. Φυσικά θα πρέπει να προσπαθήσουμε να προτείνουμε κανόνες που θα επιτρέψουν να έχουμε ένα χρηματοπιστωτικό σύστημα πολύ πιο στέρεο, πιο κεφαλαιοποιημένο, με καλύτερη ανάλυση των κινδύνων Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να αποφύγουμε το να αρχίσουμε ξανά να διατρέχουμε το κίνδυνο μια τέτοια κρίση όπω αυτή που ζήσαμε. Αυτό ο κίνδυνο θα πρέπει να εξαλειφθεί οπωσδήποτε. Ταυτόχρονα θα ήταν εξίσου άσχημο το να προτείνουμε κανόνες που θα κατέληγαν σε τροχοπέδι της χρηματοδότησης της οικονομίας μας και που θα ε, διέκοπταν οριστικά την ανάπτυξη, την μεγέθυνση όπως αυτή που γνωρίζουμε. Είναι μια εξαιρετικά ευαίσθητη ισορροπία που πρέπει να βρεθεί και θα πρέπει να το κάνουμε ε, προσωμιώνοντας τα μακροοικονομικά μέτρα τα οποία προτείνουμε. Και για να το κάνουμε αυτό, ε, στην Βασιλεία κάνουμε μακροοικονομικές δοκιμές με την ε, στήριξη διεθνών τραπεζών και όλων των χρηματοπιστωτικών ζωνών που εμπλέκονται και νομίζω πως κάτι τέτοιο είναι θεμέλιο για τις περαιτέρω εξελίξεις. θα πρέπει εξίσου εξονυχιστικά να εξετάσουμε ποιο θα είναι ο αντίκτυπο των διαφόρων μέτρων που προτείνονται με βάση την προβλεπόμενη στάθμιση. και τις ε, ιδιαιτερότητες κάθε οικονομίας, κάθε αγοράς και του τρόπου με τον οποίο γίνεται η μετατροπή της διάρκειας και η χρηματοδότηση κάθε τμήματος ε, της οικονομίας μας, για να είμαστε βέβαιοι ότι θα μπορέσουμε να διαχειριστούμε τις επιπτώσεις των αλλαγών αυτών. Δεύτερη πτυχή των ε, προβλημάτων αφορά το τι μπορούμε να κάνουμε σε περίπτωση κρίσης τι δεν είχαμε, τι δεν λειτουργήσε καλά, τι χρειάστηκε να φεύγουμε βιαστικά για να μπορέσουμε να διατηρήσουμε την ε, χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Στα όσα λείπουν, αυτό που είναι πολύ βασικό είναι η προστασία των καταθετών. Είναι ένα θέμα ιδιαίτερα προσφυλές στους ε, ευρωβουλευτές, το γνωρίζω. Υπάρχουν ε, οι εγγυήσεις ε, καταθέσεων στις διάφορες χώρες, αλλά διαφέρουν πολύ τα συστήματα. Ορισμένα βασίζονται σε συμβολές εξάντε, ορισμένες φορές υπολογίζονται όπως στη Γαλλία με βάση το κίνδυνο που παρουσιάζει κάθε συμβαλόμενο ίδρυμα. Τα ποσά των εγγυήσεων είναι εναρμονισμένα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά πιστεύω ότι μια πιο προθυμένη εναρμόνιση στη, σε σχέση με τον όγκο των εγγυημένων ε, αποθεματικών στον τρόπο με παρέμβασης των ταμείων εγγυήσεων και ένας ακόμα, ένα ακόμα στάδιο θα έπρεπε ίσως να ξεπεραστεί με ένα πραγματικό ευρωπαϊκό σύστημα ταμείο εγγυήσεων, δηλαδή ένα είδος ε, αντασφάλισης των εγγυήσεων κάθε χώρας, εκεί νομίζω θα πρέπει να προοδεύσουμε. Επίσης θα πρέπει να συζητήσουμε την ενδεχόμενη εσείς ε, ε, ε, εμπλοκή όλων αυτών των συστημάτων που θεωρούνται εξαιρετικά μεγάλα που και ε, εκ του όγκου τους αδύνατον να καταρρεύσουν. Θα πρέπει να διδαχτούμε από το πάθημα γιατί είναι σχετικά εύκολο και καθόλου προβληματικό το να φτιάξουμε ένα κατάλογο με συστημικό ορισμούς. Κάτι τέτοιο, ωστόσο μου φαίνεται πως είναι αρκετά αμφίβολο. Το να φτιάξουμε έναν κατάλογο τραπεζών ή χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων συστημικό θα μπορούσε να αποδειχθεί αντιπαραγωγικό, διότι αυτό θα αύξανε ή θα θεσμοθετούσε την ηθική τον ηθικό κίνδυνο Δηλαδή, βάζετε κάποιο ίδρυμα ε, να πληρώνει ένα φόρο και στην ουσία του λέμε ε, ότι σας βάζουμε ε, να πλη... τους λέμε θα σας θα αφήσουμε να λειτουργήσετε από τη στιγμή που θα πληρώνετε ένα συγκεκριμένο πριμ έτσι δημιουργούμε ηθικό κίνδυνο από την άλλη πλευρά ωστόσο πιστεύω πως δεν υπάρχει σχέση ανάμεσα στο μέγεθος και το συστημικό κίνδυνο Όταν βλέπουμε το μέγεθος των ιδρυμάτων που κατέρευσαν και που χρειάστηκε να σωθούν με νύχια και με δόντια από τα κράτη, βλέπουμε ότι μεγάλος αριθμός αυτών των οργανισμών δεν θα είχαν μπει στον κατάλογο των συστημικού κινδύνου αν τον είχαμε φτιάξει πριν την κρίση και ότι στην πράξη μετά από τα όσα ζήσαμε είδαμε ότι ήταν απαραίτητο τα κράτη να διοργανώσουν τη διάσωση ίσως και την ε, ρευστότητα ή τη μεταπόληση αυτών των ιδρυμάτων, αυτών των οργανισμών. Τόσο λοιπόν η ιδέα ενός καταλόγου οργανισμών, όσο και η ιδέα του να βάλουμε μια, έναν αναλογικό φόρο στον ε, ε εν κίνδυνο, είναι κάτι το πολύ αμφισβητήσιμο. Προφανώς αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να γνωρίσουμε το πρόβλημα αυτό, το οποίο συνδέεται με το λεγόμενο ηθικό κίνδυνο. Πιστεύω ότι όταν η απαράγραπτη η παρέμβαση του κράτους, των κρατικών φορέων, θα πρέπει να συνοδεύεται με ριζοσπαστικά και ατομικά μεμονωμένα μέτρα, όπως η αλλαγή των διοικητικών συμβουλίων, παραδείγματο χάρη των διευθυνόντων σε μια εταιρεία ή το γεγονό ότι οι ήδη υπάρχοντες μέτοχοι θα πρέπει να αναλάβουν τον κίνδυνο και δεν θα πρέπει να διαχυθεί αυτός ο κίνδυνος ε, σαν αποτέλεσμα της δυσμενούς κατάστασης του πιστοτικού αυτού ιδρύματος. Πιστεύω ότι είναι απόλυτα φυσιολογικό λοιπόν σε αυτές τις περιπτώσεις ένα πιστοτικό ίδρυμα το οποίο έχει αποτελέσει αντικείμενο μιας επιχείρησης διάσωσης μαζικής και μακροχρόνιας θα πρέπει να κατακαιρματιστεί είτε συνολικά είτε εν μέρη, να πολιθεί σε άλλους πιστοτικούς φορείς, να μην παραμείνει δηλαδή ως έχει, με τη μορφή που είχε, μετά από μια μαζική και μεγάλης κλίμακος διάσωση, η οποία έχει διαρκέσει και στο χρόνο. Δεν θεωρώ ότι θα ήταν παράλογο επίσης και μη φυσιολογικό το κράτος όταν διαπιστώνει ότι το κόστος μιας επιχείρησης διάσωσης η διάσωση λοιπόν αυτών των πιστοτικών φορέων όταν σημαίνει και ένα πρόσθετο άχθος για τον φορολογούμενο δεν θα ήταν λοιπόν παράλογο το κράτος να επιβάλλει εκ των υστέρων φορολογία, πρόσθετη φορολογία στο τραπεζικό σύστημα, ώστε να μπορέσει να ανακτήσει ο φορολογούμενος το κόστος το οποίο επομίστη λόγω της άφρονος ή της όχι αρκετά σόφρονος συμπεριφοράς των πιστοτικών ιδρυμάτων. Μια τρίτη πτυχή λοιπόν των ατελειών που πρέπει να αντιμετωπίσουμε είναι το λεγόμενο περιβάλλον του τραπεζικού, τραπεζικού τομέα. Πρόκειται λοιπόν για φορείς που δεν, έχουν, δεν υπόκειται απόλυτα στην τραπεζική ρύθμιση, αλλά επέχουν μεγάλη σημασία. Αναφέρομαι σε θέματα όπως είναι τα λογιστικά πρότυπα φαινός, και γενικά τον χώρο των εργαλείων τα οποία δεν υπόκειται σε ρύθμιση. Για τα λογιστικά πρότυπα. Εδώ θα πρέπει να ληφθεί υπόψη πάντα η απέτηση της χρηματοοικονομικής σταθερότητας. Αυτό σημαίνει συγκεκριμένα ότι εμείς θα πρέπει να δίνουμε μεγαλύτερη σημασία στην καταγραφή επί τη βάση της αξίας αγοράς όταν δεν υπάρχει επαρκής ρευστότητα και στη συνέχεια στην ε, αποτίμηση της πραγματικής αξίας όταν αυτό θα πρέπει, όταν αυτή η αξία θα πρέπει να καταγραφεί σε διαδικασίες ανταλλαγής ή διαπραγμάτευσης στοιχείων ε, ενεργητικού. Και επίσης, όπως ζήτησαν και οι G20, θα πρέπει να προσπαθήσουμε να επιτύχουμε τη σύγκληση όλων των συστημάτων προς ε, διεθνή λογιστικά πρότυπα υψηλής ποιότητα και προφανώς εδώ δίνω μεγαλύτερη σημασία στην ποιότητα των προτύπων. Η σύγκληση βέβαια είναι δευτερεύουσα αλλά και αυτή παραμένει σημαντική. Θα πρέπει όμως να προσπαθήσουμε να εξασφαλίσουμε ότι θα συγκλίνουν εν καιρό τα λογιστικά συστήματα προς συστήματα τα οποία λαμβάνουν πλήρως υπόψη της αναγκαιότητας σταθερότητας στον χρηματοοικονομικό τομέα και επίσης η <clears throat> ευκυβερνησία του συστήματος των λογιστικών προτύπων θα πρέπει να γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε να λαμβάνεται υπόψη η αρχή της πρόληψης και η αναγκαιότητα της σταθερότητας και να υπάρξει λοιπόν μια ομαλοποίηση και μια τυποποίηση σε όλα αυτά τα λογιστικά πρότυπα. Σε ό,τι αφορά τώρα το γενικό περίγυρο της ρύθμισης, θέλω να σας πενθυμίσω από πού προέκυψε η κρίση. Η κρίση ξεκίνησε στις ΗΠΑ με την ε, διανομή πιστώσεων σε μη φερέγγιους ε, πιστολήπτες από οργανισμούς οι οποίοι δεν υπέκυντο επαρκώς σε ρύθμιση. Επομένως, ο περίγυρος της ε, ε, περιοχής αυτής εκτός ρυθμίσεως το αρκετά περιορισμένος. Ο περιγυρος τη ρύθμιση ήταν αρκετά περιορισμενος Εδώ η Ευρώπη μπορεί να είναι πιο υπερήφανη γιατί η δική μας ρυθμιστική δραστηριότητα καλύπτει το σύνολο των δραστηριοτήτων του χρηματοπιστωτικού τομέα. Του τουλεχθέντος βέβαια, όταν θέλουμε να ανταποκριθούμε στις επιθυμίες οι οποίες διατυπώθηκαν από τους G20 και στις βασικές αρχές που διατύπωσαν, όταν είπαν ότι όλε οι αγορέ, όλοι οι παίκτε τη αγορά, όλε οι χρηματοοικονομικές αγορέ θα πρέπει να υπόκεινται σε εποπτεία και ρύθμιση, γνωρίζουμε ότι υπάρχουν ακόμα κάποιοι πρόοδοι, κάποιες πρόοδοι που πρέπει να γίνουν, ιδίω σε ό,τι αφορά τι εταιρείε πιστοληπτική αξιολόγηση, Υπάρχει μια τέτοια κίνηση ήδη σε ευρωπαϊκό επίπεδο. επίση ε, τα, τα μία ή τα κεφάλαια που βασίζονται στη μόχλευση τα, οι συμφωνίες ε, προαίρεσης που βασίζονται σε παράγωγα ε, εργαλεία μέσω ηλεκτρονικών πλατφορμών όπου καταγράφεται μεν όπου πρέπει να καταγράφονται οι συναλλαγές ακόμα και αν γίνονται εκτός χρηματιστήριων. Όλα αυτά έχουν σημασία λοιπόν για να αντιμετωπίσουμε τα συστημικά προβλήματα. Ακόμα και σε ευρωπαϊκό επίπεδο εξακολουθεί να ισχύει κάτι το οποίο ισχύει πολύ περισσότερο στο διεθνές επίπεδο ότι ο ορισμός του τι είναι χρηματοπιστωτικό ίδρυμα μπορεί να ποικίλει από μια χώρα στις άλλες. Αυτά λοιπόν κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι αυτά ήταν τα περισσότερα από αυτά που ήθελα να πω σε σχέση με το παρελθόν και σε σχέση με το ε, μοντέλο ρύθμισης. Θα είμαι πολύ σύντομο γιατί είδα ότι ο χρόνος μας πιέζει στην Ευρώπη. Η αρχιτεκτονική ρύθμιση η οποία έχει προταθεί από την ομάδα εργασίας του κυρίου Λαροζιέρ <clears throat> πιστεύω ότι αποτελεί μια ιδιαίτερα εύστοχη απάντηση στην χρηματοοικονομική κρίση. Πιστεύω ότι θα μπορούσα σχεδόν να σταματήσω εδώ αλλά προηγουμένως θέλω να επιμείνω στο να σας πω ότι ένα από τα ουσιώδη διδάγματα που πρέπει να αντλήσουμε από την κρίση είναι το ότι η εγκύτητα μεταξύ των ρυθμιστών και της Κεντρικής Τράπεζας είναι απαράγραπτη προϋπόθεση για μια ταχεία αντίδραση και μια εύκαμπτη αντίδραση ενώπιον καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης. Και παραλλήλως, η εγκύτηση του ρυθμιστού προς την, την Κεντρική Τράπεζα ή μάλλον προς το Ίδρυμα το οποίο την χάνει Ρύθμιση, εξασφαλίζει την αποτελεσματικότητα τη ρυθμίση, Δηλαδή, μια αρχιτεκτονική κατά την οποία θα έχουμε σε εθνικό επίπεδο ρυθμιστέ, με πολύ καλή δυνατότητα συντονισμού, όπω προτείνεται από την ομάδα Ντελαροζιέρ για, του Ευρωπαϊκού, για τα ευρωπαϊκά πιστοτικά ιδρύματα και όπου μπορούν να υπάρχουν επίσης ομάδες ρυθμιστών που δουλεύουν σε διαμεθοριακό επίπεδο για τη ρύθμιση αυτή, είναι μια πολύ καλή αρχιτεκτονική για τις τωρινές ε, συνθήκες. Τώρα δεν συμμεριζόμαι απόλυτα την άποψη του, της ομάδας Τελαροζιέρ για ένα μοναδικό ρυθμιστή σε ό,τι αφορά τις διαμεθοριακές ε, ε διαμεθοριακά πιστοντικά ιδρύματα, γιατί αυτό θα οδηγήσει σε απόσταση από τα ρυθμιζόμενα ιδρύματα. Υπάρχει κίνδυνος να υπάρξει κατακαιρματισμός εδώ και να υπάρξει μια δυνατότητα κατά κάποιο τρόπο ε, Διαμεσολάβηση μεταξύ διαφορετικών ρυθμιστικών συστημάτων. Επομένως, εγώ δεν πιστεύω, όπως είπα και προηγουμένως, ότι πρέπει να υπάρχει ένας κατάλογος συστημικού χαρακτήρα ιδρυμάτων που να υπόκειται σε διαφορετικούς ρυθμιστικούς κανόνες. Εν κατακλείδη, θα σας έλεγα ότι η ιδέα του λεγόμενου Twin Peaks, να υπάρχει δηλαδή παράλληλη ρύθμιση των τραπεζών και των ασφαλιστικών ιδρυμάτων, αυτό μου φαίνεται ότι είναι μια πολύ καλή ιδέα στο βαθμό που αυτό δεν διαρρυκνεί την απαραίτητη εγκύτητα μεταξύ ρυθμιστικών αρχών και κεντρικής τράπεζας που για μένα θα πρέπει να αποτελέσει την προτεραιότητα. <clears throat> θα ήταν λοιπόν μια ενδιαφέρουσα προσέγγιση το να φέρουμε πιο κοντά τη ρύθμιση των τραπεζών και των ασφαλιστικών εταιριών, ενώ παράλληλα εξασφαλίζουμε την εγκύτητα του ρυθμιστή με την Κεντρική Τράπεζα, αυτό είναι κάτι το οποίο είναι υπομελέτη ή έχει ήδη υλοποιηθεί σε ένα πολύ σημαντικό αριθμό ευρωπαϊκών χωρών και πιστεύω ότι αυτό είναι μια πολύ θετική εξέλιξη. Κύριε Πρόεδρε, Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, Σα ευχαριστώ εγώ. Περνάμε στι ε, ερωτήσει, Επειδή έχει περάσει και η ώρα, θα ήθελα να ακούσουμε πρώτα απ' όλα τους συντονιστές, αλλά ξεκινάμε βέβαια με την εισηγήτρια, με την κυρία Περβάνς Μπερές και μετά θα δώσω τον λόγο στον Οτμαρ Μαρκάρης. Ένα λεπτό ο καθένας και όταν τελειώσει το λεπτό θα σας βγάζω κόκκινη κάρτα. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ κυρία Δίκητα για αυτές τις ε, προοπτικές ε, και την ανάλυση για τις ανεπάρκειες και τις προοπτικές ε, δύο ερωτήσεις. Καταρχήν, Όσον αφορά τα ίδια κεφάλαια των τραπεζών, βλέπουμε πώ θα αντιδράσουν, ότι δεν είναι η ώρα να γίνει κάτι τέτοιο και ούτω καθεξής, αλλά ο τρόπος με τον οποίο το συνδέσατε με την υπόθεση των προϊόντων, δηλαδή της τιτλοποίησης, είναι πολύ σημαντικό για το πώς θα τεθεί το ζήτημα, γιατί θεωρητικά και σφαιρικά θα μιλήσουμε για την αντιογωνιστικότητα της οικονομίας Ευρώπης ε, προς τη ΣΥΠΑ, που δεν θα μας επιτρέψει να προχωρήσουμε πιο μακριά. Αλλά έχω την εντύπωση ότι υπάρχουν πολλές προτάσεις επιτάπη και ότι βασικά πίσω από τι εργασίε τη Βασιλεία έχουμε ήδη ξεκινήσει με την ιδέα ότι πρέπει να αυξηθούν τα ίδια κεφάλαια χωρί να γίνει συζήτηση ε, για τι εναλλακτικέ. Και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε ευρωπαϊκή κλίμακα, τι θα ήταν καλύτερο για το δικό μας τελικό στόχο, που δεν είναι τόσο η υγεία του τραπεζικού τομέα, όσο η χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας. Δεν έχω το χρόνο να θέσω μια δεύτερη ερώτηση, αλλά θα τη θέσω. Τι θέλετε να κάνετε τι πιστεύετε με τις ε, συμφωνίες της Βασιλείας και τις συνθήκες. Θα τις... Μήπως θα πρέπει να γίνουν συνθήκες. Ευχαριστώ. Βεβαίω ε, ήταν σε δύο τμήματα η παρέμβασή σα, αλλά όσον αφορά το πρώτο τμήμα δεν θα μπορέσουμε να λύσουμε όλα τα ζητήματα τη ε, εποπτεία ούτε των ιδίων κεφαλαίων κτλ. Και είμαστε τώρα στην εποπτεία και είπατε πως η έκθεση Λαροζιέρ είναι σωστή, αλλά εμείς θέτουμε το ερώτημα πως πρέπει να υπάρχει ευρωπαϊκή εποπτεία η οποία θα επιβάλλει κυρώσεις όταν η τοπική, η εθνική εποπτεία δεν δραστηριοποιείται επαρκώς ή δεν μπορεί να συμφωνήσει σε μια αγορά η οποία είναι πλέον παγκοσμιοποιημένη. Πώς βλέπετε εσείς μια ευρωπαϊκή, μια παγκόσμια εποπτεία. Και η κοινή θέση του, του Συμβουλίου που είναι πίσω από την έκθεση Λαροζιέρ, πώς βλέπετε εσείς να διαμορφώνει τις ευρωπαϊκές πιθανότητες ε, επιβολής κυρώσεων. Merci, σας ευχαριστώ Πρόεδρε για τα ίδια κεφάλαια, για την ενίσχυση των ιδιών κεφαλαίων των πιστοτικών ιδρυμάτων ή αν θέλουμε να διαλέξουμε μεταξύ κεφαλαίων ιδίων ή κεφαλαίων που θα πρέπει να κινητοποιούνται όταν χρειάζεται να αντιμετωπίσουν τις κρίσεις, εγώ πιστεύω ότι πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση στα ίδια κεφάλαια, γιατί βασικά ο στόχος μας είναι να αποφύγουμε να διαβρωθεί το προφίλ των ε, πιστοτικών αυτών ιδρυμάτων έναντι των ε, δραστηριοτήτων τους θα είναι πιο καλό για το χρηματοπιστωτικό σύστημα αν μπορέσουμε να μειώσουμε στο ελάχιστο τον κίνδυνο μιας κρίσης και της ανάγκης να υπάρξει οποιαδήποτε μορφή παρέμβασης. Φυσικά δεν μπορούμε να εξαλείψουμε τη δυνατότητα κρίση χωρίς να εξαλείψουμε και την χρηματοοικονομική δραστηριότητα. Αλλά αυτό το οποίο με ενδιαφέρει ιδιαίτερα είναι το να διατηρήσουμε την χρηματοδότηση τη πραγματική οικονομία. Πρέπει να κάνουμε λοιπόν όλα αυτά απαραίτητα. Τώρα, σε περίπτωση των αποφάσεων που έχουν ληφθεί ήδη στην Ευρώπη για να υπάρξει σημαντική ενίσχυση των απαιτήσεων κεφαλαίου για τι ε, τις ενέργειες της αγοράς, ιδίως όταν πρόκειται για τίτλοποίηση, φαίνεται ότι στην Συμφωνία της Βασιλείας 2 δεν είχε ε, αποφασιστεί σωστά Ελπίζουμε ότι σήμερα στις διεθνείς συμφωνίες οι οποίες θα ακολουθήσουμε θα είναι καλύτερα ε, σταθμισμένοι οι κίνδυνοι. Τίθεται όμως και το θέμα της ποιότητας των κεφαλαίων. Θα πρέπει να ενισχύσουμε σταδιακά τις ποιότητες του κεφαλαίου που βρίσκεται στα χαρτοφυλάκια της τράπεζας. Θα πρέπει να μπορέσουμε να έχουμε ένα σκληρό πυρήνα κεφαλαίου που να βασίζεται κυρίως από μετοχές, ή ισοδύναμα κεφάλαια ή αποθεματικό για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε κάποια σταθερότητα. Εγώ πιστεύω λοιπόν ότι προφανώς θα πρέπει να σταθούμε σε μερικά τεχνικά μέτρα, τι ακριβώς θα πρέπει να κάνουμε για να αφαιρέσουμε από το σύνολο αυτό των κεφαλαίων ορισμένα στοιχεία για να λάβουμε υπόψη την αλληλεπίδρασή τους, αλλά νομίζω το βασικό είναι να μπορέσουμε να σταθμίσουμε σωστά και τα μέτρα φερεγγιότητας και τα μέτρα ρευστότητος. Για μένα δεν είναι αντιφατικό το να θέλουμε να αναπτύξουμε τα μία εγγύησεως των ε, καταθέσεων, τα οποία να έχουν ατύχει να να είναι πιο ισχυρά και να έχουν μια εκ των προτέρων δυνατότητα παρέμβασης και να μπορούν να κινηθούν αυτά τα ταμεία εγγυήσεων ετήσι ενός ρυθμιστή για να αντιμετωπίσουν μια δύσκολη κατάσταση προτού αποβεί δραματική. Νομίζω λοιπόν ότι και οι δύο προσεγγίσεις μπορούν να είναι χρήσιμες και εγώ νομίζω ότι Είμαι πολύ κοντά σε αυτό το οποίο διέτρεχε το ερώτημά σας, ότι αν έχουμε καλύτερα ταμεία παρέμβασης χρειαζόμαστε λιγότερη, λιγότερα ίδια κεφάλαια και επομένως απελευθερώνουμε κεφάλαια για τη χρηματοδότηση τη οικονομία. Εγώ δεν είμαι τόσο πεπισμένος γι' αυτό τώρα, για τη σύμβαση της Βασιλείας. Το σύστημα λειτουργήσε τώρα μέχρι στιγμή με μια επιφύλαξη την οποία σας ανέφερα προηγουμένω, που είναι η καθυστέρηση των Ηνωμένων Πολιτειών στο να δεχτούν και να υιοθετήσουν τη Βασιλεία 2, τη Συμφωνία της Βασιλείας 2. Εγώ πιστεύω ότι από τη στιγμή που έχει προετοιμαστεί το σχέδιο της Επιτροπής επί τη βάση της πρότασης της Επιτροπής της Βασιλείας μέχρι το τέλος του έτους, θα πρέπει να αναμείνει την δέσμευση των Ηνωμένων Πολιτειών για την εφαρμογή των κανόνων της Βασιλείας 2 για να μπορέσει μετά να προχωρήσει σε ένα σχέδιο περαιτέρω διευκρίνησης και βελτίωσης του, συστήματο συστήματος αυτού Βασιλεία 2. Προφανώς θα πρέπει να εγκρίνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες την Βασιλεία 2 προτού ο υπόλοιπο κόσμος προχωρήσει σε μια τροποποίηση του συστήματος ε, Βασιλείας 2. Νομίζω λοιπόν ότι έχετε καταλάβει ποια είναι η βασική ιδέα την οποία θέλω να διατυπώσω. Σε ό,τι αφορά τώρα τον τρόπο μετά την έκθεση Λαροζιέρ, με τον οποίο οι ρυθμιστικές αρχές θα μπορούν να εφαρμόσουν κυρώσεις και να έχουν αποτελεσματική ρύθμιση. Για μένα η καλή φόρμουλα, η σωστή φόρμουλα, είναι μια φόρμουλα η οποία σταδιακά, όπως ακριβώς αναφέρεται και στο σχέδιο το οποίο είναι υποσυζήτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ένα ευρωπαϊκό σύστημα χρηματοπιστωτικών ρυθμιστών. Αν δείτε πώς λειτουργεί το σύστημα των ΗΠΑ, που για μένα είναι το καλύτερο τέτοιο σύστημα εποπτείας, το σύστημα που υπάρχει μέσα στα πλαίσια του Federal Reserve. Είναι ένα σύστημα μέσα στο οποίο ο ρυθμιστής δεν βρίσκεται στη Washington. Ο ρυθμιστής βρίσκεται σε κάθε μία από τις τράπεζες της ε, Federal Reserve, σε ό,τι αφορά την τράπεζα της Federal Reserve βρίσκεται τόπου στη Νέα Υόρκη, αντίστοιχα για το Σικάγο, αντίστοιχα στο Σαν Λούι, είναι στο Σαν Λούι και έτσι με τον τρόπο αυτό έχετε ένα πλέγμα ρυθμιστών και φυσικά στη Washington υπάρχει το Συμβούλιο των Διοικητών των Τραπεζών της Federal Reserve που εξασφαλίζει την συνεκτικότητα και αν υπάρξει κάποιο πρόβλημα αναλαμβάνει δράση. Υπάρχει λοιπόν ένα σύστημα το οποίο έχει εσωτερική συνεκτικότητα για αυτό το τμήμα της ρύθμισης γιατί το υπόλοιπο τμήμα του συστήματος είναι λιγότερο συνεκτικό από το ευρωπαϊκό σύστημα. Δεν θα πρέπει να αυτομαστιγωνόμαστε ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την πρόοδο που έχουμε επιτύχει στην ε, Ευρώπη. Πολλές φορές είμαστε σε προπορία εναντί των ΗΠΑ. Πιστεύω όμως ότι το σύστημα αυτό της ε, Federal Reserve, αυτό το ομοσπονδιακό σύστημα, γιατί ομοσπονδιακό είναι, έχει μια σωστή αντιμετώπιση των ε, προβλημάτων. Και αυτό πρέπει να γίνει και σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή να υπάρχουν ρυθμιστέ που γνωρίζουν του παίκτε τη αγορά, τι ιδιαιτερότητε τη αγορά, τι νομικέ ιδιαιτερότητε, αλλά να έχει και μια ενότητα διαχείριση. Περνάμε τώρα στον κύριο Κοφεράτη. Ένα, ένα λεπτό. Και για του φιλελεύθερου, ποιο θα μιλήσει, εντάξει. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ θέλω να ρωτήσω τον ε, προσκεκλημένο μας. Στις πρακτικές εποπτείας και ρύθμισης του συστήματος, ε, τόσο όσον αφορά την εθνική διάσταση, όσο και όσον θα αφορά την ευρωπαϊκή και υπερεθνική διάσταση. Ένα πολύ λεπτό θέμα θα είναι αυτό της διαχείρισης ε, των πληροφοριών. Γνωρίζουμε πόσο μπορούν να χειραγωγηθούν όλες αυτές οι πληροφορίες με όλες τα προβλήματα που κάτι τέτοιο μπορεί να δημιουργήσει. Θα ήθελα λοιπόν να γνωρίζω από εσά ποια θεωρείτε πως θα ήταν ο καλύτερος, μάλλον ποιος θεωρείτε ότι ήταν ο καλύτερος τρόπος, ο πιο αποτελεσματικός ε, για το ολόκληρο το χρηματοπιστωτικό σύστημα, ώστε να διατρέχουμε λιγότερους κινδύνους. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Νουαγέ, χρησιμοποιείτε, τουλάχιστον αυτό άκουσα από την ερμηνεία, λέξεις όπως ευαίσθητος, ισορροπημένος, ε, η σωστό συντονισμός, μήπως ε, ε, υπερβάλλουμε εδώ στην Ευρώπη προσπαθώντας να λύσουμε αμερικανικά προβλήματα και καταλήξουμε σε νομοθεσίες που τελικά εμποδίσουν την αγορά μας. Και τέλος, ε, κατάλαβα σωστά ότι είστε επικριτικός απέναντι στη δημιουργία ενός ταμείου σταθερότητας φερεγγιότητας ή ασφάλισης, αντασφάλισης. Σας ευχαριστώ. Για το ευαίσθητο θέμα της διαχείρισης της πληροφόρησης, νομίζω ότι η αρχή η οποία πρέπει να ανέβει, κατά την άποψή μου, και είναι, κατά την άποψή μου λοιπόν είναι αρκετά σύμμορφη αυτή η ιδέα με, την, με τις εργασίες οι οποίες εκτιλήσονται τώρα για τους κανονισμούς που συζητούνται αυτή τη στιγμή και συνίσταται στο εξή να θεσπίσουμε την αρχή ότι οι αρχές έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνούν όταν τους φανεί απαραίτητο, αλλά δεν έχουν την υποχρέωση κοινοποίηση για τις εργασίες που λαμβάνουν χώρα μέσα σε ένα πλαίσιο το οποίο μπορεί να είναι πιστευτικό. Επομένως, αυτή είναι η ισορροπία μεταξύ καθήκοντος και δικαιώματος σε ό,τι αφορά τους ρυθμιστές. Αυτό νομίζω ότι προβλέπεται και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου. Είναι μια σωστή ισορροπία, θα πρέπει να αφήσουμε κατά περίπτωση την επιλογή του να υπάρξει κοινοποίηση ή όχι ή να υπάρχουν <clears throat> διακριτικές και εμπιστευτικές συζητήσεις και ανταλλαγή μηνυμάτων. Η μόνη μορφή κοινοποίηση και επικοινωνία που μου φαίνεται ότι είναι απαραίτητη, είναι αυτή η οποία λαμβάνει χώρα σε ένα πλαίσιο όπω το σημερινό. Δηλαδή το γεγονό ότι εσεί θα πρέπει να έχετε τακτικέ ακροάσει με τον ε, πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου και φυσικά και η παρουσία του Πρόεδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που είναι ακρογωνίαος λίθος του Ευρωπαϊκού πιστοτικού συστήματος, θα πρέπει και αυτός να μπορεί να σας αναφέρει τα βασικά στοιχεία της δράσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Ό,τι αφορά τώρα την αρκετά δύσκολη και ευαίσθητη ισορροπία, το λεγόμενο fine tuning, που αναφέρθηκε από εσά. Πράγματι νομίζω ότι ορθά κατανοήσατε τα λεγόμενά μου. Αυτό το οποίο προσπάθησα να πω <clears throat> είναι ότι κατά την άποψή μου οι γενικές κατευθύνσεις, οι γενικές επικεφαλίδες των δράσεών μας, όλες οι γενικές γραμμές τις οποίες εγώ έχω συμμετάσχει σαν μέλος των G20 της Επιτροπής της Βασιλείας και του Συμβουλίου για την Σταθερότητα των Πιστοτικών Ιδρυμάτων, όλες αυτές οι κατευθύνσεις αφεαυτών είναι ορθές ή σχεδόν όλες. Αλλά από την άλλη πλευρά το, η στάθμιση η οποία γίνεται Δηλαδή, οι συγκεκριμένες λεπτομεριακές ρυθμίσεις οι οποίες έχουν θεσπιστεί, αν τις ε, αντιμετωπίσουμε όπως έχουν χωρίς να έχουμε μια εξέταση του γενικού πλαισίου, εγώ πιστεύω ότι θα μπορούσαν να θεωρούν υπερβολικές, δεν ανταποκρίνονται στα προβλήματα που έχουμε στην Ευρώπη, ως εκ τούτου μπορούν να είναι και επικίνδυνες. Αυτό λοιπόν νομίζω ότι θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας ότι μπορούν να αποβούν και επικίνδυνες για την υγεία χρηματοδότηση της παγκόσμια και ιδιαίτερα της ευρωπαϊκής οικονομίας. Γι' αυτό χρειάζεται να έχουμε αυτή τη στάθμιση η οποία βασίζεται σε μακροοικονομικά υποδείγματα. Πρέπει να βρούμε το σωστό υπόδειγμα και μετά να παίξουμε με τις παραμέτρους μέχρι να βρούμε την σωστή ισορροπία. Δεν πρέπει να θεωρήσουμε ότι αυτά τα οποία έχουν αποφασιστεί είναι η τελική, ο τελικός λόγος, η τελική λύση. Έχουμε ένα χρόνο για να κάνουμε δοκιμασίες και να προτείνουμε στους νομοθέτες, από την βάση ελπίζω μιας Παγκόσμια συμφωνίας, ένα τρόπο ρύθμισης ο οποίος να είναι ισορροπημένος. Και είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι αντίθετα με τις ΗΠΑ η δική μας οικονομία ευρωπαϊκή χρηματοδοτείται κυρίως από το τραπεζικό σύστημα, ενώ στις ΗΠΑ χρηματοδοτείται κυρίως από την χρηματαγορά. Οπότε έχουμε διαφορετικέ συνθήκε. Για τα ταμεία παρέμβαση, τα ταμεία σταθερότητα, όπω θέλετε να τα λέτε, ναι, πράγματι έχω μια κριτική στάση έναντι τη απόψεω αυτών που λένε ότι πρέπει να υπάρχει ουσιαστικά ένα ασφαλιστικό συμβόλαιο για, την, για τα πιστωτικά ιδρύματα. Φοβάμαι ότι αυτό δημιουργεί ηθικό κίνδυνο. Από την άλλη πλευρά νομίζω ότι τα κεφάλαια εγγυήσεων, και το έχουμε δει αυτό σε πολλά χρόνια, μπορούν να χρησιμοποιούνται προληπτικά. Και είναι μια αντιμετώπιση η οποία έχει λιγότερα αρνητικά στοιχεία και μπορεί να βοηθήσει μικρά και μεγάλα πιστοτικά ιδρύματα χωρίς φαινόμενο κατοφλίου και να είναι πιο λειτουργική κατά την απόψή μου. Κύριος Γκίγκο. Καλημέρα σας κύριε Νουαγέ. Δύο ερωτήματα έχω. Πρώτα απ' όλα, αν κατάλαβα καλά, είπατε ότι όσο πιο στενή είναι η σχέση του ρυθμιστή προς το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, τόσο καλύτερος είναι ο έλεγχος. Και εδώ δίλατε ως παράδειγμα το αμερικανικό σύστημα για να καταδείξετε ότι αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος να οργανωθεί ένα σύστημα ρύθμισης. Εδώ πρέπει να σας πω ότι δεν είμαι ιδιαίτερα πεπισμένο μετά από τις πρόσφατες εμπειρίες που είχαμε. Και ιδίω πιστεύω ότι η εγκύτητα όπως και η απόσταση θα πρέπει να βρίσκονται σε σωστή ισορροπία για να είναι αποτελεσματικός ο έλεγχος. Δεύτερο, θα ήθελα να σας θέσω το εξής ερώτημα. Αν μέσω αυτής της κρίσης έχουμε διδαχθεί ότι η χρηματοοικονομική κρίση οδηγεί σε μια εξωτερικότητα, σε πρόσθετο κόστος για όλη την οικονομία. Μήπως θα μπορούσαμε να έχουμε ένα Ευρωπαϊκό Ταμείο το οποίο χρηματοδοτείται από το χρηματοοικονομικό σύστημα για να υπάρξει σωστή κατανομή αυτού του άχθους και κατά την άποψή σας πώς θα έπρεπε να οργανωθεί και πώς θα έπρεπε να λάβει η χώρα μια τέτοια κατανομή του κόστους. Ο κύριος Μποργέζιου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Δίκητα πέραν των ασαφών κανόνων, υπάρχουν και πολλά στοιχεία της χρηματοοικονομικής καινοτομίας που οδήγησαν στην κατάσταση αυτή που αντιμετωπίσαμε ενός σκιώδους τραπεζικού συστήματος με διάφορα χρηματοοικονομικά προϊόντα τα οποία εκφεύγουν σε μεγάλο βαθμό από τη ρύθμιση. αναφερθήκατε σε καινοτόμα συστήματα ελέγχου και αναφερθήκατε φυσικά και στα λογιστικά πρότυπα υψηλής ποιότητας. Αλλά το ερώτημά μου είναι το εξής. Αυτό το σκιώδες τραπεζικό σύστημα, το οποίο έχει δημιουργήσει όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία γνωρίζουμε και μπορεί να δημιουργήσει νέες χρηματοοικονομικές φούσκες στο μέλλον. Αυτό το σύστημα δεν λειτουργεί ακόμα και ποια είναι τα μέτρα τα οποία είναι απαραίτητα και κατεπήγοντα, τα οποία θεωρείται ότι πρέπει να ληφθούν εναντίον αυτής της δραστηριότητας του σκιώδου του τραπεζικού συστήματος για να αποφύγουμε και τους κινδύνους που προέρχονται από αυτό, γιατί να υπενθυμίσουμε και το ότι όλο αυτό το πλέγμα των, ε, των ε, χρεών που προέρχεται από τα εκτός ισολογισμού εργαλεία των τραπεζών συνδέεται με αυτά τα προβλήματα και τελικά την ύφη την πληρώνουν οι, οι καταναλωτές και οι φορολογούμενοι. Θα πρέπει να συνεχίσουμε εμείς να πληρώνουμε λοιπόν για όλα αυτά τα οποία γίνονται από την κερδοσκοπία των ε, χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ίσως δεν εκφράστηκα σωστά. Είπα ότι όσο πιο κοντά είναι ο ρυθμιστής με το πιστοτικό ίδρυμα, αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρχει ένας ρυθμιστής σε κάθε πόλη, σε κάθε περιοχή και να έχουμε παραγωγικά 300 ρυθμιστές σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό το οποίο ήθελα να τονίσω είναι ότι με το να συγκεντρώσουμε σε ένα μονάχα γεωγραφικό τόπο, τις ομάδες οι οποίες προβαίνουν σε αναλύσεις και επιθεωρήσεις για να ρυθμίσουμε τον αχανή ουσιαστικά ευρωπαϊκό χρηματοοικονομικό χώρο δεν θα ήταν πρόσφορο. Νομίζω ότι η πρόταση της έκθεσης Λαροζιέρ που λέει ας κρατήσουμε τους ρυθμιστές εκεί που βρίσκονται αλλά ας τους συνδέσουμε μέσα σε ένα σύστημα όπως το σύστημα του Federal Reserve στις Ηνωμένες Πολιτείες με τη δυνατότητα να υπάρξει μια συνεκτικότητα και μια ενοποίηση των μεθοδολογιών και να υπάρχει μια κοινή πολιτική εφαρμογή των ρυθμίσεων, αυτό για την Ευρώπη νομίζω ότι είναι πιο αποτελεσματικό. Αυτή είναι η ανάλυση την οποία εγώ υποστηρίζω. Δεύτερον, σε ό,τι αφορά το λεγόμενο εξωτερικό κόστος το οποίο προκύπτει την κρίση. Και όσον αφορά την δημιουργία ενός ταμείου. Αυτό δεν με ενοχλεί, αυτό με ενοχλεί είναι ότι δεν θέλω να φτιαχτεί ένας κατάλογος συστημικών ε, ε, ιδρυμάτων. Υπάρχουν τράπεζες ε, που δεν θέλω να αναφέρω τώρα ονόματα, αλλά σίγουρα δεν θα είχαν μπει μέσα στο κατάλογο των ε, συστημικών κινδύνων πριν από τέσσερα χρόνια. Αυτό δημιουργεί ένα πρόβλημα. Θα πούμε, να πούμε δηλαδή ότι υπάρχουν 20 ιδρύματα στην Ευρώπη που ποτέ δεν πρόκειται να, να, να, και θα τους εξασφαλίσουμε και αυτό που θα τους κάνουμε είναι να τους βάλουμε να πληρώνουν ένα πρίμα μια ανασφάλεια. Δηλαδή το ίδιο πράγμα είναι. Εγώ το λέω αυτό ταμείο εγγυήσεων, γιατί έχω αυτή την εμπειρία από τη Γαλλία, ταμείο εγγυήσεων των καταθέσεων που δεν είναι εξαιρετικά ε, στεναρόλα. αλλά υπάρχουν άλλες χώρες στην Ευρώπη που έχουν πιο δυνατά τέτοια ταμεία αλλά εν πάση περιπτώσει εξάντε πρόληψη για την ε, αντιμετώπιση της κατάστασης ε, θα μπορούσε να γίνει από τον επόπτη, δηλαδή από μένα τον ίδιο. Και έχουμε εξουσίες που μπορεί να οδηγήσουν μέχρι και την ε, απόλυση ενός ε, μάνατζερ και του Διοικητικού Συμβουλίου και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν η δημιουργία ενός ταμείου ε, που θα χρηματοδοτείται από το τραπεζικό τομέα και από ένα φόρο ε, που θα επιβληθεί σε αυτό. Συμφωνώ με τις αναλύσεις σας και αυτό είναι ο τρόπος με τον οποίο εγώ σκέφτομαι τα πράγματα και τέλος όσον αφορά το θέμα του τι δεν είναι ένα τραπεζικό σύστημα, το σύστημα, το σκιώδες σύστημα όπως μεταφράστηκε, η απάντηση δεν μπορεί να δοθεί με μια λέξη. Γιατί υπάρχουν πολλά σημεία που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Την εδραίωση, την παγίωση των ε, μέσων που δίνει η τράπεζα, τον αριθμό των λογιστών που χρησιμοποιούν αυτά τα οχήματα εκτός προϋπολογισμού, εκτός ισολογισμού, συγγνώμη, ε, Αυτά άλλαξαν ε, και στις ΗΠΑ με βάση το, τα προγράμματα δράσης για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες. Ε, θα πρέπει εξίσου να ληφθούν υπόψη οι δεσμεύσεις εκτός ισολογισμού και η χρήση αυτών των ε, πολύ ιδιαίτερων οχημάτων είναι κάτι το οποίο πρέπει να γίνει μέσω του πυλώνα 2. Προσπαθούμε σήμερα να το λάβουμε υπόψη όσο γίνεται περισσότερο ακόμη περισσότερο δηλαδή από πριν την κρίση ε, ε, ώστε να αναπτυχθούν αυτές οι εξωτραπεζικές δραστηριότητες που έχουν όντως αυτές τις επικίνδυνες επιπτώσεις που αναφέρατε. Ευχαριστώ. Νομίζω πως στάσαμε στο τέλος της πρώτης, ε, του πρώτου τμήματος αυτής της ακρόσης. Ευχαριστώ πολύ που δεχτήκατε την πρόσκλησή μας και που απαντήσατε στις ερωτήσεις. Υπάρχουν ακόμα περισσότερες βέβαια, αλλά δεν έχουμε άλλο χρόνο. Σας ευχαριστούμε που ήρθατε. Περνάμε λοιπόν στο πρώτο πάνελ. Κύριε Σάνιο, σα δίνω τον λόγο. Έχετε 15 λεπτά να τα καταφέρετε και σε 12, ακόμη το καλύτερο. Αυτό δύσκολο, δύσκολο. Θα προσπαθήσω. Δεν θα ξεκινήσουμε πάλι με τους ουρανούς που πέφτουν στο κεφάλι μας. Όσοι έχουν δει τον ουρανό να πέφτει στο κεφάλι τους, και εγώ μεταξύ αυτών, πιστεύουν πως ε, οτιδήποτε πλέον μπορεί να συμβεί στις ε, χρηματαγορές. Και βεβαίως το να ζούμε μονίμως με ένα φόβο της αποκαλύψεως είναι κάτι το ανθιγεινό και απαράδεκτο. Αυτό το οποίο βλέπουμε και χρειαζόμαστε τώρα είναι μια αλλαγή καθεστώτος όπως λέγεται, μια θεμελιώδης επανεξέταση του συστήματος που έχει πλέον αποσταθεροποιηθεί μοιραία πριν, όμως βιαστείτε με το να αλλάξετε τις παραμέτρους ενός απειχαιωμένου συστήματος, πρέπει πρώτα απ' όλα να γίνει μια σοβαρή ανάλυση των αδυναμιών και να δούμε ποιοι είναι οι παράγοντες εκείνοι που μπορούν να κάνουν μια απλή κρίση καταστροφή. Το ρυθμιστικό πλαίσιο έχει υποστεί κριτική, η οποία βεβαίω είναι δίκαιη. Η κρίση αυτή απέδειξε πέραν πάσης αμφιβολίας πόσο ανεπαρκές και, λανθασμένο, και ένα ανεπαρκές και λανθασμένο ρυθμιστικό πλαίσιο μπορεί να επιφέρει μόνιμη βλάβη στο χρηματοοικονομικό σύστημα. Αυτό το οποίο είχαμε τα τελευταία 20 χρόνια ήταν οι κανονισμοί σαν ελβετικό τυρί, δηλαδή διεθνή πρότυπα τα οποία κατά βάση ήταν σωστά αλλά ήταν γεμάτα τρύπε. Επίση, υπήρχαν και υπάρχουν ακόμα μεγάλοι τομεί, οι οποίοι δεν υφίστανται καθόλου εποπτεία. ω αποτέλεσμα αυτού ακόμα και εταιρείε υπό στενό έλεγχο μπόρεσαν κάποιου κινδύνου του να του αποκρύψουν τελείω από τι εποπτικέ αρχές εκμεταλλευόμενε στιγνά τα παραθυράκια αυτά. Θα ήθελα να εξηγήσω λίγο τι εννοώ εδώ πέρα. Ένα. Εδώ πέρα. Η Βασιλεία 1 το διεθνές ε, πρότυπο φερεγγιότητας του 1988 που συμπληρώθηκε από ένα στοιχείο κινδύνου των αγορών ε, το 1996 είχε ως στόχο το να μην επεκτείνονται αφρόνως οι αγορές ε, διασφαλίζοντας πως οποιαδήποτε τέτοια επέκταση σήμαινε και κάποια ανάλογη επέκταση στο κεφάλαιο. Όμως άφηνε κάποια παραθυράκια τα οποία χρησιμοποίησαν οι τράπεζες για να υποβαθμίσουν τι βασικές αυτές διατάξει. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η έλλειψη κεφαλαίου που ε, υπήρχε ως απέτηση για τους κινδύνους στα βιβλία που κρατούσαν οι τράπεζες όσον αφορά τίτλοποιημένες ε, υποχρεώσεις, όπως χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν τα στεγαστικά δανεία, τα λεγόμενα subprime στην Αμερική. Ένα άλλο παραθυράκι ήταν εξίσου σοβαρό, σοβαρό παραδείγματο χάρη δεν χρειάζονταν να έχουν κεφάλαια τα οποία κρατούσαν τράπεζε όταν είχαν μακροπρόθεσμε δεσμεύσει με αρχική οριμότητα μέχρι ένα έτο. Και το αποτέλεσμα ήταν ότι γίνονταν συνεχή δανεισμό με μια βάση κυλιόμενη 364 ημερών και αυτά κρύβονταν πίσω από το σχετικά κακό όνομα της διευκόνησης ρευστότητας και τελικά αναγκάστηκαν να λάβουν τις ευθύνε για όλα αυτά όταν πλέον δεν μπορούσαν να μετακυλήσουν πλέον. Οπότε υπήρχε ένας πάρα πολύ μεγάλος κίνδυνος χρεοκοπίας από αυτό. Ένα, μια άλλη παραγωγή του ιδίου παιχνιδιού ήταν τα λεγόμενα special purpose vehicles όπου δισεκατομμύρια τέτοια ε, τίτλοποιημένα χρεόγραφα είχαν αποθηκευτεί και το βασικό ερώτημα ήταν εάν θα έπρεπε να ενσωματωθούν αυτά στις τράπεζες ή όχι. Και η απάντηση προήλθε από τα μία ακριβή διεθνή λογιστικά πρότυπα, τα οποία έκαναν αποδεκτά οι ρυθμιστικές αρχές. Στην περίπτωση αυτή ε, πρόκειτο για το διεθνές λογιστικό πρότυπο 27 μαζί με την ερμηνεία την λεγόμενη 12 που ήταν η πηγή του προβλήματος. Για όσους βεβαίως σχεδίασαν αυτά τα μέσα με έναν αρκετά έξυπνο τρόπο, οι ελεγκτές ε, βεβαίωναν πως ε, ήταν ε, δική τους επιλογή να αποφασίσουν εάν θα τα ενσωματώσουν ή όχι και στο τέλος αυτή η ενσωμάτωση δημιούργησε το μεγαλύτερο αυτό σκιώδες το λεγόμενο τραπεζικό σύστημα, δηλαδή μια σαθρή δομή η οποία δεν στηρίζει καθόλου από κεφάλαιο, η οποία βέβαια μπορούσε να καταρρεύσει υπό δύσκολε συνθήκε, όπως και τελικά συνέβη. όσοι υπέθονταν πως, υπέθονταν πως ε, έτσι μπορούσαν να, κάνουν, να επιχειρήσουν χωρίς κίνδυνο βεβαίως έκαναν λάθος κάτι το οποίο αποδείχθηκε στο τέλος και όσοι αγόραζαν τα ε, χρεόγραφα τα οποία εκδίδαν τα λεγόμενα special purpose vehicles για αναχρηματοδότηση βεβαίως δεν είχαν σκοπό να αναλάβουν τον κίνδυνο των, των επενδύσεων αυτών και εξανάγκασαν τις τράπεζες που χειρίζονταν αυτά τα special purpose vehicles να αναλάβουν τους ε, κινδύνους. Βεβαίως, όπως ε, όλοι γνωρίζουμε, αν δεν γινόταν κάτι τέτοιο θα είχαμε καταστροφικές συνέπειες και είχαμε επιτρέψει σε αυτό το σημείο να είναι τεράστιες οι διαστάσεις και οι εποπτικές αρχές δεν επιτέλεσαν την βασική τους λειτουργία, δηλαδή να, να περιορίσουν την πιστοτική επέκταση. Το αποτέλεσμα βεβαίω ήταν η τιτλοποίηση σε υπόθηκα χρεόγραφα και μετά αυτά μετατράπηκαν όπως σας είπα σε υπόθηκα χρεόγραφα και για να χειροτερεύσουν ακόμα τα πράγματα, το τελικό αποτέλεσμα ήταν κάτι περισσότερο από μια τέτοια απλή ε, δομή. Ε, πρόκειται για συνεχή βήματα τίτλοποίησης με ονόματα όπως CDO στο τράγωνο και CDO στον κύβο και καθώς αυτά τα προϊόντα γίνονταν όλο και πιο περίπλοκα πλέον δεν υπήρχε καμία δυνατότητα οι αγοραστές να τα αντιληφθούν όταν αγοράζουν τέτοια προϊόντα οι αγοραστές θα πρέπει να είναι σε θέση να μπορέσουν να αξιολογήσουν στο δυνατόν καλύτερα τον εγγενή κίνδυνο ανταυτού οι αγοραστές αποπροσανατολίζονταν από το πόσο ομιχλώδη ήταν αυτά τα προϊόντα και δεν μπορούσαν να αντιληφθούν τον πραγματικό κινδυνοπόριζαν τα δεδομένα. Στο τέλος δεν μπορούσαν να διακρίνουν με το, μεταξύ του τι ήταν πραγματικό και του τι ήταν απάτη. Οπότε έπεφταν θύμα των διαφόρων τεχνασμάτων που χρησιμοποιούνταν για να κρύψουν την βασική χαμηλή ποιότητα των ε, τίτλων αυτών, δηλαδή τα ε, κακά θα λέγαμε στεγαστικά δάνεια. Πώς μπόρεσε λοιπόν αυτή η απάτη να συνεχιστεί για τόσα χρόνια. Η απάντηση ήταν τόσο απλή. Από τις ΙΠΑ όπου είχαν ξεκινήσει όλα αυτά δεν υπήρχε αρκετή εποπτεία και η χρηματοοικονομική αυτή κρίση οπωσδήποτε γεννήθηκε στις ΙΠΑ ε, η, απο... η απουσία πανεθνικής ε, εποπτείας της ΕΠΑ που θα στηρίζονταν από αποτελεσματική επιτήρηση της αγοράς οδήγησε σε δανεισμό πέρα από κάθε όριος και σε κλίμακα που δεν είχε ξαναδεί ποτέ ο κόσμος. Οπότε από πλευράς των αρχικών εκδοτών αυτών των ε, τίτλων δεν υπήρχε ανάγκη να αξιολογηθούν σωστά. Οι κίνδυνοι καθώς μπορούσαν να τους υλοποιήσουν και να τους δώσουν μετά σε ανύποπτους, θα λέγαμε, αγοραστές. Εάν φτάσουμε ξανά σε τέτοια τιτλοποίηση, γιατί αυτή τη στιγμή πρόκειται για κάτι το τελείως νεκρό, πρέπει να μην υπάρχουν πλέον αυτά τα περίεργα. Αφύσικα κίνητρα πρέπει πλέον και αυτοί οι οποίοι τα δημιουργούν να έχουν κάποιο συμφέρον στην όλη υπόθεση. Επίσης όλοι οι συμμετέχοντες στην αγορά και αυτοί οι οποίοι τα δημιουργούν και όσοι τους βοηθούν πρέπει να υποστούν αυστηρό έλεγχο στις χρηματαγορές η ρύθμιση είναι το μόνο αποτελεσματικό εργαλείο περιορισμού της ανθρώπινης ε, συμπεριφοράς, ε, ειδικά της απληστίας. Σε αυτό το σημείο βεβαίως η ιστορία της τηλεοποίησης δεν μπορεί να υποθεί χωρίς να αναφέρουμε στις υπηρεσίες ε, αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας που ανήκουν επίσης σε αυτούς οι οποίοι συμμετέχουν χωρά και δεν υφίστανται καμία εποπτεία. Υποτίμησαν σε μεγάλο βαθμό το συστημικό κίνδυνο την κατάρρευση δηλαδή της ε, αγοράς των ακινήτων στις ΙΠΑ συνολικά. Τα μαθηματικά τους ε, μοντέλα δούλευαν υπό την υπόθεση πως ε, οι κίνδυνοι αυτοί δεν συνδέονταν μεταξύ τους, κάτι το οποίο βεβαίως αποδείχθηκε τελικά πως ήταν υπεραισιόδοξο και λανθασμένο. Ένα μεγάλο σημαντικό ζήτημα είναι οι αγορές των πιστοτικών παραγόγων όπου εμπορεύονταν αυτά τα προϊόντα όπου υποτίθεται ότι θα γίνονταν η διάχυση του κινδύνου υπομορφή ειδικά των credit default swap συμφωνιών ανταλλαγής κινδύνων ανθέτησης. Όλα αυτά βεβαίω είναι ένα περίπλοκο ασφαλιστικό προϊόν, πολύ επικίνδυνο και δεν υφίσταται σε καμία ρύθμιση. Κατά κανόνα υπάρχει μια αλυσίδα τέτοιων προϊόνων. Βεβαίως λόγω της έλλειψης αναγκάστηκε η Αμερικανική κυβέρνηση όντω να σώσει εταιρείε που έπαιζαν σε αυτέ τι αγορέ, κυρίω δηλαδή την ασφαλιστική εταιρεία AEG, αλλιώ το διεθνέ χρηματοπιστωτικό σύστημα κυριολεκτικά θα κατέρε εν μία νυχτή. Οπότε υπάρχει μια ανάγκη να έχουμε νέε αρμοδιότητε των ελεγκτικών αρχών. Και αφού κατέρευσε και η Lehman Brothers, ήταν πλέον σαφέ πω καμία τράπεζα η οποία θεωρούνταν κεντρική για το σύστημα δεν θα επιτρέπονταν πλέον να καταρρεύσει καθώ αυτό θα οδηγούσε στην κατάρρευση ολόκληρου του συστήματο κάτι το οποίο πλέον λέμε με την φράση ότι είναι πολύ μεγάλη ή πολύ διασυνδεδεμένη για να καταρρεύσει. Η ύπαρξη αυτής της ε, ασφάλειας αλλάζει την συμπεριφορά όσον αφορά την ανάληψη κινδύνου. Ο ηθικός αυτός λοιπόν κίνδυνος αποτελεί σημαντικό σημαντική απειλή στην σταθερότητα και θα πρέπει να βρούμε τρόπους να λύσουμε αυτό το φαινομενικά άλλο το πρόβλημα. Υπάρχουν πολλές λογικές λογικές προτάσεις. Τώρα το εάν είναι τελικά βιώσιμες είναι κάτι που θα πρέπει να δούμε, αλλά πρέπει να συζητηθεί. Εγώ προσωπικά είμαι υπέρ του να έχουμε ένα καθεστώς το οποίο θα καταστήσει δυνατόν το να κλείνουν τράπεζες οι οποίες είναι προβληματικές χωρίς να μεταδίδεται το πρόβλημα αλλού. Καθώ μία τράπεζα, αν κλείσει με αυτόν τον τρόπο, αυτομάτω το θέμα του ηθικού κινδύνου εξαφανίζεται. Επιπλέον, οι τράπεζε οι οποίε δεν θα είναι σίγουρε ότι θα διασωθούν, θα είναι πολύ προσεκτικέ στην διαφορά του, Αυτό το οποίο χρειαζόμαστε λοιπόν είναι μία διεθνή ε, συμφωνία για ένα σύστημα επίλυση, κατά το οποίο δεν ξέρω πω είναι όνειρο απατηλό, καθώ τα τελευταία 50 χρόνια έχουν δείξει πώ οι χώρε δεν θέλουν να θέσουν υπό διεθνή υποπτία την εθνική τους νομοθεσία περί χρεοκοπίας. Κυρίες και κύριοι, ο χρηματοοικονομικός κόσμος βεβαίω πάντα περνάει περίοδο τρέλα και μόλις είδαμε μια τέτοια και θα συνεχίσει να το κάνει αυτό ως ε, ρυθμιστικές αρχέ δεν μπορούμε να προβλέψουμε ποια θα είναι η μελλοντική συμπεριφορά των αγορών αλλά πρέπει να παρακολουθούμε στενά του συμμετέχοντες στην αγορά. Μόλι δείξουν ξανά σημάδια ότι αναλαμβάνουν υπερβολικού κινδύνου, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τα νέα μας εργαλεία της άμεσης διορθωτικής δράσης και να τα χρησιμοποιήσουμε αμέσως. Το αποτέλεσμα δεν θα τους αρέσει βεβαίως. Βεβαίως, όπως λέει και ένα γερμανικό ποίημα, και εδώ πέρα τελειώνω, μπορεί κάποιος βεβαίως, η τρέλα είναι σύντομη, αλλά μπορεί κάποιος να μετανιώσει με την ησυχία του. Σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ για την ομιλία η οποία είχε και στοιχεία αυτοκριτική για τον κλάδο σας. Θα ήθελα τώρα να δεχτούμε κάποιες ερωτήσεις. Πρώτα πριν περάσουμε βεβαίω και στους λοιπούς ομιλητές, την κυρία Μπετίνα Κόρβε Βούντερερ. Καλημέρα σας κύριε Πρόεδρε, καλημέρα αγαπητοί βουλευτέ. Um, let me σχόλιά μου, με μια σύνοψη των κυρίων αιτίων της χρηματοοικονομικής κρίσης που μετετράψει η οικονομική κρίση. Επα... Ανεπαρκής έλεγχος οδήγησε σε υπερβολική χρήση μόχλευσης και εργαλείων μόχλευσης αυτή η υπερβολική μόχλευση οδήγησε σε υπερβολική ρευστότητα και ροές ρευστότητας μεταξύ τραπεζών και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και τόσο τα υποδείγματα όσο και οι ρυθμιστές δεν είχαν εκτιμήσει σωστά την έκταση αυτού του κινδύνου. Αυτή η ρευστότητα προέρχεται και από τις κεντρικές τράπεζες και ιδίω στι ΗΠΑ και κεντρικέ τράπεζε των ΗΠΑ, αλλά και από κυβερνήσει μέσω των δημοσίων ελλημάτων. Σε ορισμένε χώρε είδαμε να υπάρχει ανεπαρκέ περιβάλλον ρύθμιση και πρέπει να θυμόμαστε ότι παραδείγματο χάρη στι ΗΠΑ μόνο 25% των χρηματοπιστωτικών οντοτήτων υπόκεινται σε αυτό το ρυθμιστικό πλαίσιο, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως από τον κύριο Σάνιο. Αλλά αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα το οποίο πρέπει να το τονίσω. Επίσης υπήρξε υπερβολική εμπιστοσύνη σε μαθηματικά μοντέλα, συγκρούσεις συμφερόντων επίσης, συνέβαλαν και αυτές σε ανεπαρκή εκτίμηση κινδύνου από τις εταιρείες πιστοληπτικής αξιολόγησης. Και πρέπει να τονίσω επίσης και τα αδιαφανή και όχι αρκετά εναρμονισμένα λογιστικά πρότυπα τα οποία σε ορισμένε περιπτώσεις οδήγησαν σε υπερκυκλική συμπεριφορά. Έρχομαι τώρα σε ένα άλλο σημαντικό τομέα αιτίων που θα ήθελα να αναφέρω. Η κρίση οφείλεται επίσης και σε μεγάλο βαθμό σε ελλείψεις σε ό,τι αφορά την διακυβέρνηση των επιχειρήσεων. Υπήρξε ανεπαρκής διαχείριση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού καθώς και της ρευστότητας. Και επίσης υπήρξε ανεπαρκής εκτίμηση, τιμολόγηση και αντιμετώπιση των, ε, των κινδύνων. Επίσης η βραχυπρόθεσμη ουσιαστικά αποζημίωση και των ε, στελεχών και τα συστήματα κινήτων. Επίση, το γεγονό ότι δεν υπήρξαν αρκετέ ικανότητες και εμπειρία στον τομέα τη διαχείριση κινδύνου και επίση και τρόποι συμμόρφωση στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Επίση όμω θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι υπήρχε μία πληθώρα παικτών στην αγορά που όλοι προσπαθούσαν να επιτύχουν μη ρεαλιστικές αποδόσεις χωρίς να σκέφτονται συγχρόνως τον κίνδυνο ο οποίος συνοδεύει τέτοιου είδου υψηλές αποδόσεις. Πρέπει να αναφέρω επίσης ότι υπάρχουν ακόμα οργανώσεις καταναλωτών που προωθούν τις χαμηλότερες τιμές και τις ε, υψηλότερες αποδόσεις, χωρίς όμως να λαμβάνει υπόψη τον σχετικό κίνδυνο. Έρχομαι σε κάποιες γενικές παρατηρήσεις τώρα. Αυτό το οποίο είδαμε είναι ότι ο χρηματοοικονομικός τομέας αντιμετωπίστηκε διαφορετικά σε διάφορες χώρες μπορείτε να το καταμετρήσετε στο, στο ποσοστό των ενεργειών διασώσεων, του κόστους διάσωσης μάλλον προς το ΑΕΠ, που ήταν από κάτω του 1% μέχρι ε, διψήφιους αριθμούς. Επίσης, ο τομέας ασφαλίσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν πιο, απεδείχθη πιο σταθερός από τον, από τον τραπεζικό τομέα και επίσης η ποικιλία αρμοδιοτήτων και ποιότητα των αριθμιστών οδήγησε και αυτή σε μεγάλες διαφορές μεταξύ των φορέων αυτών. Α σταθούμε τώρα στα εργαλεία ρύθμιση. Θα ήθελα να τα ταξινομήσω σε τέσσερα η οργάνωση και οι αρχές της ρύθμισης, τα ποσοτικά, οι ποσοτικές απαιτήσει φερεγγιότητος, η προστασία των επενδυτών και των καταναλωτών και φυσικά και η διακυβέρνηση των επιχειρήσεων. Νομίζω επίσης ότι η χρηματοοικονομική κρίση κατέδειξε ότι είναι απαραίτητο να υπάρξει ισχυρό συντονισμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ότι η ρύθμιση και η υποπτία σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα πρέπει να γίνεται σε στενή συνεργασία με του εθνικού επόπτε η εποπτεία θα πρέπει να βασίζεται και σε ορισμένες βασικές αρχές. Τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι μια ιδιαίτερα κυριολεκτική και σχολαστική ερμηνεία των ε, προτύπων λογιστικής μπορεί να οδηγήσει σε υπερκυκλική συμπεριφορά η οποία οδηγεί σε κρίση. Νομίζω ότι οι οργανωτικές αρχές της εποπτείας θα πρέπει να λάβουν υπόψη και τις σαφείς διαφορές στο επιχειρηματικό μοντέλο μεταξύ του τραπεζικού και του ασφαλιστικού τομέα. Αυτό το οποίο χρειαζόμαστε στην πράξη είναι αποτελεσματική ρύθμιση χωρίς υπερβολική γραφειοκρατία και χωρίς ασυνάρτητες απαιτήσει για την ε, παροχή εκθέσεων. Οι αρχές της ρυθμισής θα πρέπει να μεταφράζονται σε ποσοτικές απαιτήσει φερεγγιότητας. Εδώ θα πρέπει να θέσουμε κάποια ερωτήματα σε σχέση με αυτές τις ποσοτικές απαιτήσεις για τη φεραγιότητα. Η... Τα ποσοστά κεφαλαίου, τα ποσοστά αποθεματικού δηλαδή κεφαλαίου, θα πρέπει να αντιμετωπίζουν καλύτερα τους κινδύνους της αγοράς, τους κινδύνους των spread και τους κινδύνους ρευστότητος. Θα πρέπει να υπάρχει επίσης δοκιμασία σε σχέση με τα ε, οχήματα εκτός ισολογισμού και θέλουμε να εξετάσουμε επίσης κατά πόσο ορισμένε κατηγορίες ενεργητικού είναι επαρκείς για να θεωρούνται στοιχεία εγγύσεως. Και επίσης κανόνες για την διαχείριση στοιχείων ενεργητικού και παθητικού για να μην υπάρχει υπερβολική βραχυπρόθεσμη αναχρηματοδότηση μακροπρόθεσμης ε, δανειοδότησης. <clears throat> Είναι απαραίτητο λοιπόν να υπάρξει μια συγκεκριμένη ερωτη... απάντηση στα αυτά τα ερωτήματα για να υπάρξει μια σωστή ισορροπία μεταξύ απαιτήσεων κεφαλαίου και της απαραίτητη μακροχρόνια ανταγωνιστικότητα των χρηματοοικονομικών μα ιδρυμάτων σε παγκόσμιο επίπεδο. Ένα τρίτο στοιχείο που αφορά και πάλι τη ρύθμιση είναι η προστασία των καταναλωτών και των επενδυτών. Είναι απαραίτητο να υπάρξει επάρκεια των προϊόντων αλλά και διαφάνεια των προϊόντων, δηλαδή να υπάρχει σαφήνεια σε σχέση με τη σχέση κινδύνου απόδοσης για αυτά τα προϊόντα. Αυτό αφορά όλα τα προϊόντα, είτε είναι καταναλωτική πίστη, ενυπόθηκα δάνεια ή πολύπλοκα χρηματοοικονομικά εργαλεία. Ο ρόλος των ε, εταιριών πιστοληπτικής αξιολόγησης θα πρέπει να γίνει σαφέστερος, να εξασφαλιστεί η διαφάνειά τους, να αποφευθούν συγκρούσεις συμφέροντος και να υπάρχουν τα κατάλληλα στοιχεία δεξιοτήτων σε αυτές τις ε, επιχειρήσεις. Είναι απαραίτητο επίσης να εξασφαλίσουμε καλύτερη προστασία των καταναλωτών <clears throat> και επίσης οι πελάτες του ε, πιστοτικού συστήματος πρέπει να ξέρουν ότι η μεγαλύτερη απόδοση συνδέεται με μεγαλύτερους κινδύνους. Μας ενδιαφέρει επίσης η ευκυβερνησία των επιχειρήσεων. Εγώ είμαι πεπισμένη πρέπει να βελτιώσουμε τη λειτουργία αξιολόγησης κινδύνου, διαχείρισης κινδύνου και συμμόρφωσης στα χρηματοπιστωτικά α, ιδρύματα. Θα πρέπει να είναι ένα τμήμα του γενετικού υλικού κατά κάποιο τρόπο των χρηματοπιστωτικών οργανώσεων. Δηλαδή δεν μπορεί να είναι απομονωμένη η διαχείριση του κινδύνου επί τη βάση υψηλού επίπεδου μαθηματικών μοντέλων που απλώς δίνουν αποτέλεσμα. Η διαχείριση κινδύνου θα πρέπει να είναι μια κουλτούρα μέσα σε ένα χρηματοπιστωτικό ε, ίδρυμα που επηρεάζει όλες τις αποφάσεις που λαμβάνουν σε καθημερινό επίπεδο σε ένα τέτοιο φορέα. Χρειαζόμαστε επίσης διαφανείς και εναρμονισμένους κανόνες λογιστικής για να υπάρχει καλύτερη αξιολόγηση κινδύνου μεταξύ χωρών και μεταξύ τομέων του συστήματος. Επίσης χρειάζονται αρχές για την αποζημίωση. Να εξασφαλίσουμε ότι γίνονται με τρόπο ο οποίος είναι διάφανος, να περιλαμβάνουν στόχους και επίσης να υπάρχουν και συστήματα αμοιβή των στελεχών τα οποία να μπορούν να αναβληθούν στην εφαρμογή τους. Είναι απαραίτητο για μένα λοιπόν να βασίζονται όλα αυτά σε κοινέ ηθικές αρχέ, και εδώ θέλω να υποστηρίξω ότι πρέπει να επανέλθουμε σε μια ευκυβερνησία που να βασίζεται σε κοινέ αρχές. εν κατακλείδη. Χρειαζόμαστε μια καλύτερα συντονισμένη και καλύτερα σταθμισμένη εποπτεία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η χρηματοοικονομική εποπτεία, η εποπτεία αφαιρεγιότητα και η προστασία των καταναλωτών πρέπει να γίνεται με ένα εναρμονισμένο και συντονισμένο τρόπο. Η ευκυβερνησία των επιχειρήσεων πρέπει να βασίζεται σε σαφεί ειδικέ αρχέ και χρειαζόμαστε Νομίζω ότι αυτό φαίνεται από τη σημερινή συνεδρίαση. Χρειαζόμαστε συνεχή και ενισχυμένο διαλόγο μεταξύ των πολιτικών, των υποπτικών αρχών και των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Ευχαριστώ. Disclaimer. Σας ευχαριστώ που παραμείνετε στα πλαίσια του χρόνου σας. Ερχόμαστε στον τελευταίο ομιλητή του πρώτου πάνελ, τον Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ μπορώ να είμαι συγκεκριτικά σύντομο, γιατί δεν χρειάζεται να επαναλάβω όλα όσα είπαν πολλοί από τους συναδέλφους. Καθώ φαίνεται να υπάρχει γενικά συνένεση. Να αρχίσω με το τίτλο. Στο ποιο βαθμό δηλαδή η οι ρυθμίσεις και η εποπτεία μάλλον ε, απέτυχαν να αντιμετωπίσουν, να εμποδίσουν την κρίση. Θα θέσω λοιπόν το ρητορικό ερώτημα σε ποιο βαθμό η αστυνομία και ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας προλαμβάνουν τα τροχαία ατυχήματα. Βέβαια ε, παίζουν κάποιο ρόλο, αλλά ο υπεύθυνος είναι ο οδηγός από τα όσα ακούσαμε σήμερα, επιβεβαιώνεται σε μεγάλο βαθμό αυτό που πολλοί κόσμος πιστεύει, πως η εποπτεία και η ρύθμιση σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά και σε ευρωπαϊκό κατά επίπεδο, δεν ήταν καλά προσαρμοσμένες στην πραγματικότητα μιας παγκοσμιοποιημένης αγοράς, δεν ήταν καλά προσαρμοσμένες σε περίπλοκα προγράμματα, προϊόντα και προφανώς δεν ήταν προσαρμοσμένες στην για τα μη εποπτευόμενα προϊόντα και τα μη ρυθμισμένα τμήματα της αγοράς. Και πολύ συχνά βέβαια η, τα μη ρυθμιζόμενα τμήματα της αγοράς και τα μη εποπτευόμενα προϊόντα ήταν οι τομεί όπου έγιναν και οι ενέργειες ε, που ήταν ενάντια στην εποπτεία και τις ε, ισχύουσες ρυθμίσει. Και αυτό θα πρέπει να το κατανοήσουμε γιατί είναι σημαντικό να δούμε τι μπορεί να κάνει η εποπτεία και οι κατάλληλε ρυθμίσει στο μέλλον. Οι αναλύσει διαφέρουν, αλλά όχι και σε πολύ μεγάλο βαθμό. Και προφανές είναι ότι η ρύθμιση και η εποπτεία σε αυτή τη μεγάλη αλυσίδα αιτίων και αποτελεσμάτων έπαιξαν μεγάλη μεγάλο ρόλο και είμαι ένας από, τους, αυτούς που πιστεύουν ότι η, μόνο στην αρχή της αλυσίδας ε, η εποπτεία Συγγνώμη, όχι, πολύ αργότερα στην αλυσίδα αιτίου αποτελέσματος παίζει ρόλο η υποπτία και η ρύθμιση και ίσως και για τον ίδιο ακριβώς λόγο θα έβλεπα και έναν διαφορετικό ρόλο όσον αφορά την τιτλοποίηση από ότι ο κύριος Σάνιο από παρουσίασε νωρίτερα ότι εγώ δεν, θα, δεν θεωρώ πως η τιτλοποίηση η ίδια ήταν κακή ούτε και εκείνος νομίζω αλλά υπάρχει ένας κίνδυνος να μπατάρει το πλοίο <laughs> αν υπερβάλλει κανείς την τιτλοποίηση. Και αντί να, ωστόσο υπάρχει τρόπος να περιοριστεί ο κίνδυνος αντί να επεκταθεί. Όμως αν δεν γίνει σωστή διαχείριση γίνεται πολύ γρήγορα κλιμάκωση και φτάνει σε επικίνδυνα σημεία. Ποιο ήταν το πρόβλημα της εποπτείας και αυτό αναφέρθηκε και νωρίτερα ότι είχε πολύ ισχυρό εστιασμό στην ε, μικροπρόβλεψη. Υπήρχε εποπτεία, υπήρχε εποπτεία και το χρηματοπιστωτικό σύστημα θεωρούσαμε πως ήταν ε, εποπτευόμενο και άρα ασφαλές. Πράγμα το οποίο ήταν μύθος, από ό,τι φάνηκε συνέχεια κίνδυνοι εντό των συστημάτων. Είναι προφανές ότι από αυτό καταλάβαμε πως δεν μπορούσαμε, το, μάλλον το ότι να αντιμετωπίσουμε το κίνδυνο δεν αφορούσε την αντιμετώπιση μεμονωμένου κινδύνου και μεμονωμένων ε, ιδρυμάτων. Δεν είναι βασική αριθμητική, δεν είναι βασικά μαθηματικά, είναι περίπλοκα μαθηματικά τα οποία δεν καταλαβαίνουμε καλά και τα οποία έχουν ε, πιθανές δυνατότητες εξάπλωσης πολύ ψηλότερων ε, βαθμών. Επίσης, έχουμε να κάνουμε και τους ενδογενείς κινδύνους που προκύπτουν από τη συλλογική συμπεριφορά. Και εδώ οι περισσότεροι υπόπτες μπορούν να φτιάξουν ωραία μοντέλα, αλλά κανένας ρυθμιστής δεν μπορεί να το εμποδίσει. Μπορούμε κάπως να δούμε τα υπερκυκλικ... τις υπερκυκλικές επιπτώσεις, την πτυτικότητα, αλλά δεν μπορεί να εξαφανιστεί ένας τέτοιος κίνδυνος, γιατί δεν αφορά την ατομική συμπεριφορά, αλλά την συλλογική συμπεριφορά. Και κάποτε θυμάμαι τότε ε, προείδρευα μιας επιτροπής του ΟΣΑ για τις χρηματοπιστωτικές αγοράς, ε, αγορές και οι συμμετέχοντες στην επιτροπή συνέχεραν ε, αλλήλους για το γεγονός ότι ο κίνδυνος είχε φύγει από το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Και εγώ τους ρώτησα, μα πού πήγε τότε. Ε, το είπα ότι αφορά τους επενδυτές. Εκείνοι δεν είναι μέρος. Εκείνοι δεν είναι μέρος του χρηματοπιστωτικού συστήματος και είπαν, όχι, όχι, είναι τα μεμονωμένα νοικοκυριά. Και αυτό ήταν τμήμα του μύθου που ίσχυε τότε. Σε κάποιο βαθμό υπήρχαν ιδιωτικά χαρτοφυλάκια με τον τρόπο, ας πούμε, όπως τα συνταξιδοτικά εκείνα τα μία και τα προϊόντα τους, αλλά εν πάση περιπτώσει γενικά οι άνθρωποι πίστευαν ε, ότι δεν υπήρχε κίνδυνος τότε. Ακόμα και οι χρηματομεσίδες το πίστευαν. Αυτό ήταν ένας ε, κίνδυνος ε, που υπήρχε εκ των προτέρων γιατί πριν από δύο-τρία χρόνια θεωρούσαμε, πιστεύαμε, πως η αλληλεπίδραση μεταξύ των διαφόρων κινδύνων εξομαλύνει τον κύκλο αλλά υπό ορισμένε συνθήκε συμβαίνει το εντελώ αντίθετο, όπω είδαμε. Και αυτό θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη καθώς προχωρούμε. Για τέτοια θέματα όπως η μόχλευση, η... ο κίνδυνος, ε, μάλλον η αναχέτηση του κινδύνου και πώς ε, λειτουργούν οι δυναμικές που είναι γεννή στο σύστημα. Η εποπτεία των χρηματοπιστωτικών ε, ε, ιδρυμάτων ε, έχει αποτύχει. Αυτό έχει γίνει πλέον ένα ρεφρέν που επανέρχεται. Πρέπει να αυξηθεί ο έλεγχος από πλευρά των, και των, των διοικήσεων, αλλά αυτό ισχύει όταν έχουμε ένα συγκεκριμένο επίπεδο κινδύνου. Ίσως λοιπόν θα πρέπει πιο στενά να δούμε γιατί υπήρχε τόσο πολύ κίνδυνος εντός του συστήματος. Και αυτό μας παραπέμπει στα αίτια που πιστεύω ότι βρίσκονται στην ε, πολιτική ε, εποπτείας και την υπερβολική ε, πρόβλεψη ρευστότητας με την οποία συνεχίζουμε να ζούμε εντό παρενθέσεως και όχι μόνο σε κάποια συγκεκριμένη χώρα, αλλά γενικά στην Ευρώπη και σε ολόκληρο τον κόσμο, αυτός ήταν ένας εγγενής ε, λόγος για τον οποίο υπήρχαν τόσο, υπήρχε τόσο πολύ μεγάλος κίνδυνος εντός του συστήματος. Διαχείριση καλύτερη του κινδύνου, αυτό ναι, αλλά δεν είναι η μόνη απαραίτητη προϋπόθεση για να αποτύχουμε άλλη αποτυχία και την επόμενη κρίση, αν ποτέ καταφέρουμε να βγούμε από τούτην εδώ. Τι συμβαίνει λοιπόν. Πολλά γίνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τα οποία βεβαίως θα γνωρίζετε το ζήτημα της εποπτείας που ακολούθησε την έκθεση Λαροζιέρ που, που πολύ σωστά απευθύνθηκε και στο μάκρο και στο μικρό επίπεδο. Ακούσαμε πάρα πολλές σήμερα για τις ε, κεφαλογικές απαιτήσει και αυτό βεβαίως ανάγεται στη ρευστότητα που υπάρχει μέσα στο σύστημα. Πρέπει να γίνει το κεφάλαιο πιο ακριβό κατά τρόπον ώστε να κατευθύνουμε την παροχή κεφαλαίου στην οικονομία, κατά το οποίο έχει μακροοικονομικές επιπτώσεις. Οι απαιτήσει ρευστότητα αναφέρθηκαν, οι λογιστικοί κανόνες επίσης ε, αναφέρονται το Διεθνές Ζωολογικό Πρότυπο το 39 είναι κάτι βεβαίως που κάθε φορά με απασχολεί. Στο εδώ ευρωπαϊκό επίπεδο αποδείχθηκε πως ήμασταν μάλλον πολύ προετοιμασμένοι αλλά για μια άλλη κρίση είχαμε ένα πολύ ωραίο μνημόνιο Είχαμε γύρω στις 142 υπογραφές νομίζω, ήμασταν προετοιμασμένοι για την αποτυχία ενός διοσυνοριακού ε, χρηματοπιστωτικού οργανισμού, αλλά όχι για μια τέτοια κρίση, οπότε νομίζω έχουμε ακόμα δρόμο. Ναι, κάπου κάπου στα σιρτάρια μας είναι, θα το ξεσκονίσουμε το μνημόνιο το 2011. Πρέπει να δούμε λοιπόν τι γίνεται με την, ε, τις δυνατότητες διαχείρισης συστημικής κρίσης και ζητήματα βεβαίως όπως ε, η εγγύηση των καταθέσεων, ε, τα της φερεγγιότητας κτλ. αναφέρθηκαν. Πράγματι λοιπόν ε, απέτυχε η εποπτεία και η ρύθμιση στο να προλάβει την κρίση και να στο να περιορίσει την κρίση. Ήμασταν πίσω από τα γεγονότα. Τώρα η απάντηση είναι αναστροφή της παγκοσμιοποίησης. Προφανώς όχι. Λιγότερη Ευρώπη, προφανώς όχι. Λιγότερη περιπλοκότητα, επίσης όχι αυτό το οποίο χρειάζεται να κάνουμε και επανέρχομαι εδώ πέρα στα αρχικά μου ερωτήματα, να επεκταθεί το εύρος της εποπτείας και της ρύθμισης. Πρέπει να γίνει μια πολύ προσεκτική ανάλυση του πώς θα αποφύγουμε το να παγιδευτούμε στην ρύθμιση στο μέλλον που θα παίξει σημαντικό ρόλο σε μικρές και σε μεγάλες χώρες και δεν έχουμε τώρα χρόνο να τα πούμε αλλά ήταν ένα σημαντικό γεγονός αυτό και να αναφέρω επίσης την συζήτηση του μήπως πάμε προς μια υπερβολική ρύθμιση. Εγώ θα έλεγα πως αυτό εξαρτάται από το πώς το βλέπει ο καθένας, από την σκοπιά αυτών που ε, υφίστανται τη ρύθμιση, μάλλον υπάρχει ο κίνδυνος, αλλά πρέπει να γίνει μια προσεκτική μακροοικονομική ανάλυση και εκεί πέρα νομίζω πως θα έλεγα πως υπάρχουν κίνδυνοι και προς τις δύο κατευθύνσεις και υπερβολικής και όχι αρκετής ρύθμισης και μια προσεκτική ανάλυση νομίζω θα μας δώσει το σύστημα το οποίο θα είναι ολιστικό και συνεκτικό. Την κατάλληλη στιγμή μου δείξατε το ρολόι και όλες γιατί τελείωσα. Ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστώ. Θα ήθελα τώρα να ζητήσω τους συναδέλφους, να ζητήσω τους συναδέλφους να κάνουν ερωτήσεις. Πρώτα απ' όλα δύο μέλη του ΕΛΚ λοιπόν. Ποιος θέλει τον λόγο. Okay. Uh, uh, Τζονάτα και... και Ότμαρ. Ευχαριστώ πολύ, λέει η κυρία Χούμπνα. Θέλω απλώς να πω ότι το γεγονός ότι εμείς δεν προβλέψαμε και δεν εμποδίσαμε την κρίση μας ε, φέρνει σε μια παγκόσμια πολύ καλή παρέα. Δεν ήμασταν οι μόνοι Αλλά το θέμα είναι πώς θα μπορέσουμε να αποσοβήσουμε την επανάληψη τέτοιων κρίσεων και τέτοιων σεισμών στο μέλλον. Το πρόβλημα το οποίο εγώ βλέπω ότι, το, ότι δεν ξέρουμε κατά πόσο αυτό το σύστημα το οποίο θέλουμε να δημιουργήσουμε θα είναι αποτελεσματικό και θα επιτύχει τους στόχους τους οποίους θέλουμε να επιζητήσουμε. Δεν ξέρουμε πότε θα το εγκρίνουμε καν, δεν ξέρουμε πώς θα εφαρμοστεί στην πράξη αυτό το νέο πλαίσιο. Αναρωτιέμαι αν τα κράτη-μέλη σκέφτονται για το αν χρειάζεται να συμπληρωθεί αυτό το σύστημα με εθνικές μεταρρυθμίσεις. Ούτε ξέρουμε καν πολλά σε σχέση με τις αλλαγές που λαμβάνουν χώρα αυτή τη στιγμή στα ίδια τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που θα προσαρμοστούν βέβαια στο νέο πλαίσιο αλλά κάνουν και εσωτερικές τομικές αλλαγές. Υπάρχουν επομένω πάρα πολλέ αβεβαιότητες <clears throat> και γι' αυτό αυτό το οποίο εγώ πιστεύω ότι είναι απαραίτητο είναι να εξασφαλίσουμε ότι όλες αυτές οι προσαρμογές θα συμμορφωθούν και θα καλυφθούν από τη λεγόμενη στρατηγική εξόδου που και αυτή είναι αρκετά βέβαια. Το ερώτημά μου είναι λοιπόν πολύ απλό. Πότε νομίζετε ότι θα έχουμε αρκετή σταθερότητα και αρκετή βεβαιότητα ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το νέο σύστημα. Πόσο καιρό θα χρειαστούμε να λάβετε υπόψη όλα αυτά τα στοιχεία. Ο κύριος Μαν. <coughs> Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Έχω ένα ερώτημα για τον κύριο Σάνιο. Αναφέρατε την ρύθμιση που είναι σαν ελβετικό τυρί, ότι υπάρχουν πάρα πολλά παραθυράκια, πως δεν ήταν αρκετά γνωστοί οι κίνδυνοι, δημιουργήθηκαν εταιρείε ειδικού σκοπού, δηλαδή μία σειρά μέτρων τα οποία δεν επέτρεπαν τη διαφάνεια. Επίσης, μιλήσατε για τους ε, αγοραστές, αλλά πώς ξέρετε πως αυτοί οι οποίοι αγοράζουν και που λένε γνωρίζουν και κυρίως αυτοί βέβαια που αγοράζουν γνωρίζουν περί τίνος ακριβώς πρόκειται σε αυτά τα προϊόντα. Επίσης είπατε εσείς για τη δική σας υπηρεσία πως δεν ήμασταν αρκετοί και πως δεν μας έπαιρναν σοβαρά. Τι είπα να πει δεν μας έπαιρναν σοβαρά. Μπορούμε να ξαναδούμε αυτή την κατάσταση γιατί εμείς θεωρούμε πως η δική σας υποπτική υπηρεσία μπορεί να κάνει αρκετά πράγματα. Το πρώτο ερώτημα προς τον κύριο Βίζερ και, το, στον κύριο Βίζερ και στο δεύτερο στον κύριο Σάνια. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Χρησιμοποίησα ένα παράδειγμα για το αν η αστυνομία και οι τροχονόμοι μπορούν να αποσοβήσουν όλα τα τροχαία ατυχήματα στο μέλλον. Και μπορούν να με εμποδίσουν να οδηγώ μες φορές πολύ γρήγορα. Αν έχουν ένα εξαιρετικά αποτελεσματικό σύστημα, πάρτε το παράδειγμα της Αυστρίας, εγώ θα είμαι πάντα νυφάλιος και θα οδηγώ πάντα και σωστά και δεν θα υπάρξει κίνδυνος ατυχήματος. Επομένως, είναι δυνατόν να φτιάξουν οι ρυθμιστές και οι επόπτες ένα σύστημα χωρίς εντάσεις και χωρίς δυσκολίες. Πίστευω όχι. Αλλά το ερώτημα είναι το νέο πλαίσιο το οποίο θέλουμε να δημιουργήσουμε, το νέο περιβάλλον το οποίο θεωρούμε ότι είναι πιο ασφαλές. Είναι εφικτό κάτι τέτοιο. Πιστεύω μετά από προσεκτική ανάλυση ότι μπορούμε να το κάνουμε αυτό <clears throat> γιατί αντιμετωπίζει Καταρχήν, το θέμα της σύνδεσης μεταξύ μακροοικονομικής και μικροοικονομικής εποπτείας. Και δεύτερον, δίνει περισσότερη Ευρώπη με την έννοια ότι όλοι μας γνωρίζουμε ότι με το να υπάρχουν ευρύτερες εξουσίες στους ρυθμιστές μπορούν να βελτιωθούν τα πράγματα. Είναι τέλειο αυτό το σύστημα, τίποτα δεν είναι τέλειο φυσικά. Και υπάρχουν και ορισμένα συνταγματικά πλαίσια τα οποία δεν μπορούμε να υπερβούμε προς το παρόν τουλάχιστον. Προϋπόθεση για να λειτουργήσει αυτό το σύστημα είναι ότι θα υπάρξει και παγκόσμια συνεργασία, ενισχυμένη παγκόσμια συνεργασία. Γιατί δεν σταματούν τα χρηματοοικονομικά προϊόντα και οι κίνδυνοι στα σύνορα της Ευρώπης. Μπορεί όμως να είναι θετικό το σύστημα αυτό για να αντιμετωπίσουμε τον κίνδυνο, να αναχαιτήσουμε τον κίνδυνο που έχω δει πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια να υπάρξει μια από ολοκλήρωση και επανεθνικοποίηση των χρηματοοικονομικών αγορών στην Ευρώπη. <clears throat> Αυτή τη στιγμή είναι πιο κατακαιρματισμένη η χρηματοοικονομική αγορά στην Ευρώπη από ό,τι ήταν πριν από δύο χρόνια. Πρέπει να γυρίσουμε λοιπόν το ρολόι πίσω. Θα πρέπει να αναδυθεί πάλι μια ευρωπαϊκή χρηματαγορά η οποία να είναι πιο ισχυρή από το παρελθόν αλλά με την πρέπουσα μακροοικονομική ε, εποπτεία για να αντιμετωπίσουμε την επόμενη κρίση η οποία αδειρήτω θα έρθει ο κύριος Σάνιο. Και εγώ συμφωνώ απόλυτα με αυτά που λέτε. Ότι η αρχή αυτή η Μπάφιν μπορεί να προχωρήσει θετικά και ότι θα έχει ένα, ένα θετικό χαρακτήρα στο μέλλον. Για το παρελθόν τώρα πρέπει να κάνουμε και μία διάκριση. Εγώ δεν είχα αρκετό χρόνο και δεν μπορούσα να αντιμετωπίσω όλα αυτά τα ουσιαστικά ερωτήματα. Αλλά μπορώ να πω κάτι το οποίο νομίζω ότι είναι κέριο. Εγώ περιέγραψα τους διεθνείς κανόνες ρύθμισης, οι οποίοι ήταν γραβιερόδεις. Αυτοί οι κανόνες είχαν εφαρμοστεί σε εθνική βάση μεμονωμένα. Ή για να το πω διαφορετικά, δεν υπήρχε κάποια αυστηρότητα στην εφαρμογή τους. Όλοι ξέραν ότι υπήρχαν παραθυράκια λοιπόν όταν τα πράγματα <clears throat> ξεκίνησαν και όλοι αποδεχόντουσαν τις ελλείψεις των συστημάτων. Η κρίση αυτή είχε ένα εκρηκτικό χαρακτήρα. Αμέσως μετά από τρεις δεκαετίες μεγάλης διαδικασίας απελευθέρωσης Και τελικά η διαδικασία αυτή απελευθέρωσης ε, οδήγησε στο, στην απροθυμία των πολιτικών να προχωρήσουν σε ένα νέο βήμα αριθμισή. Δεν λέω ότι φταίνε οι νομοθέτες, απλώς έτσι εξελίχθηκαν τα πράγματα. Ποιο ήταν το πραγματικό τώρα πρόβλημα πίσω από όλα αυτά και θέλω να το τονίσω τουλάχιστον να το αναφέρω. Το πραγματικό πρόβλημα πιστεύω για τις ρυθμιστικέ αρχές, για αυτού οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τη διαδικασία ρύθμισης, είναι ένα θέμα γνώσης. <clears throat> Σα είπα πω εξαπολύθηκε η κρίση. Ήταν σαν ήταν πυρηνικό πυροκροτητή. πυροκροτητής. Ήταν ο τομέας των subprime, των δευτεροκλασσάτων υποθηκών στι ΗΠΑ, τα λεγόμενα τοξικά αυτά ε, αξιόγραφα, τα οποία οδήγησαν σε απώλειες της τάξης των 3 εκατομμυρίων. Όλοι μας γνωρίζουμε ως ρυθμιστές ότι πρέπει να παρακολουθούμε πολύ προσεκτικά τη μακροοικονομική πλευρά για να δούμε πού υπάρχουν προβλήματα σε παγκόσμιο επίπεδο. Εγώ είμαι μέλος της FSP ή FSF αν θέλετε και σε όλες τις συναντήσεις μας συναντού, συζητούσαμε πάντα ποιες είναι οι τάσεις και τα δυνητικά προβλήματα σε παγκόσμιο επίπεδο στο χρηματοοικονομικό χώρο. Από πού μπορούν να προέλθουν οι κρίσεις και είχαμε πολλούς υποψηφίους. Αλλά κάτι το οποίο δεν είχαμε καταλάβει καθόλου ήταν ο δανεισμός με ενυπόθηκα δάνεια χαμηλής ποιότητας. Τα λεγόμενα subprime. <clears throat> το ίντερνετ έχει μια μνήμη. Μπορείτε να κοιτάξετε να δείτε τι ακριβώ έχει γίνει στο παρελθόν. Αν κάποιο είχε προειδοποιήσει αυτή την κρίση, κανεί δεν είχε προειδοποιήσει. Βλέπω την κόκκινη κάρτα και σας λέω εν κατακλείδη ότι δεν είμαστε καλά πληροφορημένοι για πράγματα τα οποία γίνονται κάτω από τη μύτη μας. Για να είμαι ειλικρινής δεν ξέρω πώς να λύσουμε αυτό το πρόβλημα πληροφόρησης. Περνάμε τώρα στους σοσιαλιστές με δύο ε, συναδέλφους. Κάποιος άλλος, ο Κοφεράτη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εμένα μου έχει προκαλέσει πολύ την περιέργεια ένα θέμα και γι' αυτό θα ήθελα να ξέρω ποια είναι η άποψη των συνομιλητών μας. Εμείς Μιλάμε με, με βάση μια προϋπόθεση ότι οι λύσεις δηλαδή είναι αντικείμενο εμβάθυνσης και συζήτησης και αφορούν βασικά ένα, ένα τρίγωνο που αποτελείται από τις ε, ρυθμιστικές υποπτικές αρχές, από την πολιτική που εδώ αντιπροσωπεύεται από μας και η άλλη γωνία είναι οι τράπεζες και τα χρηματοδοτικά ιδρύματα. Στην πράξη δεν μιλάμε για το τέταρτο υποκείμενο που είναι οι χρήστες, οι επιχειρήσεις, οι οικογένειες ή άτομα μεμονωμένα. Εφόσον λοιπόν μιλάμε για τις ρυθμίσεις, τις νέες, δεν θα έπρεπε από τώρα να σκεφτούμε ένα σύστημα σχέσεων με τον χρήστη που θα είναι παρόντες σε πολύ σε ολόκληρο τον κόσμο, ξεκινώντας από την Ευρώπη, ώστε να μην έχουμε μαζί τους απλά μία σχέση που θα φαίνεται μόνο όταν ε, ξεσπάει μία κρίση ή ένα δράμα. Εγώ σκέφτομαι τι έγινε με ορισμένες τράπεζες και επιχειρήσεις στη χώρα μου. Η παρέμβαση στη συνέχεια, μάλλον κατόπιν εορτής ε, με τον καταδίκη ή την δίωξη, ήταν πολύ αργά πια. Θα ήθελα τώρα να ζητήσω την, την κυρία Βούντερερ να απαντήσει και μετά ίσως να συμπληρώσουν και... να συμπληρώσει αν έχει να πει κάτι. Για να απαντήσω στο ερώτημα αυτό νομίζω πως πράγματι επικεντρωνόμαστε πάρα πολύ στην στο κομμάτι που αναφέρατε και οι καταναλωτές μένουν απ' έξω. Το πρόβλημα είναι πως ε, έχουμε μεγάλη ε, ποικιλία στην πλευρά των καταναλωτών. Υπάρχουν ίσως κάποιες οργανώσεις καταναλωτών, αλλά δεν υπάρχει έτσι ένα οργανωμένο κομμάτι αυτού του τετραγώνου, όχι τριγώνου για να μπορούν έτσι αυτά τα συμφέροντα να ομαδοποιηθούν και να συνοψιστούν. Πρέπει να το σκεφτούμε αυτό, να το εξετάσουμε. Αυτό το οποίο κάνουν οι οργανώσεις των καταναλωτών είναι σωστό, αλλά η άποψή μου είναι πως τελικά η προστασία των καταναλωτών πρέπει να αποτελέσει συστατικό κομμάτι της ε, εποπτείας. Δεν πρέπει να φτάσουμε σε μια κατάσταση στην οποία θα δημιουργήσουμε έναν τέταρτο ας πούμε πυλώνα αξιολόγησης ε, ε, ή ανάπτυξης μοντέλων και κριτηρίων αξιολόγησης αλλά νομίζω πως η προστασία του καταναλωτή πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των εποπτικών αρχών και θα πρέπει να κινητοποιηθούν σε αυτόν τον τομέα. Κύριε Σάνιο, θέλετε να πείτε κάτι. Ναι, ένα πολύ σημαντικό κομμάτι, η προστασία των καταναλωτών. Είναι κάπως ηρωνικό εδώ πέρα αυτό το οποίο συμβαίνει. Αυτό το οποίο περιέγραψα εγώ, έτσι, για να είμαι λίγο κοινικός, είναι πως κάποιοι από τους θεσμικούς ε, παίκτες, ε, αγοραστές και πολιτές, ήθελαν ίσως προστασία καταναλωτών γιατί δεν αντιλαμβάνονταν το προϊόν, ενώ αυτό συνήθως συμβαίνει με τους πελάτες της Λιανικής που πρέπει να προστατευτούν από τα επικίνδυνα προϊόντα, αλλά κοντολογής δεν υπάρχει ε, αρκετή προστασία για τους πελάτες Λιανικής, αλλά σε όλη αυτή την ε, κρίση δεν έχει βλαφτεί κάποιος καταναλωτής Λιανικής, αλλά τα θεσμικά όργανα την πλήρωσαν επειδή δεν αντιλαμβάνονταν τα προϊόντα, μανθισμικοί παίκτες, γιατί δεν αντιλαμβάνονταν ε, τα προϊόντα. Τώρα δεν θέλω να πω και εγώ τα όσα λέει ο Warren Buffett. Τα προϊόντα αυτά είναι υψηλού κινδύνου, υψηλού συστημικού κινδύνου και βεβαίω όσο πιο επικίνδυνα τόσο λιγότεροι τα αντιλαμβάνονται, παρόλα αυτά τους επιτρέπεται να τα αγοράσουν, να τα χρησιμοποιήσουν. Και είναι δύσκολο άρα το ερώτημα. Αν θέμε δηλαδή να περιορίσουμε την ελευθερία των συμμετεχόντων στην αγορά. Κύριος Μπούλμαν, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρο. Το κοινοβούλιο μας έχει το στόχο να δημιουργήσει την απαραίτητη νομοθεσία για ένα νέο σύστημα εποπτείας και βέβαια πρέπει να διαβουλευτεί και να αντιμετωπίσει το σύστημα για τη σωστή ισορροπία, πόση πρέπει να είναι η αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πόση αρμοδιότητα πρέπει να παραμείνει στα πλαίσια των κρατών μελών, τι είναι απαραίτητο για να μπορέσουν να λειτουργήσουν τα διάφορα συστήματα εποπτείας αρμονικά μεταξύ τους. Εγώ θα ήθελα να ξέρω αν εσείς θεωρείτε αν βρίσκεται ότι η πρόταση της Κομισιόν έχει επιτύχει την κατάλληλη ισορροπία. Βλέπετε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέλει μια πιο δυναμική αντιμετώπιση. Όλες οι πολιτικές ομάδες θέλουν μια πιο δυναμική άποψη. Εσείς από την οπτική γωνία του, του Συμβουλίου Συστημικών Κινδύνων και των Εποπτικών Συμβουλίων. Μήπως θεωρείτε ότι θα έπρεπε να υπάρχουν περισσότερες αρμοδιότητες σε καταστάσεις κινδύνου, οι οποίες θα μπορούσαν να μας εξασφαλίσουν καλύτερα. Το ερώτημα στον Τόμας Βίζε. Μα έχουμε και το δεύτερο πάνελ, το οποίο θα ξεκινήσει αμέσως τώρα και που ασχολείται ακριβώς με το θέμα αυτό. Ποιο υπόδειγμα πρέπει να έχουμε για το μέλλον. Μα έχουμε τόσο ενδιαφέροντες ε, ομιλητές που είναι χρήσιμο να ακούσουμε και την άποψή τους. Ο κύριος Βίζεν, ευχαριστώ πολύ. Είναι προφανές ότι ως εκπρόσωπος της Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επιτροπής έχω και μια συγκινησιακή και θεσμική προσήλωση στα κείμενα τα οποία εμείς έχουμε ε, δώσει στο Συμβούλιο και που έχουν εγκριθεί από το Συμβούλιο ΕΚΟΦΗΝ. Επομένως είμαι κάπως μεροληπτικός από συγκινησιακή και θεσμική άποψη. Το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο δεν νομίζω ότι διαφέρουν σε ό,τι αφορά την πεποίθηση ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρξει μια ισχυρή και στεναρή μακροεποπτική ε, πτυχή στα μέτρα αυτά. Και ξέρω ότι συζητήθηκαν όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία αναφέρεται και στο Συμβούλιο. Ότι δηλαδή πρέπει να συνοδεύεται όλο, όλη αυτή η προσέγγιση μακρο εποπτική σε μία, με μία ισχυρή μικροεποπτική διαδικασία. Εδώ δεν υπάρχει καμία διαφορά μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου. Τώρα προφανώς μέσα στο Συμβουλίο μεταξύ των 27 κρατών μελών υπήρχαν 28 διαφορετικές απόψεις για το πόσο μακριά θα μπορούσε κανείς να προχωρήσει για να έχει περισσότερη Ευρώπη και όπως φαντάζεστε ήταν μια πολύ προσεκτική συμβιβαστική λύση στην οποία κατέληξε το Συμβούλιο. Αυτό το οποίο εγώ θα ήθελα να δω να γίνει αποδεκτό θα ήταν κάτι περισσότερο, αλλά αυτό στο οποίο καταλήξαμε πιστεύω ότι ήταν επαρκές. Στο στάδιο που είχαμε φτάσει θα ήταν καλύτερα να έχουμε ε, περισσότερη Ευρώπη στο τωρινό επίπεδο και όχι μια Ευρώπη που βρίσκεται πολύ μακριά στον ορίζοντα. Γι' αυτό τονίζω ότι είναι μια πολύ καλή συμβαστική λύση, αλλά καταλαβαίνω και την άποψη του Κοινοβουλίου ο κύριος Σάνιο. Δεν θέλω να υπάρξει παρεξήγηση. Εγώ δεν είμαι εδώ εκπρόσωπος γερμανικής κυβέρνησης, κάθε άλλο. Αλλά μπορώ να κάνω κάποια σύντομα σχόλια γιατί νομίζω ότι είναι σημαντικό το θέμα της μακροοικονομικής εποπτείας. Όπως είπα προηγουμένως, πολλές φορές η κοινή γνώμη θεωρεί ότι οι μακροοικονομικές πτυχές ήταν άγνωστες μέχρι τώρα αλλά και το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο βρίσκονται στη σωστή πορεία όταν υπογραμμίζετε τη σημασία της μακροοικονομικής εποπτείας και όταν προσπαθείτε να δημιουργήσετε ένα θεσμικό πλαίσιο που να δίνει προεξάρχοντα ρόλο στην μακροοικονομική εποπτεία. Για μένα αυτό είναι το πιο δύσκολο το οποίο θα πρέπει, το πιο δύσκολο εγχείρημα για το μέλλον. Αν δούμε το παρελθόν, <clears throat> αν φανταστώ να υπήρχε ήδη το Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου, θα είχε καταλάβει ότι επίκειται αυτή η κρίση για τα subprime ε, ενυπόθηκα δάκτυα. Θα ήξερε πώς να αντιμετωπίσει εγκαίρως αυτό το πρόβλημα όταν ανα, Και μιλάμε για παγκόσμιες τάσεις. Θα μπορούσε παραγωγικά η κυβέρνηση των ΗΠΑ να δεχτεί την Συμβουλή τη Ευρωπαϊκής Ένωση και πώς θα προχωρούσε κάτι τέτοιο. Αυτό το οποίο με ενδιαφέρει είναι να δούμε με ποιο τρόπο θα μπορέσουν να συνεργαστούν όλες οι πτυχέ και πώς θα είναι επιτυχής σε αυτή την κατεύθυνση. Υπάρχει μια αγγλική παροιμία ότι ο χρόνος δοκιμάζει δοκιμάζει πάντα την αλήθεια. Εγώ θα προτιμούσα λοιπόν να μην γίνονται όλα με δοκιμές και μόνο. Κυρία Γένσερ, τελευταίο ερώτημα. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ για τις ε, παρεμβάσεις σας. Ε, μιλήσατε όλοι για την ε, ελβετική γραβιέρα με τη, που είναι διάτρετη και επίσης για το ότι η αστυνομία δεν μπορεί να εμποδίσει όλα τα τροχαία ατυχήματα. Και μάλιστα να σας πω ότι όταν ήρθα μέχρι εδώ ε, έφυγα με πολύ χιονισμένη Δανία, πολλοί οδηγούσαν πολύ σιγά, ωστόσο υπήρχαν και διάφοροι στην άκρη του δρόμου που είχαν τρακάρει. Πτέ παράδειγμα ότι πρέπει να είμαστε ακόμα πιο προσεκτικοί. Εσείς ε, τι λέτε, οι, οι, οι ρυθμιστές όντως δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα, όλα ήταν τόσο χαλαρά. Ε, προηγουμένως είμαστε όπως είπε και ο κύριος Νουαγέ, ο κροθυγός, υπερ ε, αντιδρούμε. Υπάρχει στον τραπεζικό τομέα συνείδηση για τη σοβαρότητα των όσων συνέβησαν. Αρχίζουν να βλέπουν ε, την ανάγκη για πιο συνετή και δράση. Κύριε Ζάνιο, θα ήθελα να σας το πω στα γερμανικά αυτό που θέλω να πω. Έχουμε ένα θέμα εδώ πέρα σήμερα. Δηλαδή μετά την αποτυχία της εποπτείας και της ρύθμισης Μιλήσατε μόνο για τη ρύθμιση, όχι για την εποπτεία, για την δική σας ευθύνη και τα δικαιώματά σας τα οποία δεν εξασκήσατε. Μπορούσατε να πάει στιγμή να λάβετε μέρος. Ξεκαθαρίστηκε αυτό στην Εξεταστική Επιτροπή της Γερμανικής Βουλής, πως δεν προειδοποιήσατε αρκετά. Χτες, επίσης, δεν είπατε πως... Ο επίσκοπος ε, παρετήθηκε γιατί οδηγούσε μεθυσμένη και εσείς ε, που είσαστε υπεύθυνος για την απώλεια δισεκατομμυρίων πότε θα αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κοιτάξτε, είναι επιπροσωπικού η ερώτηση, κύριε συνάδελφε. Ε, δεν ξέρω, μήπως θα μπορούσατε να την αναδιατυπώσετε ε, κάπως πιο θεσμική. Και, κύριε Σάνιο, μετά απαντήστε. Κοιτάξτε, όταν με προσκαλούν ε, ως ε, εμπειρογνώμονα συνήθως δεν μου ζητάνε την παρέτησή μου. Ε, με ενοχλεί λιγάκι, ομολογώ. Έρχομαι ως, ως εμπειρογνώμονας και όχι για να μπω εγώ σε μια πολιτική διαμάχη. και ε, δεν, δεν, θα σας απαντήσω, δεν είναι και συμπεριφορά αυτή. Ε, ιδιωτικά, ε, αν θέλετε... Οι δυο μας βεβαίως να σας απαντήσω τώρα για την άλλη ερώτηση, δεν ξέρω αν θέλει να απαντήσει ο κ. Βίζερ. Πού βρισκόμαστε τώρα. Συμφωνώ με την άποψη του διοικητού του κυρίου Ναγέ. δεν ήταν ε, έτσι πολύ έντονη η διατύπωσή του. Πώς πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί να μην κάνουμε πάρα πολλά ταυτόχρονα. Νομίζω αυτό είπε και εκείνος. Ποιο θα είναι το αποτέλεσμα τους επόμενους μήνες. Θα έχουμε πάρα πολλά πράγματα για τις τράπεζες, αν και δεν ξέρουμε τις ε, ποσότητες, οπωσδήποτε θα ανεβούν οι κεφαλαϊκές απαιτήσεις Ταυτόχρονα από πλευράς ε, Αμερικανών ε, θα πούμε οπωσδήποτε. Βλέπετε πως έχουν εκεί νέες ιδέες, πως το κόστος το ανακτούν, παίρνουν τα λεφτά τους πίσω. Μετά υπάρχει άλλη ιδέα δημιουργίας ταμείων, υπέρ ταμείων που θα πρέπει να γεμίσουν με πολλά χρήματα βέβαια και μπορεί να έχουμε έτσι ένα σωρευτικό αποτέλεσμα που ίσως θα προκαλέσει το να μην δανείζουν πλέον οι τράπεζες. Και κάποιος το ανέφερε επίσης, ε, συζητάνε και στρατηγικές εξόδου οι κεντρικές τράπεζες, δηλαδή να αποσύρουν το φτηνό χρήμα από την αγορά, το οποίο υποστηρίζει τη ρευστότητα της αγοράς. Ε, για να γίνουν όλα αυτά τους επόμενους ε, μήνες θα είναι κάτι το πολύ δύσκολο και εύχομαι σε όλους τους συμμετέχοντες, ειδικά στις κεντρικές τράπεζες που έχουν τη βασική ευθύνη, ε, καλή επιτυχία γιατί κανένας ε, άλλος στο παρελθόν δεν είχε τόσο δύσκολο καθήκον όσον αφορά τώρα την αλλαγή των ε, ρυθμιστικών δομών. Νομίζω πως σε ερχόμενους μήνες ε, θα δείτε πως ε, τα πιο θεμελιώδη ερωτήματα θα απαντηθούν η απάντηση μπορεί να είναι οπωσδήποτε αρνητική. Τι εννοώ αρνητική? Ότι δεν θα έχουμε παγκόσμιους κανόνες. Για εμένα αυτό είναι το σημαντικότερο. Εάν δεν μπορέσουμε να ορίσουμε παγκόσμιους κανόνες, εάν επανεθνικοποιήσουμε τις παγκόσμιες αγορές, κάτι το οποίο είναι αντιφατικό από μόνο του, τότε νομίζω πως θα καταλήξουμε σε μια κατάσταση επικίνδυνη γιατί μετά όλα τα ζητήματα που οφείλονται στο που είναι εγκατεστημένη μια εταιρεία όπως τα ζητήματα offshore κτλ θα ανακύψουν ξανά και θα δούμε μετά πως η ρύθμιση της αγοράς συνεχώς θα μειώνεται, θα έχουμε ένα ανταγωνισμό προς τα κάτω. Επίσης η ρύθμιση είναι οι κανόνες. Αυτό που έχει σημασία είναι πώς εφαρμόζονται από τις υποπτικές αρχές και πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στο να α, ανεβούν, αν θέλετε, οι προδιαγραφές και τις υποπτίας και όχι μόνο οι κανόνες. Ευχαριστώ. Περνάμε στο δεύτερο πάνελ. Ευχαριστώ τους ε, πρώτου πανελίστε που είναι εδώ ακόμα για τη συμμετοχή τους και τις απαντήσεις τους και θα ακούσουμε τώρα τους ε, τρει συμμετέχοντες του δεύτερου μέρους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 pronounce your name? Perso? That's, that will be a European pronunciation. And how do you pronounce it? I say Persaud. Persaud, okay. Oh, no, no, it's okay. I'm just Persaud. Depends on the French people. Okay, yeah, yeah. So, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir kommen zum... Λοιπόν, συνάδελφοι, περνάμε στο δεύτερο τμήμα του απογεύματος. Ποιο είναι το μελλοντικό μοντέλο της Ευρώπης, το ερώτημα που ανέφερε ο κ. Μπούλμαν. Έχουμε τρία μέλη εδώ πέρα. Ξεκινάμε με τον κύριο Αβινάς Περσό στο κέντρο, καθηγητή επίτιμο του Gresham College και η γνωστή Ίκε Φαντενμπούρχ που ήταν μέχρι τις προηγούμενες εκλογές συνάδελφος εδώ πέρα και είχε ε, συντάξει μια έκθεση που ασχολούνταν με αυτά τα ζητήματα και ο Ράσου και της Σβέντμπανκ, ε, ο επικεφαλής ε, οικονομολόγος. Ε, θα σας δώσω λοιπόν τον λόγο και παρακαλώ να σεβαστείτε το χρόνο. Μικρόφωνο παρακαλώ. Thank you very much, ladies and... Ευχαριστώ πολύ κυρίες και κύριοι. Μεγάλη τιμή είναι για μένα να είμαι εδώ παρόν ενώπιον σας. Θέλω να ευχαριστήσω την Επιτροπή σας και να σας συγχαρώ για το σημαντικό και πάρα πολύ υπεύθυνο ρόλο που παίζετε σε αυτή την τόσο σημαντική συζήτηση για τα οικονομικά θέματα. Επομιζόσαστε λοιπόν μια μεγάλη ευθύνη για να εξασφαλίσετε για να εξασφαλίσετε ότι τεράστιες οικονομικές, κοινωνικές, ανθρώπινες συνέπειες αυτής της κρίσης δεν θα επαναληφθούν στο άμεσο μέλλον. Όταν σκεφτόμαστε για το μελλοντικό υπόδειγμα που θα πρέπει να έχουμε, το μοντέλο, τη λύση, την ρυθμιστική λύση που θα εμποδίσει μελλοντικέ κρίσεις και συγκεκριμένα <clears throat> το ευρωπαϊκό αυτορυθμιστικό μοντέλο, θα πρέπει καταρχήν να εντοπίσουμε και να περιγράψουμε σωστά το πρόβλημα το οποίο θέλουμε να λύσουμε. Και αυτό θέλω να το πω γενικά. Καταρχήν, γιατί πάντα υπάρχουν πολύ συγκεκριμένα προβλήματα σε κάθε κρίση. Αλλά εμείς θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε πρώτα το γενικό πρόβλημα. Και πρέπει να το πράξουμε αυτό. Γιατί η κατάσταση πάντα στις αγορές είναι δυναμικές. Είναι δυναμική. Όταν έχουμε μόλις κερδίσει τον τελευταίο πόλεμο, δεν είμαστε πάντα έτοιμοι να ξεκινήσουμε τον επόμενο. Το δυναμικό στοιχείο στο χρηματοοικονομικό σύστημα είναι ότι σε κάθε κίνηση των ρυθμιστών απαντά και ανταποκρίνεται το χρηματοοικονομικό σύστημα, χρηματοπιστωτικό σύστημα. Πρέπει λοιπόν να εξασφαλίσουμε ότι η λύση θα είναι εφικτή και πρακτική. Εγώ πιστεύω μπορούμε να φτάσουμε σε μια πρακτική λύση σήμερα που θα έχει σημαντικό ε, αντίκτυπο και θα μπορέσει να μετριάσει και να αντιμετωπίσει τις μελλοντικές χρηματοπιστωτικές κρίσεις. Μιλάω για τη λεγόμενη μακροοικονομική εποπτεία και ρύθμιση ιδίως ό,τι αφορά τις απαιτήσει κεφαλαίου, τη μακροπολιτική μάλλον εποπτεία και σε ό,τι αφορά επίσης τη δομή του χρηματοπιστωτικού μας συστήματος. Από πολιτική άποψη είναι πολλές φορές δελεαστικό να περιγράψει κανείς αυτά τα οποία ήταν η αιτία του προβλήματος ως η πονηρή και ύπουλοι καλοπληρωμένοι τραπεζίτες οι οποίοι βρισκόντουσαν στα όρια του σωστού και του, της ρύθμισης και οι οποίοι πουλούσαν ενσυνείδητα τοξικά αξιόγραφα στους πολίτες. Πάντα υπάρχει ένα στοιχείο και αυτής της πτυχής σε κάθε κρίση και αυτό πρέπει να το αποσοβήσει η ρύθμιση η οποία πρέπει να εφαρμοστεί. Αλλά πιστεύω ότι αυτό από μόνο του δεν φτάνει. Αυτή είναι μια πολύ ανεπαρκής χαρακτήριση τη κατάσταση Είναι πάρα πολύ βολική σε πολιτικό επίπεδο, αλλά σε τελική ανάλυση αυτή δεν είναι η πρώτη και δυστυχώ ούτε η τελευταία χρηματοπιστωτική κρίση και κατάρρευση. Οι καταρρεύσει οδηγούν πάντα την ταχεία ανάπτυξη. Γι' αυτό η ρυθμιστική μας απάντηση θα πρέπει να αντιμετωπίσει και την ταχεία ανάπτυξη, την ταχεία χρηματοοικονομική επέκταση οποιαδήποτε πρόταση που θα θέσετε η οποία δεν αντιμετωπίζει το φαινόμενο των φουσκών της ταχείας αυτής χρηματοπιστωτικής επέκτασης δεν θα είναι αποτελεσματική. Τι οδηγεί λοιπόν σε αυτή την ταχεία επέκταση. Είναι κυρίως οι τραπεζίτες αλλά είναι και όλη η κοινωνία η οποία πιστεύει ότι κάτι είναι που να έχει κάνει τον κόσμο πιο ασφαλή. Και επειδή ο κόσμος έχει γίνει πιο ασφαλής μπορούν να αναλάβουν περισσότερους κινδύνους από ό,τι στο παρελθόν. <clears throat> Πολλές φορές υπάρχει μια τεχνολογική αλλαγή. Η σιδηρόδρομοι, η χρήση του ηλεκτρισμού, η χρήση του ίντερνετ. Θεωρούν πολλές φορές ότι οι πολίτες έχουν, ότι ο κόσμος έχει αλλάξει, ότι έχει γίνει κάτι το ουσιαστικό και επομένως έχουν εξαλειφθεί κίνδυνοι η παγκοσμιοποίηση έχει αλλάξει τα πράγματα. Και αυτό το οποίο είναι εκπληκτικό για αυτή την ιδιαίτερη κατάσταση που αντιμετωπίσουμε είναι ότι η καινοτομία δεν αφορούσε το λογισμικό ή το υλικό. Ήταν καθαρά στον τομέα της χρηματοοικονομικής καινοτομίας. Κάποιοι πίστεψαν ότι η χρηματοοικονομική καινοτομία, χρηματοοικονομικης καινοτομια καποιοι μάλλον καινοτομία, έκανε τον κόσμο πιο ασφαλή. Δεν είναι μονάχα ότι οι τραπεζίτες βγάλαν όπλα μαζικής καταστροφής από τις εσωτερικές τους τσέπες και τα ρίξανε σε ένα απορριμμένο κοινό καταναλωτών και μετά το βάλαν στα πόδια. Όχι. Απλώς οι τραπεζίτες έβγαλαν όπλα μαζικής καταστροφής, τα ρίξανε σε ένα κόσμο γεμάτο από απορριμμένους καταναλωτές και μετά έτρεξαν μαζί με τους καταναλωτές. Γιατί θέλανε κι άλλα οι καταναλωτές. Τα βάλαν στις τσέπες τους και ζητούσαν περισσότερο. Οι τράπεζες που απέτυχαν, που κατέρευσαν, ήταν τίγκα με τέτοια προϊόντα. Αυτό δείχνει κάτι το οποίο είναι σημαντικό. Οι κρίσει οφείλονται σε αυτούς που πιστεύουν ότι οι κίνδυνοι είναι υποδέστεροι από αυτούς που είναι στην πραγματικότητα. Δεν κάνουν κάτι ηθελημένα, ρισκαρισμένο και προσπαθούν να ξεφύγουν. Υπάρχει και αυτό. Το βασικό όμως σε μια πάντα ταχεία επέκταση σε μια φούσκα είναι ότι αυτά τα χρηματοοικονομικά προϊόντα είναι ασφαλή και γι' αυτό μπορώ να αυξήσω την έκθεση του, της τραπεζάς μου σε τέτοια προϊόντα. Και δεν ήταν μονάχα οι τραπεζίτες και οι ρυθμιστές έπεσαν στη λούμπα. Θεώρησαν ότι ο κόσμος ήταν πιο ασφαλής. Θεωρούσαν ότι με την επέκταση της τιτλοποίησης και των ανταλλαγών συμβολέων αφέτησης πληρωμών ότι όλα αυτά θα κάνουν το σύστημα πιο ασφαλές. Σε κάθε έκθεση χρηματοοικονομικής και χρηματοπιστωτικής ε, σταθερότητας λέγανε το ίδιο πράγμα. Ο κίνδυνος διαχέεται μακρά, μακράν του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Και θεωρούσαν ότι οι υποθήκες subprimes δημιουργούσαν μεγαλύτερη περιεκτικότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος, που έφτανε πια άτομα τα οποία στο παρελθόν δεν είχαν τη δυνατότητα να έχουν τραπεζικούς λογαριασμούς και υποθήκες. Ήταν ένα στοιχείο καινοτομία που επέκτηνε την κατανομή του κινδύνου σε όλους. Αυτό ήταν τουλάχιστον η θεωρία. Και εδώ και οι τραπεζίτες και οι ρυθμιστές πίστεψαν σε αυτή την ιστορία. Αυτό λοιπόν πρέπει να το αντιμετωπίσουμε σε ένα μελλοντικό μοντέλο ρύθμισης. Το μέλλον της ρύθμισης θα πρέπει να αντιμετωπίσει την αποτυχία της αγοράς να αξιολογήσει σωστά τους κινδύνους. Οποιοδήποτε τέτοιο σύστημα λοιπόν ρύθμισης θα πρέπει να αντιμετωπίσει την ανικανότητα και την αποτυχία της ε, αγοράς να εκτιμά τους κινδύνους. Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα με τη Βασιλεία 2. Γιατί όπως ξέρετε η Βασιλεία 2 έδωσε έμφαση στην αξιολόγηση που κάνει η αγορά για τους κινδύνους στους πυλώνες 1, 2 και 3. Και γι' αυτό η κρίση αυτή ήταν πιο βαθιά από την προηγούμενη. Πρέπει να κάνουμε λοιπόν τροποποίηση στη Βασιλεία 2 σε δύο συγκεκριμένους τομείς. Για να το πω με άλλα λόγια. Η Βασιλεία 2 ξεκίνησε από την ιδέα ότι μπορεί να υπάρχει μια στατιστική εκτίμηση του κινδύνου, ότι είναι ποσοτικοποιήσιμο ο κίνδυνο. Μπορούμε να το καταμετρήσουμε, μπορούμε να δούμε συσχετισμού, μπορούμε να δούμε την, ε, την πτυτικότητα των κινδύνων, να έχουμε στατιστικές μετρήσεις του κινδύνου. Αν θέλουμε λοιπόν να προστατευτούμε έναντι του κινδύνου της αγοράς, ότι δεν μπορεί να εκτιμήσει σωστά τον κίνδυνο, θα πρέπει να έχουμε μια πιο δομημένη αντιμετώπιση του κινδύνου, ώστε να μην φερόμαστε και να από τις στατιστικές. Θα πρέπει να έχουμε μια δομική αντιμετώπιση του κίνδυνου. Πώς. Καταρχήν, με το να καταλάβουμε ότι το κύριο στοιχείο αποτυχίας των στατιστικών αξιολόγηση κινδύνου οφείλεται στον οικονομικό κύκλο. Όταν τα πράγματα πηγαίνουν καλά, ο κόσμος στατιστικά είναι πιο ασφαλής. Είναι λιγότερες οι αποτυχίες πιστοτικών ιδρυμάτων και είναι λιγότερες από την προηγούμενη φορά που είχαμε μια ταχεία επέκταση. Αυτό οδηγεί σε μεγαλύτερη μόχλευση. Πρέπει να βάλουμε λοιπόν τον οικονομικό κύκλο πίσω μέσα στην οικονομική και χρηματοπιστωτική ρύθμιση. Και η Επιτροπή της Βασιλείας και το Συμβούλιο ε, Συστημικών Κινδύνων θέλει να, να ενσωματώσει αντικυκλικά μέτρα μέσα στη ρύθμιση. Θα έπρεπε τα ίδια κεφάλαια να αυξάνονται με την οικονομική επέκταση και όχι απλώς να μειώνεται. Ένα δεύτερο πρόβλημα είναι η δομή του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Δεν μπορούμε να πιστεύουμε τις στατιστικές για τους κινδύνους και πρέπει οι ρυθμιστές να ξεκινούν από αυτό. Θα πρέπει οι ρυθμιστές να χαροτήσουν τους τράπεζες. Κάντε περισσότερες στατιστικές για τους κινδύνους σας. Άμα δεν πιστεύω τις στατιστικές δεν μπορώ να διαχειριστώ τους κινδύνους. Όχι. Σημαίνει ότι πρέπει να κοιτάζω τις διαρθωτικές πτυχές του κινδύνου. Αυξάνουν τα ενεργητικά ή το παθητικό μιας τράπεζας πολύ ταχύτερα. Υπάρχει μεγαλύτερη συγκέντρωση κινδύνων από ό,τι στο παρελθόν. Και πιο σημαντικό από όλα. Βλέπουμε να υπάρχει αναντιστοιχία μεταξύ της ικανότητας ενός πιστοτικού ιδρύματος να απορροφήσει ενδεχόμενες ζημίες και τις, ε, ε τα ανοίγματα στα οποία προχωράει. Νομίζω ότι ένας ουσιαστικός τρόπος να το αντιμετωπίσουμε αυτό είναι να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση στη ρευστότητα από ό,τι στο παρελθόν. Σκέφτονται για τα μαξιλάρια ρευστότητα οι ρυθμιστέ. Αυτό δεν φτάνει αρκετά μακριά. Πρέπει να έχουμε ένα, <clears throat> μια απέτηση για περισσότερα κεφάλαια όταν υπάρχει αναντιστοιχεία ρευστότητα μεταξύ των στοιχείων του, του ενεργητικού. Αυτό θα δώσει λοιπόν μια θετική μορφή κατακαιρματισμού του συστήματος. Αυτοί που έχουν μεγάλη έλλειψη ρευστότητας δεν θα παίρνουν κινδύνους ρευστότητας. Τα πιστοτικά ιδρύματα τα οποία έχουν στοιχεία ενεργητικού σε μακροπρόθεσμη τοποθέτηση μπορούν να πάρουν περισσότερους κινδύνους ρευστότητας. Λοιπόν, δεν μπορώ, δεν θέλω να σας ε, χρησιμοποιήσω να πάρω και περισσότερο από το χρόνο σας. Θέλω να έρθω τώρα στην μακροπροληπτική εποπτεία. Αυτό είναι ένα πρόβλημα για όλους μας και εγώ είμαι Ευρωπαίος που πιστεύω ιδιαίτερα στο ευρωπαϊκό σύστημα και στο ευρώ. Η μακροπροληπτική εποπτεία φοβάμαι ότι γίνεται καλύτερα σε εθνικό επίπεδο. Οι οικονομικοί κύκλοι λειτουργούν σε εθνικό επίπεδο. Η Ιρλανδία, η Ισπανία, η Πορτογαλία και η Ελλάδα έχουν προβλήματα γιατί η διαδικασία οικονομική επέκταση δεν ήταν παράλληλη με αυτή άλλων χωρών. Θα πρέπει να σκεφτούμε λοιπόν για ένα δίκτυο εθνική μακροπροληπτική εποπτεία με την εποπτεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία δίνει και μια επαρκή απόσταση. Γιατί εγώ φοβάμαι ότι δεν θέλουμε ότι να έχουμε μια ουσιαστικά κατάληψη της ρυθμιστικής εξουσίας μόνο από τα εθνικά κράτη. Η ΙΚΕ. Thank you. Uh, ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ που με προσκαλέσατε να ξανάρθω στις ε, Βρυξέλλες. Έχω κάνει βεβαίω μια παρουσίαση με PowerPoint. Θυμάμαι πως όταν ήρθα να παρουσιάσω την τελευταία μου έκθεση με τον κύριο Νταϊάνου στην Επιτροπή δεν ε, το θεωρήσαμε σωστό μια βουλευτής να, να κάνει παρουσίαση με PowerPoint, οπότε τώρα δράτω με τις ευκαιρίες να το κάνω αλλά είναι αρκετά μακροσκελής αυτή η παρουσίαση γιατί ήθελα να σας υπενθυμίσω κάποια πράγματα από εκθέσεις που έχουμε κάνει εδώ για να σας δείξω τι είχε κάνει το Ευρωπαϊκό ε, Κοινοβούλιο στο παρελθόν ειδικά στο τμήμα της εποπτείας και της ρύθμισης να αναφερθώ κυρίως ε, σε αυτό το τστάτο εδώ πέρα από την πρώτη εκθεσή μου το 2002 στο επεξηγηματικό σημείωμα έλεγα Η εισηγήτρια στοιχηματίζει πως σε μία δεκαετία θα υπάρχει ευρωπαϊκό ρυθμιστικό όργανο, γιατί αυτό ήταν το όνειρό μου τότε, ότι θα πρέπει να οδηγηθούμε σε ευρωπαϊκή εποπτεία ειδικά για τους πιο μεγάλους παίκτες που ήδη τότε κυριαρχούσαν στην ε, αγορά και θυμάμαι πως ε, πολλοί μου είχαν πει τότε ε, πως πρώτα απ' όλα θα χρειαζόταν μια κρίση πριν μπορέσουμε να μπούμε σε μια τέτοια συζήτηση για την δημιουργία ευρωπαϊκής εποπτείας. Και αυτό ακριβώς συνέβη. Τώρα δεν θα σας δείξω όλες τις διαφάνειες. Θα σας αναφέρω διάφορα σημεία από διάφορες εκθέσεις, από την έκθεση του 2002, η οποία δεν ανέφερε ξεκάθαρα την επιθυμία ευρωπαϊκής ε, εποπτείας γιατί δεν το ήθελε αυτό η πλειοψηφία το 2005 ήδη ανέφερα κάποια προτίμηση το σύστημα αυτό των δύο επιπέδων ε, για ευρωπαϊκή εποπτεία των μεγάλων οργανισμών, τον κύριο Νόιε και ήταν κατά και νομίζω πως αυτό ε, έπρεπε ε, να γίνει λόγω ακριβώς αυτού του ζητήματος της ε, ρύθμισης ε, σε μια απόσταση από το εθνικό επίπεδο και τους εθνικούς πρωταθλητές. Αλλά θα επανέλθω σε αυτό. Μετά αυτό το οποίο τελικά κάναμε ήταν ένα σύστημα ε, επιτροπών και συνεργασίας. Μετά είχαμε την έκθεση του πρώην συναδέλφου του κ. Μουσκά που αφορούσε την συγκέντρωση στον χρηματοοικονομικό τομέα. Στην έκθεση αυτή λέγαμε ήδη πως θεωρούσαμε πως ε, συντονισμός ε, και συνεργασία δεν θα αρκούσε για να αντιμετωπίσουμε μια σοβαρή κρίση και ήδη σε αυτή την έκθεση προσπαθήσαμε να πείσουμε την Κομισιόν και το Συμβούλιο πως έπρεπε να συσταθεί μια επιτροπή σοφών για να καταλήξουμε σε κάποιες προτάσεις για ένα ευρωπαϊκό σύστημα. Μετά είχαμε μια άλλη έκθεση δική μου το 2007 για το FSAP, το πρόγραμμα δράσης για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και εκεί πέρα έλεγα πως είχαμε περίπλοκες διατυπώσεις και ήπιες διατυπώσεις για το πώς θα έπρεπε να υπάρχει εποπτεία σε ευρωπαϊκό επίπεδο γιατί δεν υπήρχε μια κοινή άποψη, αλλά τουλάχιστον υπήρχε ως απειλή ότι αν ο συντονισμός και η συνεργασία δεν επαρκούσε πρέπει να σκεφτούμε τι θα γίνει με εποπτεία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό ήταν λοιπόν στην έκθεση του 2007. Μετά 2008 είχαμε την έκθεση με τον κύριο Ντανιάνου δεν, δεν βλέπω εδώ. Δεν λειτουργεί το σύστημα. Να το, το βρήκα. Νομίζω πως ε, γνωρίζετε το περιεχόμενο. Το ενδιαφέρον ήταν πως ε, ψηφίσαμε ε, αυτή την έκθεση μία εβδομάδα πριν την ε, κρίση της Lehman Brothers και μετά από την κρίση της Lehman Brothers έγινε η ε, Ολομέλεια. Οπότε κάποια σημεία καταψηφίστηκαν στην Επιτροπή αλλά υιοθετήθηκαν στην Ολομέλεια γιατί είχε μεσολαβήσει η κρίση η οποία έπεισε τον κόσμο ότι κάτι έπρεπε να γίνει και τα ζητήματα αυτά πέραν σύνδεση του μάκρο και του μικρο επίπεδου που τώρα περιέχονται στην έκθεση Τελαροζιέρ και τις ε, προτάσεις της Κομισιόν αφορούσε ειδικά τις υποχρεωτικές επιτροπές και τις υποχρεωτικές εξουσίες διαμεσολάβησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό ήταν ένα από τα ευαίσθητα ζητήματα που αρχικά καταψηφίστηκε στην Επιτροπή Οικονομικών Θεμάτων και το άλλο ζήτημα ήταν βεβαίως ανεξάρτητη πρόεδρη και αντιπρόεδρη για τις ευρωπαϊκές αυτές επιτροπές για να υπάρχει έτσι ένα, κάποιο άλλο επίπεδο πέραν του εθνικού. Λοιπόν, μετά, όπως σας είπα, ε, αυτά τα ζητήματα τα ανέφερε και η εκθεσή Ντέλα Σε ένα ποσοστό 95% κάλυπτε πράγματα τα οποία είχαμε προτείνει στην έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά σαφώς η έκθεση Ντέλα ήταν μετά την κρίση και ήταν διαφορετικό το ε, πλαίσιο στην έκθεση Ντέλα και θα ήθελα αυτό να το αναφέρω και να εστιάσω εδώ πέρα, σαφώς ε, υπήρχε το δίλημα πως μπορούμε να έχουμε είτε περισσότερη Ευρώπη και συντονισμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο ή ο καθένας για την πάρτη του σε εθνικό ε, επίπεδο και αυτό ήταν άλλο ένα σημαντικό μήνυμα που ήθελα να τονίσω δηλαδή πρέπει να ξεκινήσουμε σταδιακά αλλά να ξεκινήσουμε αμέσως γιατί ασκήθηκε κριτική στην έκθεση για δεν ήταν αρκετά φιλόδοξη, αλλά από την άλλη ε, επικεντρώθηκε στα ε, πρακτικά ζητήματα και νομίζω πως αυτό είναι ακόμα σημαντικό. Βεβαίως ε, έχουμε και την έκθεση Τέρνερ που είναι και αυτή στο ίδιο δίλημα, περισσότεροι. Ευρώπη ή περισσότερες ε, εθνικές αρμοδιότητες, αλλά βεβαίως ε, μιλούσε και για συντονισμό και συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο μεταξύ των, ε, Ευρωπαίων, των εθνικών εποπτικών αρχών, αλλά χωρίς να μεταφερθεί αρμοδιότητα στο μακροεπίπεδο δηλαδή στην εποπτεία τραπεζών από το εθνικό στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Και αυτό ακούσαμε σήμερα και από τον επικεφαλής της Μπάφιν τον κύριο Νόγιε πως είναι κάτι το οποίο ακόμα τα κράτη-μέλη δεν θέλουν να κάνουν. Επίσης και στη ΣΥΠΑ υπάρχει μια αναλογική συζήτηση, είναι κατακαιρματισμένο το τοπίο Σοκαρίστηκα λίγο από αυτό το οποίο είπε ο κ. πως το σύστημα ήταν καλό της εποπτείας, δηλαδή σε εθνικό επίπεδο. Και πως η Κεντρική Τράπεζα τον ΗΠΑ δεν ε, έκανε τίποτα, γιατί βεβαίως σαφώς εδώ πέρα υπήρχε μία σύνδεση μεταξύ της Wall Street και της Ομοσπονδιακής Τράπεζας Νέα Υόρκη. Αυτό ακριβώ ήταν το πρόβλημα που είχαμε. στι ΔΕΗ είπα ένα νέο στοιχείο είναι αυτή η ιδέα Ομπάμα και Βόλκερ περί ανωτά του ορίου στο μέγεθος των ε, τραπεζών και να υπάρξει περιορισμός ε, της ε, ιδιωτική δραστηριότητας των τραπεζών για να περιοριστεί. Αυτή η δραστηριότητα μπορούμε να την περιγράψουμε ως καζίνο στον τομέα και αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη στις ευρωπαϊκές ε, συζητήσεις. Ε, οπότε αυτή συμπεριφορά των ρυθμιστικών αρχών υπάρχει και στις ΗΠΑ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή είναι πάρα πολύ ε, στενές οι σχέσεις εποπτευομένων και εποπτών, ο, καθώς τα κράτη-μέλη βεβαίως έχουν εθνικά συμφέροντα, ο κλάδος έχει γίνει πάρα πολύ σημαντικό τμήμα της εθνικής ε, ε, οικονομίας, γι' αυτό θέλουμε να παραμείνει σε εθνικό επίπεδο η αρμοδιότητα. Ένα άλλο στοιχείο βεβαίως είναι το ότι αλλάζουν συχνά θέσεις μεταξύ των επιχειρήσεων και των εποπτικών αρχών οι ίδιοι άνθρωποι. και μεταξύ των εταιριών πιστοληπτικής αξιολόγησης και γενικά κινούνται στον κλάδο. Οπότε εκεί είναι το, το ευαίσθητο ζήτημα. Δηλαδή η ανεξαρτησία, η υποχρεωτική διάδοση των πληροφοριών και η δεσμευτική διαμεσολάβηση και επίλυση διαφορών. Και τώρα κάτι κάνει το Κοινοβούλιο για π.χ. ασχολείται με την υπόθεση φόρτης, βλέπετε εκεί πέρα πως η ε, ανταλλαγή προφοριών γινόταν τα Σαββατοκύριακα όταν ασχολούνταν με, ε, το πρόβλημα Άμπεν Άμρο και Φόρτη, το ίδιο και με την Ισλανδία. Δεν υπήρχε λοιπόν, βλέπετε εκεί πέρα αρκετή εμπιστοσύνη στις ρυθμιστικέ αρχές. Το ζήτημα αυτό λοιπόν των στενών σχέσεων είναι και βεβαίω το ότι υπάρχει και η κυριαρχία της πλευράς του πολιτή στην αγορά αυτή. Και το βλέπουμε και εδώ πέρα και στις Βρυξέλλες πως υπάρχουν εκατοντάδες ε, ειδικοί από πλευρά των πολιτών και μια χούφτα μόνο άνθρωποι που εκπροσωπούν τα συμφέροντα των ε, αγοραστών ειδικά όσον αφορά το, τους χρήστες, ε, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ε. και οι θεσμικοί επενδυτές ε, συνταξιοδοτικά ταμεία δραστηριοποιούνται μόνο όσον αφορά την πλευρά της πώληση και όχι τόσο πολύ από την πλευρά του αγοραστή. Και εκεί πέρα λοιπόν πρέπει να διασφαλίσουμε πως ε, θα υπάρχει αυτή η συνεισφορά ε, και όσον αφορά το ρυθμιστικό κομμάτι και την υποκτία για να είναι πιο ισορροπημένη η κατάσταση. Και αυτό ε, το υιοθέτησα και σε μία από τις εκθέσεις μου Λέγαμε δηλαδή στην Κομισιόν να δημιουργήσει μια σχετική γραμμή στον προπολογισμό, κάτι το οποίο έχει το Κοινοβούλιο την, την δύναμη να, να κάνει. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Επίσης, τελευταία διαφάνεια, Βόλφα, τα βήματα τα οποία προτείνω εγώ για το μέλλον. Προτείνω μια μεικτή επιτροπή με τα Εθνικά Κοινοβούλια για να δούμε σε ποιο βάθος να κάνουμε μια έρευνα για το τι συνέβη στην ε, κρίση, ειδικά όσον αφορά την μη ανταλλαγή πληροφοριών και την έλλειψη εμπιστοσύνης. Ε, δεύτερον, να συμπεριληφθεί η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού να ξεκινήσει ξανά η έρευνα την οποία έχουμε ζητήσει πολλές φορές ε, τα τελευταία χρόνια να μελετηθεί ο χρηματοοικονομικός τομέα η Νέλη Κρούς παραδέχτηκε πως έπρεπε να το είχε κάνει αυτό, ειδικά όσον αφορά τις εταιρείες αξιολόγησης τη ικανότητας. Ε, μπορεί λοιπόν νομίζω να γίνει μια τέτοια έρευνα κατόπιν το είπα ήδη να υιοθετηθεί η πρόταση της ε, Κομισιόν να ξεκινήσουμε με τις ε, επιτροπές ε, επίπεδου 3 και μια νέα υπηρεσία γιατί εργαζόμαστε βράχη πρόθεσμα και να δημιουργηθεί πάλι μια ομάδα σοφών για να επεξεργαστεί τα περαιτέρω βήματα ειδικά για την κορυφή ε, της ε, αγοράς, για τις ε, 4-5 μεγα, εκεί οργανισμούς χρηματοοικονομικούς που παίζουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο και άλλη μια ομάδα υψηλού επίπεδου για να βρει μια καλύτερη δομή για τον καταναλωτή θα λέγαμε και για την προστασία των επενδυτών και για την νομοθεσία και την εποπτεία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σε ευχαριστώ και τον λόγο έχει ο Ερκύρα Σούκε. Μεγάλη χαρά για μένα, μεγάλη τιμή για μένα να είμαι παρόν. Και βέβαια είναι, είναι δύσκολο για μένα να μιλώ τελευταίος και να είμαι κάποιος ο οποίος έρχεται από την άλλη άκρη του φράκτη κατά κάποιο τρόπο ο διευθύνων σύμβουλος μιας μη ευρωπαϊκής μιας ε, τράπεζας η οποία λειτουργεί στην ε, Σουηδία, στη Σουηδία, στην ε, Λετωνία και τη Λιθουανία και η οποία έχει λειτουργήσει επιτυχώς τα τελευταία χρόνια και είμαι ο ο πρόεδρος της Εποπτικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Αποταμιεύσεων Εμείς ήμασταν μια, ένα τράπεζα ταμιευτηρίου στο παρελθόν, αλλά τώρα πια έχει πάψει να είναι μόνο μια τέτοια τράπεζα ταμιευτηρίου. Εν πάση περιπτώσει αυτή η Επιτροπή εποπτεύει περίπου το 1 τρίτο των Ευρωπαϊκών Πιστοτικών Ιδρυμάτων. Είναι πάρα πολύ επίκαιρη συζήτηση για τα θέματα αυτά, γιατί έχουμε αυτό το οικονομικό τσουνάμι, το οποίο ίσως έχει ξεπεράσει την κορυφή του αλλά θα επέλθει ένα άλλου είδου τσουνάμι ρυθμιστικού χαρακτήρα και δεν ξέρουμε πώς θα αντιδράσουμε ανάμεσα στα δύο. Αυτό που μας ενδιαφέρει εμά είναι να αντιμετωπίσουμε πρακτικές ανάγκες και πρακτικά προβλήματα ως ε, ε, ευρωπαϊκές ε, τράπεζες στο λιανικό τραπεζικό χώρο Θέλουμε λοιπόν να εξετάσουμε τα θέματα του ρυθμιστικού πλαισίου, τα οποία αναφέρθηκαν προηγουμένως, και της κατεύθυνσης στην οποία θα αναλάβει αυτό το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο. Για το ίδιο το πλαίσιο, προφανώς θεωρούμε ότι η κατεύθυνση που ακολουθείται είναι σωστή, και παρά το γεγονός ότι είμαστε περιφερειακού χαρακτήρα, μας ικανοποιεί αυτή η διαμεθοριακή αντιμετώπιση και θα θέλαμε να υπάρχει ένα ίδιο είδος κανόνων για όλους. Ένα άλλο στοιχείο που αφορά την ευρωπαϊκή αγορά είναι το εξής, το οποίο έχει ένα ποικίλο χαρακτήρα. Ένα από το στοιχεία που έδειξε η κρίση είναι ότι η διαφοροποίηση αυτή είναι ένα ισχυρό στοιχείο, ένα στοιχείο σταθερότητας και όχι ένα πρόβλημα. Είναι λοιπόν πιστεύω κίνδυνος για αυτή την πολυμορφία το να έχουμε μια ενιαία ρυθμιστική αρχή η οποία τα καλύπτει όλα. Οι μικρές τράπεζες λοιπόν δεν έχουν παίξει σημαντικό ρόλο στη χρηματοοικονομική κρίση. Πολλοί από, εμά βρεθήκαμε μπλεγμένοι στη μέση αυτής της κρίσης για πολλούς λόγους, για διάφορους λόγους. Γιατί η παγκόσμια κρίση ε, επηρέασε πάρα, πολλές, ε, πάρα πολλά ψηφιακά ιδρύματα. Η παγιοποίηση λοιπόν είναι απαραίτητη στο πιστοτικό σύστημα, αλλά επίση πρέπει να διατηρηθεί και η πολυμορφία η οποία έχει σταθεί πολύ θετική στο παρελθόν. Όταν ερχόμαστε στο θέμα της, του συντονισμού των ρυθμιστικών αρχών κατά τη διάρκεια της κρίσης, μπορώ να σας δώσω ένα πραγματικό παράδειγμα από τις ε, χώρες της Σκανδιναβίας και της Βαλτικής. Έχουμε μονάχα θετικά σχόλια για το ρόλο των ρυθμιστικών αρχών. Ήταν πάρα πολύ θετική η δράση των Σουηδικών ρυθμιστικών αρχών που ήταν έγκαιρη η παρέμβασή τους και επιτυχής. και ίσως αυτή η πατερναλιστική στάση του ρυθμιστικού συστήματος στη Σουηδία που δεν θα ήταν αποδεκτή σε άλλες χώρες ήταν πολύ θετική για την αντιμετώπιση της κρίσης. Υπήρξε λοιπόν πλήρης ανταλλαγή πληροφοριών, είχαν απόλυτα επίκαιρη πληροφόρηση οι ρυθμιστικές αρχές, δεν είχαν επικάλυψη μεταξύ τους και εμείς ως τράπεζα που υφίστατο τη ρύθμιση θεωρούμε ότι είχαμε μεγάλη υποστήριξη από τις ρυθμιστικές αρχές σε όλη τη διάρκεια της κρίσης κράτησε μια συνεπή πορεία και έχουν κρατήσει μια ενιαία στάση. Εκεί λοιπόν που προσπαθούμε να δημιουργήσουμε μια νέα δομή στην Ευρώπη, ίσως θα πρέπει να τονίσω ότι τουλάχιστον στη δική μας περιοχή η ρύθμιση δούλεψε πολύ καλά. Τώρα έρχομαι στο προτινόμενο νέο σύστημα. Εδώ θα ήθελα να ξεκινήσω λέγοντας Αν δούμε λοιπόν τι γίνεται στην ε, διαχείριση της ρευστότητα και στην διαφάνεια που είναι απαραίτητα στοιχεία σε ένα καιρό ε, κρίσης, νομίζω ότι αυτές είναι οι σωστές κατευθύνσεις για μια ρύθμιση. Αλλά προτού αυτές οι προτάσεις μπορέσουν να υλοποιηθούν και να αποτελέσουν τμήματα του ρυθμιστικού συστήματος, πρέπει να σκεφτούμε και μερικές από τις πιο λεπτομεριακές ανησυχίες που υπάρχουν. Στους κανόνες για το κεφάλαιο που προτείνονται εισάγονται νέοι, νέα ποσοστά μόχλευσης. Νομίζουμε ότι αυτό είναι ένα βήμα προς τα πίσω. Ναι, το τωρινό σύστημα έδειξε είναι κάτι το οποίο μας γυρίζει πίσω δεκαετίες. η μόχλευση δεν είναι ευαίσθητη στο, στους κινδύνους και αν δεν υπάρχει ευαισθησία προς τους κινδύνους στο μακρο, μακροσκοπικό ή μικροσκοπικό επίπεδο, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε αυξανόμενο ηθικό κίνδυνο και σε αυξημένη ανάληψη κινδύνων. αλλά υπάρχουν πολλά τα οποία μπορούν να γίνουν με το να εφαρμοστούν άλλα μέτρα και όχι να γυρίσουμε σε ε, ανώτατα, ανώτατα ποσοστά μόχλευσης που μας γυρίσουν δεκαετίες πίσω. Επίσης, στον τομέα της χρηματοδότησης, νομίζω ότι η σωστή κατεύθυνση έχει ακολουθηθεί. Αν δούμε λοιπόν τις προτάσεις οι οποίες έχουν διατυπωθεί πιστεύω ότι προς το παρόν δεν είναι σωστά σταθμισμένες και νομίζω ότι χάνει το στόχο, του, το στόχο της ρύθμιση με μεγάλη απόσταση. Η παραδοσιακή τραπεζική δραστηριότητα έχει μειωμένη ευαισθησία σε σχέση με την αγορά. Δηλαδή τα περισσότερα από τα δάνεια ε, χρηματοδοτούνται από τις καταθέσεις, ενώ στις νέες ρυθμίσεις έχουμε μια <coughs> νέα αντιμετώπιση που λέει ότι η τράπεζα αυτή θα πρέπει να πηγαίνει στις διεθνείς χρηματαγοράς και να δανείστε το 15 με 20% ή περισσότερο του χαρτοφυλακίου του. Δεν καταλαβαίνω ποιο είναι καλό σε αυτή τη ρύθμιση. Εμείς λοιπόν δεν είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι με την στάθμιση της δομής που αναφέρεται. Εγώ προφανώς <coughs> θέλω να κάνω το πιστοτικό μου ίδρυμα ισχυρό και ανθεκτικό στις ε, αλλαγές που προέρχονται από τη ρύθμιση. Οι μελέτες οι οποίες έχουν γίνει, οι οποίες οδηγούν σε νέες απαιτήσει σε επίπεδο κεφαλαίων μπορεί να οδηγήσουν σε ένα συνολικό ε, έλλειμμα στην ευρωπαϊκή τραπεζική αγορά σε επίπεδο 1,5 <clears throat> με 3, 3 εκατομμύρια ευρώ. Πού θα έρθουν λοιπόν αυτά τα χρήματα και φοβάμαι ότι τα μικρά πιστοπτικά ιδρύματα θα βρεθούν χωρίς καμία άμυνα μέσα στα πλαίσια αυτά. Εμείς λοιπόν σαν μικρή τράπεζα θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε ε, μια δύσκολη κατάσταση γιατί η, τα δάνεια τα οποία διαχειριζόμαστε και οι φάκελοι που, διαχειριζόμαστε, που διαχειριζόμαστε δεν έχουν να κάνουν με τις αγορές. Υπάρχει λοιπόν ένας μεγάλος κίνδυνος σε αυτές τις ρυθμίσεις να περιστήλουν το δανεισμό στις επιχειρήσεις. Βλέπω ότι ο χρόνος τελειώνει και προσπαθώ, θα προσπαθήσω να κλείσω σε σχέση με το ρυθμιστικό πλαίσιο και επίσης σε σχέση με την νέα ρύθμιση από την Επιτροπή της Βασιλείας. Νομίζω ότι εκεί έχουν αντιμετωπίσει τα σωστά θέματα, αλλά παρόλα αυτά πρέπει να γίνουν πολλά με μελέτες αντικτύπου, ώστε να μην αντιμετωπίσουμε πάλι μια νέα κρίση. Για την χρηματοδότηση όμως των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και τη χρηματοδότηση ε, μικρών ποσών θα πρέπει να υπάρξει ιδιαίτερη μνήμα γιατί αυτό δεν έχει αντιμετωπιστεί ακόμα στην αντιμετώπιση της κρίσης. Ευχαριστώ και τους τρεις ομιλητές μας. Έχουμε τώρα κάποια λεπτάκια για ερωτήσεις. Επειδή μίκρινε η ομάδα θα πάρουν το λόγο όσοι εδώ πρώτα απ' όλα. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ακούσω τις ε, αντιδράσεις του κυρίου Πέρσον για τα όσα είπε ο τελευταίος ομιλητής. Εγώ άκουσα τις επικρίσεις για τη Βασιλεία 2, για τους τρεις πυλώνες. Τι σημαίνει όταν ε, για το μέλλον των εργασιών μάλλον της Βασιλείας 2 πιστεύετε πως πρέπει να ξαναρχίσουν από την αρχή και θα θέσω και την ίδια ερώτηση που, έστε, που έθεσα στον ε, κύριο Νοαγέ. Ότι μια από τις δυσκολίες των Ευρωπαϊκών Τραπεζών είναι ότι είχαν ε, γίνει συμφωνίες μονομερείς, ε, ενώ οι Αμερικανοί είχαν επηρεάσει την συγγραφή των συμφωνιών. Αυτές οι συμφωνίες δεν θα έπρεπε να είναι συνθήκες. Έπειτα, σε σχέση με τη ρευστότητα ε, και την υπερβολική ρευστότητα ή την έλλειψη ρευστότητας. Τι μπορούμε να κάνουμε. Για το θέμα τώρα της ΦΕΔ, το μόνο πράγμα που είναι προφανές ε, είναι η σύνδεση ανάμεσα στην τοπική ΦΕΔ και την κεντρική ΦΕΔ είναι ενδιαφέρον ως δομή διακυβέρνησης ε, σύνδεση ε, ανάμεσα στο τοπικό και το ομοσπονδιακό επίπεδο. Το μόνο πράγμα που είναι ενδιαφέρον, δεν χρειάζεται να υπερεκτιμούμε Λοιπόν, για την ε, πλευρά των πωλήσεων. Εσεί τι πιστεύετε για την ιδέα ότι ανεξάρτητα από το τι κάνουμε εμεί για τις ρύθμι, τη ρύθμιση τη απαιτήσει περικεφαλαίων κτλ, τη δημιουργία μια υπηρεσία προστασία των καταναλωτών και των επενδυτών στον τομέα των χρηματοπιστωτικών αγορών και θα πρέπει αυτό να γίνει και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τρίτη παρατήρηση, αλλά αυτό είναι μια μακρά συζήτηση μεταξύ μα, ότι εγώ δεν συμφωνώ απόλυτα με την ιδέα ότι πρέπει να γίνεται μια απόλυτα ολοκληρωμένη εποπτεία για τους μεγάλους παίκτες γιατί στους Lehman Brothers, στην ε, AIG και τα λοιπά όλοι αυτοί οι φορείς δεν θα είχαν εντοπιστεί ως συστημική κίνδυνη και ωστόσο από αυτούς προήλθε η δυσκολία. Τελευταία παρατήρηση για τους τρεις παρεμβαίνοντες, τους τρεις ομιλητές. Μιλάμε για το μέλλον της εποπτείας εντός της Ένωσης. Εσείς δεν μιλήσατε για το clearing του OTC και του CDS για το μέλλον του management και του burden sharing. Και ωστόσο για μένα αυτά είναι πράγματα τα οποία θα πρέπει να εξετάσουμε πολύ προσεκτικά. Δεν θα σας προξενήσει η κατάπληξη ότι είναι πολλές ερωτήσεις ε, βεβαίως και πολύ σημαντικές. Κοιτάξτε, εγώ ήμουν ένας από τους πρώτους που πρότειναν την Βασιλεία 3 το 2004. Τώρα όλοι μιλάνε για τη Βασιλεία. Ε, 3, με συγχωρείτε. Τώρα όλοι μιλάνε για τη Βασιλεία 3. Αλλά δεν είμαι τόσο σίγουρο γιατί βεβαίω ένα από τα καλά τη Βασιλεία 2 έχει πολλά ελαττήματα. Αλλά πάρα πολύ ευσυνείδητοι άνθρωποι δούλεψαν πάνω σε αυτήν και ένα από τα καλά της είναι ο πυλώνας 2 και η διακριτική ευχέρεια στην εποπτεία και πολλά πράγματα μπορούν να αλλάξουν στη Βασιλεία 2 χρησιμοποιώντας την διακριτική ευχέρεια στην εποπτεία. Μπορούν δηλαδή οι εθνικές εποπτικές αρχές να έχουν κανόνες με κάποια διακριτική ευχέρεια το δεύτερο ζήτημα για τις συνθήκες, εγώ δεν είμαι νομικός του Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου. Δεν ξέρω ε, εάν ε, θα πρέπει να υπάρχει μια συνθήκη ή όχι. Δεν είμαι ειδικό. Εκεί που θα διαφωνούσα με ε, τους συναδέλφους μου είναι πως δεν χρειάζεται ένα ποσοστό μόχλευσης και αντίστοιχη χρηματοδότηση εάν είμαστε απολύτως σίγουροι πως μπορούμε να υπολογίσουμε σωστά τον κίνδυνο. Άρα σαφώς το χρειαζόμαστε γιατί δεν μπορούμε να υπολογίσουμε σαφώς τον κίνδυνο. Βεβαίως είναι μια πολύ βαριά προσέγγιση αν το να έχουμε ένα ποσοστό μόχλευσης. Αν θεωρούμε ότι μπορούμε να είμαστε πάρα πολύ καλοί, δεν το χρειαζόμαστε. Εάν δεν μπορούμε να υπολογίσουμε σωστά το κίνδυνο, το, το χρειαζόμαστε. Νομίζω είναι σημαντικό αυτό το στοιχείο. Τώρα όσον αφορά τον ανταγωνισμό, νομίζω πως Φοβόμασταν πάρα πολύ να εφαρμόσουμε κανόνες ανταγωνισμού στις τράπεζες και θα πρέπει να είμαστε πιο επιθετικοί ως προς αυτό. Επίσης θα προειδοποιούσα το να μην ε, λέμε πως κάποιες τράπεζες ε, είναι πολύ μεγάλες ε, για να αποτύχουν και αν ήταν πιο μικρές οι τράπεζες δεν θα υπήρχε το πρόβλημα. Αλλά σε μια κρίση δεν έχει τόση σημασία το μέγεθος γιατί σε μια κρίση το πολύ μεγάλο για να αποτύχει είναι αρκετά μικρό τελικά και δυστυχώς εγώ ξέρω πιο πολύ την ε, οικονομική βρετανική ιστορία αλλά η μεγαλύτερη κρίση που είχε η Βρετανία ήταν των μικρών τραπεζών όπου η Τράπεζα της Αγγλίας έπρεπε να σώσει 30 μικρές τράπεζες. Εάν οι μικρές τράπεζες κάνουν όλες λίγο πολύ το ίδιο πράγμα, αυτό είναι πολύ πιο επικίνδυνο από μια μεγάλη τράπεζα Οπότε χρειάζεται περισσότερος ανταγωνισμός, περισσότερη επίβλεψη σε μεγάλες βεβαίως ε, κίνδυνες, αλλά, ε, σε μεγάλες κίνδυνες τραπεζές, αλλά αυτό δεν είναι πανάκια. Πρέπει να είμαστε πολύ πιο εύρωστοι, αν θέλετε, στην υποδομή της αγοράς, να υπάρχει κεντρική εκαθάριση και τέτοια μέσα. Αυτό είναι πολύ πιο σημαντικό από το να υπάρχουν κάποιες... Γιατί ε, κάποιες βεβαίως κάποιε αλλαγές δεν θα είναι σέρευστο, αλλά πρέπει να υπάρχει κεντρική εκαθάριση και διακανονισμός. και θέλεις και εσύ να Ναι. Δεν θα μπορούσα να συμφωνώ περισσότερο για το θέμα του ανταγωνισμού, αλλά χαίρομαι που επανέρχεται το θέμα αυτό, γιατί είχα θέσει και στο παρελθόν ερωτήματα για αυτό το ζήτημα. Είπατε ότι οι τραπεζίτες ρίξανε όπλα μαζικής καταστροφής στο, στους καταναλωτές, στους ε, επενδυτές, αλλά ήταν προσεκτικοί για να προστατευτούν από τα δικά τους όπλα προτού εκραγούν. Επομένως και εδώ θα πρέπει να εξετάσουμε τις συγκρούσεις συμφερόντων με στο χρηματοπιστωτικό τομέα τους τραπεζίτες της Wall Street. Γιατί δεν ήταν τελείως τυχαίο ότι κάποιες από τις επενδυτικές εταιρείες ε, ε, επέζησαν γιατί είχαν καλύτερη αξιολόγηση κινδύνου. Ήταν καλύτεροι λοιπόν από τους ανταγωνιστές τους. Και φυσικά ήταν απλώς πιο ισχυρό το μονοπόλιο το οποίο είχαν στους τομείς αυτούς για το φορέα, ο οποίος προστατεύει, θα πρέπει να προστατεύσει τους καταναλωτές. Εγώ δεν υποστηρίζω να υπάρξει ένας χωριστός φορέας. Και συμφωνώ με αυτά που είπε η κυρία από την Alliance. Είναι απαραίτητο να είναι πιο καλά ενσωματωμένος αυτός ο φορέας με άλλους φορείς, γιατί είναι απαραίτητο μέσα στις ε, ρυθμιστικές αρχές να γνωρίζουμε και ποια είναι η άποψη όχι μόνο των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, αλλά και από τις ίδιες τις αγορές και τους ε, ρυθμιστές των οικονομικών αγορών. Από τις οι φορείς λοιπόν προστασίας για τους καταναλωτές θα πρέπει να γνωρίζουν τι γίνεται από τις αρχές εποπτείας των χρηματαγορών που έχουν μία άλλη προσέγγιση από ό,τι έχουν οι κεντρικές τράπεζες. Και η μικροπροληπτική επόπτες. Γι' αυτό θα ήθελα να υπάρχει μια εγκάρσια προσέγγιση και όχι κατά οικονομικούς χρηματοπιστωτικούς τομείς. Και κοιτάζοντας εν τάχει το έγγραφό σας, νομίζω ότι κάποιος από τους ε, εμπειρογνώμονες είχε κάνει μια έκκληση να περνάνε τα πάντα από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. <clears throat> Εγώ δεν θα υποστήριζα κάτι τέτοιο γιατί υπάρχει το φαινόμενο της ρυθμιστικής σύλληψης, όπως λέμε σε εισαγωγικά, ότι κατά κάποιο τρόπο μπορεί να καταληφθεί μια ρυθμιστική αρχή από αυτούς τους οποίους υποτίθεται ρυθμίζει. Και το τελευταίο σημείο αυτό για την μακροπολιτική εποπτεία ότι πρέπει να γίνει σε πιο εθνικό επίπεδο. Εγώ πιστεύω ότι πράγματι έχει νόημα να το κάνουμε αυτό σε εθνικό επίπεδο, αλλά εγώ κάνω μια διάξη μεταξύ των 40-50 μεγάλων πιστοτικών ιδρυμάτων που επέχουν φυσικά συστημικό κίνδυνο. Βέβαια και μια μικρή τράπεζα μπορεί να έχει συστημικό κίνδυνο, αλλά υπάρχει μεγαλύτερος κίνδυνος να επηρεάσουν τους ρυθμιστές, να γίνει λεγόμενη σύλληψη, ρυθμιστική σύλληψη, μπορούν να έχουν μεγαλύτερη επιρροή στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας των χωρών τους κτλ. Υπάρχει μεγαλύτερος κίνδυνος λοιπόν να μεταφέρεται αυτό το θέμα της ρύθμισης στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να υπάρχει ένα καλύτερο αποτέλεσμα παρά αν παραμείνει σε εθνικό επίπεδο ακριβώς για, λόγω αυτού του φαινομένου ότι μπορούν να ασκήσουν μεγαλύτερη πίεση σε εθνικό επίπεδο. Ελπίζω να είμαι σαφής. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να σας ευχαριστήσω, λέει κύριε κυρία για τις πάρα πολύ ενδιαφέρουσες ε, παρουσιάσεις τους. Έχω την εξ, τα εξή ερωτήματα. Πρώτο για τη Βασιλεία 2. Μιλάμε τώρα ήδη για τη Βασιλεία 3, αλλά στην Αμερική δεν, έχουμε, δεν έχουν καταφέρει ακόμα να εφαρμόσουν τη 2. Άσε και τη μία ακόμα που εμείς στην Ευρώπη την έχουμε εφαρμόσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Λοιπόν, είναι γεγονός ότι η χρηματοοικονομική κρίση ξεκίνησε στι Ηνωμένε Πολιτείε και αυτό συνδέεται με το γεγονό ότι δεν είχαν φτάσει στο επίπεδο τη Βασιλεία 2. Επίση, τώρα θα ήθελα να σταθούμε στο θέμα των, των μεσαίων επιχειρήσεων και πιστεύω ότι αν υπάρχει μια υπερκυκλική αντιμετώπιση, αν έχει κανείς αρκετά διαθέσιμα χρήματα, μπορεί να αποκτήσει και περισσότερα. Ενώ οι εταιρείε οι οποίες δεν έχουν αρκετά χρήματα, δεν έχουν αρκετά κεφάλαια, αυτές έχουν πραγματικά έλλειψη και παθαίνουν ασφυξία από έλλειψη κεφαλαίων και τελικά χάνονται αυτές. Επομένως, το θέμα δεν είναι η παροχή των ε, υπηρεσιών, η ρευστότητα. Το θέμα είναι αν μπορεί να υπάρξει η ροή κεφαλαίων με έναν τρόπο ο είναι τελείως αδιαφανής. Νομίζω ότι εδώ πρέπει να κάνουμε μια διάκριση και γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να δώσουμε μια διαφορετική αντιμετώπιση σε περιφερειακές τράπεζες οι οποίες τροφοδοτούν τις τοπικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι οποίες αντιμετωπίζουν μονάχα ένα περιφερειακό περιβάλλον και πρέπει να τι αντιμετωπίσουμε διαφορετικά από τι εταιρείε τι τράπεζε οι οποίε δρούν σε διεθνέ επίπεδο. Επίση, οι εταιρείε πιστοληπτική αξιολόγηση. Νομίζω ότι είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα το γεγονό ότι έχουν αδιαφανή κριτήρια αξιολόγηση, τα οποία δεν μπορεί κανεί να γνωρίζει με ποιο τρόπο γίνεται και οι οποίε είναι δυνατόν να έχουν τα ιδιαίτερα συμφέροντά του λόγω τη ιδιοκτησία του από μεγαλύτερε εταιρείε και με τον τρόπο αυτό δημιουργούν προβλήματα για τις ε, χρηματαγορές. Μπορεί ας πούμε μια επιχείρηση να έχει τριπλό αλφα σαν αξιολόγηση και να έχει ε, χρεοκοπήσει, ενώ αυτές που ήταν β μείον να έχουν επιβιώσει την κρίση. Λοιπόν, είναι απαραίτητο να ξαναδώσουμε την ευθύνη στους επικεφαλείς των τραπεζών και όχι να την κάνουμε πάσα στις εταιρείες πιστοληπτικής αξιολόγησης. Ελπίζω λοιπόν ότι δεν θέλουμε να προωθήσουμε μια οργανωμένη μορφή ανευθυνότητας και έρχομαι στο ερώτημα Πρώτον, πώς θα δημιουργήσετε κριτήρια διαφάνειας, Δεύτερον, πώς θα προωθήσετε τον ανταγωνισμό. Και τρίτον, πώς θα αποφύγετε τις συγκρούσεις συμφερόντων σε επίπεδο ιδιοκτησία. Κυρία ο κύριος, και ο κύριος μετά. Uh, Εγώ δεν θα έλεγα πως η Βασιλεία 2 έχει προκαλέσει υπερκυκλική ε, συμπεριφορά με όσον αφορά τη χρηματοδότηση μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Περισσότερο τμήμα ε, μπήκε στις ε, τράπεζες από τις διεθνείς αγορές κεφαλαίου και καθώς ε, αλλάζει βεβαίως γρήγορα το ρυθμιστικό πλαίσιο Και υπάρχει εδώ πέρα, πρέπει βεβαίως να δούμε τι θα γίνει όσον αφορά το πώς ε, θα επιβάλλουμε μια στη συμπεριφορά το στο μέλλον για το τι θα κάνουμε και με, τις, με τα εθνικά τους ανοίγματα. Οπότε, Να δούμε τώρα την περισσότερη αγορά μέσω της κρίσης, δεν ξέρω εάν έχει υπάρξει μια ιδιαίτερη επιδείνωση στον τομέα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Υπήρχαν κάποιες φούσκες όσον αφορά τα κίνητα. Αυτό ε, βέβαια ισχύει και στη ΣΥΠΑ και, στις, ε, και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπήρχε επίσης κάποια δυσκολία χρηματοδότησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αλλά η Βασιλεία 2 δεν νομίζω να παίξει κάποιο ρόλο εδώ. I would uh, beg to Εγώ ε, διαφωνώ με τον συνάδελφο. Ε, οι ρυθμιστικές αρχές λένε πως η Βασιλεία 2 δεν θα μπορούσε να είχε προκαλέσει το, πρόγραμμα, το πρόβλημα. Αλλά νομίζω πως δεν είναι έτσι τόσο σωστό αυτό, γιατί η αρχή της Βασιλείας 2 είναι ακριβώς η ευαισθησία στον κίνδυνο που είχε ξεκινήσει ήδη και προ Βασιλείας 2 όταν είχαμε την οδηγία κινδύνου αγοράς του 1995 οπότε οι ρυθμιστικές και υποδικές αρχές ε, εφαρμόζουν, ένα μέτρο ευαισθησίας στον κίνδυνο πριν από τη Βασιλεία 2 για να είμαι δίκαιος βεβαίως ένα πολύ σημαντικό κομμάτι αυτής της ευαισθησίας κινδύνου και αγοράς που είναι πολλά πράγματα είναι βεβαίως ε, η λογιστική ε, διαδικασία που και μαζί με την ευαισθησία στην αγορά έπαιξε ένα σημαντικό ρόλο στην ενισχύση της κυκλικής συμπεριφοράς και βεβαίως δικαίως επομίζεται και κάποιο το βάρος. Η συμπεριφορά αυτή σημαίνει πως όταν υπάρχει πτώση ή μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ή ευαίσθητη δανειζόμενοι θα έχουν πρόβλημα. Και γενικά πρέπει να προστατεύσουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις βεβαίως και τα στεγαστικά δάνεια, αλλά πρέπει να είμαστε προσεκτικοί γιατί ίσως έτσι να υπάρχει υπερβολικός δανεισμός χωρίς να υπάρχει μια ε, αρκετά μεγάλη βεσία στους κινδύνους. Να τελειώσω όμως με κάτι που ε, συμφωνώ με τον συνάδελφο όταν μιλάει βεβαίως για ποικιλομορφία δεν θα πρέπει να εξαφανιστεί αυτή από το ευρωπαϊκό χρηματοοικονομικό σύστημα γιατί είναι η πηγή της ρευστότητα. και ποικιλομορφία σημαίνει ότι κάποιο πρέπει να αγοράζει όταν όλοι οι άλλοι πουλάνε και για μένα για να, είμαστε, να υπάρχει έτσι μια διαφορά, μια ποικιλομορφία πρέπει να δούμε πώς αναλαμβάνουν κινδύνους ε, οι οργανισμοί και να σκεφτόμαστε και τα αποτελέσματα και όχι μόνο τις διαδικασίες. Ένα επικεντρωθούμε μόνο στις διαδικασίες θα εξαφανίσουμε τους μικρούς οργανισμούς και μόνο οι μεγάλοι που μπορούν να αγοράσουν μεγάλες τράπεζες δεδομένων θα επιβιώσουν. Äh, Έχουμε ακόμη δύο συναδέλφους, ο Λεσμίτ και Σβενκέκλου. Νομίζω μπορούμε να ακούσουμε τις ερωτήσεις μαζί και αν κάποια απευθύνεται σε κάποιον συγκεκριμένο. Ναι, ευχαριστώ. Εγώ απενθύνομαι στον κύριο Ρασούκε. Είπατε πως υπάρχει ένα ειδικό ρυθμιστικό πλαίσιο στη Σκανδιναβία και στη Βαλτική που λειτουργεί πάρα πολύ καλά και είχε έναν προληπτικό ρόλο, αλλά η Σουηδική Τράπεζα, η Βασιλική Τράπεζα είπε πως θα μπορούσε να λειτουργήσει καλύτερα γιατί υπάρχουν ε, προβλήματα σε κάποιες βαλτικές χώρες και θα μπορούσε να έχει λειτουργήσει ορολογητικά. Κάπου ήσασταν επιθετικοί όσον αφορά την αγορά ρευστότητα και το ερώτημά μου είναι εάν θεωρείτε πως οι τωρινές προτάσεις θα απέφευγαν αυτή την κρίση στις ε, σκανδιναβικές και βαλτικές χώρες. Και θα ήθελα να τελειώσω λέγοντας πως εγώ είμαι μέτοχος της Swedbank. Yes, a to Mr. Ναι, ένα ερώτημα στον κύριο Περσό. Δεν είναι μόνο ενδιαφέρον να ακούμε αυτά που λέτε, αλλά είναι και πολύ διασκεδαστικό. Ένα ακόμα ερώτημα. Αν πιστεύετε ότι υπήρχε υπερβολική ρευστότητα, συνολική ρευστότητα, κατά τη διάρκεια της κρίσης, κατά τη δική σας άποψη, Ποιο ήταν το αίτιο αυτής της υπερβολικής ρευστότητος, ποιες ήταν οι αιτίε του φαινομένου και ποιες είναι οι θεραπείες για αυτό το φαινόμενο, κατά την άποψή σας, και δεν λέω τίποτα άλλο γιατί έχουμε αργήσει ήδη. Νομίζω ότι είναι αρκετά δύσκολο αυτό το ερώτημα ούτως ή άλλως. Να προσπαθήσω να διευκρινίσω αυτό που είπα για τις ρυθμιστικές αρχές στη Σουηδία. Ήταν ότι ήταν πολύ καλή συνεργασία αλλά από μόνη της η συνεργασία δεν μπορεί να λύσει τα προβλήματα. Και την ανάγκη της κατανόησης του αν υπάρχει μία φούσκα η οποία διαστέλλεται. Μπορούμε να πούμε λοιπόν ότι τόσο οι ρυθμιστές όσο και οι παίκτες στην αγορά όλοι παραπλανήθηκαν. Εγώ απλώς αναφέρθηκα θετικά στην συνεργασία των ρυθμιστικών αρχών μεταξύ τους και με τις επιχειρήσεις στον πιστοτικό τομέα και πράγματι η μακροπροληπτική εποπτεία θα ήταν χρήσιμη για όλη την περιοχή μας. Υπάρχουν δύο, υπήρξαν δύο πηγές υπερβολικής ρευστότητας. Εγώ έχω υπεραπλοποιήσει λιγάκι τα πράγματα. Καταρχήν ήταν η νομισματική πολιτική της, Ευρωπαϊκής, της των ΗΠΑ που ήταν πολύ χαλαρή για πάρα πολύ χρόνο και δεύτερον ήταν τα οι υπερκυκλικές απαιτήσει κεφαλαίου των κεντρικών τραπεζών. Αυτά τα δύο. <clears throat> Τώρα, αυτό το οποίο προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε είναι ο υπερκυκλικός χαρακτήρας της ρύθμισης με αντικυκλικές απαιτήσει κεφαλαίου. Δεν μπορούμε όμως να αντιμετωπίσουμε την νομισματική πολιτική άλλων χωρών με εξίσου εύκολο τρόπο. Αγαπητοί συνάδελφοι, Νομίζω ότι το ορολόγιο μας δείχνει ότι φτάνουμε στο τέλος της συνεδρίασής μας. Θέλω να ευχαριστήσω τους, ε, τα μέλη του πάνελ για τις τόσο ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις τους και μας έχουν δώσει μια πολύ καλή εικόνα για την πραγματικότητα. Έχουμε λοιπόν πάρα πολύ τροφή για σκέψη για το μέλλον. Θα βρεθούμε πάλι στις 3.30. Όχι. Περβάνς, νόμιζα ότι είχε ήδη αντλήσει τα συμπεράσματά του ή όχι. Das tue ich doch nie. Das tue ich nicht. Okay. Να λάβει το λόγο τότε. Εγώ έθεσα ερωτήσεις αλλά δεν έχω κάνει τα πορίσματα. Πιστεύω ωστόσο πως στο τέλος μιας ακρόσης είναι σημαντικό να μπορέσουμε να καταγράψουμε τα όσα ακούσαμε και επί των οποίων θα πρέπει να επανέλθουμε στην έκθεση. Εγώ θέλω να πω ποια ήταν τα σημαντικά θέματα τα οποία ακούσαμε ε, για την έκθεση. Όλοι ε, σχεδόν οι ομιλητέ ε, έκαναν έκκληση για την ενίσχυση των ιδίων κεφαλών των τραπεζών και ότι αυτό μπορεί να αποτελέσει μειονέκτημα ανταγωνιστικό για την Ένωση δεν, δεν στηρίχτηκε. Αντίθετα, δεν μιλήσατε για άλλες πτυχές ανάληψης κινδύνου ενσωματωμένες ε, στις ε, δυνατότητες δημιουργίας ενός Ευρωπαϊκού Ταμείου Εγγυήσεων των μάλλον. Ε, μακροοικονομική προοπτική τώρα για όλες τις προτάσεις που γίνανε εγώ λόγω του, της μου θεωρώ ότι είναι μακροοικονομική η προέλευση της ίδιας της κρίσης και ο χαρακτήρας της. επίσης η ιδέα γύρω από το too weak to fail, too big to fail, too big to fail συγγνώμη, ε, ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει πολύ νόημα και θα ήταν καλύτερο να το χρησιμοποιήσουμε ε, να μην το χρησιμοποιήσουμε απέναντι στους φορείς της αγοράς. Δύο ακόμα σημεία επέμειναν στις ε, λογιστικές προδιαγραφέ και στις εργασίες του Κοινοβουλίου ανέκαθεν επιμέναμε ότι είναι σημαντικό στοιχείο την ανάγκη να καλυφθεί το shadow banking system Ό,τι και αν συμβαίνει σε ευρωπαϊκή κλίμακα, η ευθύνη των Ευρωπαίων να παρέμβουν και σε αυτό το τομέα και την ανάγκη, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της Islands αλλά που παρενέβη από αυτού την ανάγκη να ενσωματωθούν αξίες ηθικής στην εποπτεία και τη διακυβέρνηση των χρηματοπιστωτικών ε, ιδρυμάτων. Επίσης ε, σημειώνω την προειδοποίηση του κυρίου Βίσερ ότι οι κίνδυνοι όσον αφορά την υπερβολική ρευστότητα εξακολουθούν να υπάρχουν και ότι ε, όσον αφορά την προστασία του καταναλωτή και εδώ συμμερίζομαι απόλυτα την θέση της Σίκη Βαντεμπούρκ και προς αυτή την κατεύθυνση τροποποίησα κάποιες από τις προτάσεις που βρίσκονται ήδη επιτάπητος πως υπάρχει τρόπος στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού συστήματος που φτιάχνουμε να ενισχυθεί αυτή η προστασία των καταναλωτών μέσω του SMART δηλαδή την ε, αρχή για την εποπτεία των αγορών. Δηλαδή να καλύπτεται Καλύπτεται τα προϊόντα όλα μαζί.